Ο πρόεδρος. Παρακαλώ, συναδέλφοι, καθίστε. Εξ ονόματος του Κοινοβουλίου και εκ μέρους μου προσωπικά θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στους συγγενείς και στα θύματα, στους συγγενείς και στους φίλους των θυμάτων του τραγικού ατυχήματος του Ουκρανικού σκάφους που συνετρίβει λίγο μετά την απογείωσή του από την Τεχεράνη την Τετάρτη. Έχασαν τη ζωή τους και οι 176 επιβάτες και μέλη του πληρώματος θα γίνει μια έρευνα σε βάθος και διαφανής ελπίζουμε ούτως ώστε να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη στη μνήμη των θυμάτων. Σας καλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή προς μνήμη τους. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ράζα, Γιώργο Κνεβιτσένα, έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Η κυρία, συγγνώμη. Θα συνεχίσω στα λιθονικά, Πρόεδρε. Στις 13 Ιανουαρίου του 1990 δόθηκε η τελευταία μάχη στα βαλτικά κράτη και με καθυστέρηση γιατί είχαν περάσει 50 χρόνια από το σύμφωνο Μολοτοφ-Ρίμπεντροπ. Όμως ήταν νικηφόρα αυτή η μάχη στο πέτο ε, ευτυχώς που δεν έχετε και εσείς το ρουλούδι είναι μια μέρα με τραγικές απώλειες σήμερα γιατί είχαμε το θάνατο πολλών ηρωικών υπερασπιστών της χώρας μας. Μέρα νίκης. Προλύανε τον δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Για μας, δύο χρόνια μετά την πρώτη η Ενάτου του 1993, τέλειωσε ο πόλεμος, όταν ο στρατός κατοχής της ΕΣΔ αποσύρθηκε. Αυτό το λουλούδι είναι ένα δείγμα ανάμνηση όσων έδωσαν τη ζωή του σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, σε Βουλγαρία, τα εκατομμύρια εκείνων των ε, θυμάτων και μέσα στην ίδια την Ρωσία. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που τον Νοέμβριο ψήφισαν υπέρ εκείνου του κρίσιμου ψηφίσματος για τις έρευνες σε σχέση με την 13η Ιανουαρίου. Αυτά είναι οι πραγματικές ευρωπαϊκές αξίες. Σας ευχαριστούμε κύριε Ευρωβουλευτή. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα σας καλωσορίζω. Ελπίζω να περάσατε καλά στις διακοπές. Συνεχίζεται η σύνοδος του Κοινοβουλίου που έχει διακοπεί στις 19 Δεκεμβρίου του 2019. Πρακτικά τη συνόδου της 19 Δεκεμβρίου έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Τα πρακτικά λοιπόν εγκρίνονται. Κάποιε ανακοινώσει τώρα. Οι ομάδες ΕΛΚΑ και ECR μου κοινοποίησαν ορισμένες ε, αποφάσεις, ε, τροποποίησεις όσον αφορά τους ορισμούς σε αντιπροσωπείες ε, και επιτροπές. Οι αποφάσεις αυτές θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά της σημερινής συνόδου και θα τεθούν σε ισχύ την σημερινή ημέρα της ανακοινώσης. Μετά από την εκλογή της κυρίας Κάρολιν Σαντλέρ στην κυβέρνηση της Αυστρίας το Κοινοβούλιο δηλώνει το ότι παραμένει καινή η θέση της από τις 7 Ιανουαρίου του 2020. Σύμφωνα με τον ιστορικό μας κανονισμό, η συναδελφός μας έγινε υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της ευχόμαστε ότι καλύτερο για τη μελλοντική της θέση. Μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τη 19 η Δεκεμβρίου του 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει την έκλογη ε, μελών ε, στο εκ μέρου της Ισπανίας των κυρίων Ριολιον Κύρα Ιβίε, κύριο Ποκτεμόνη Κασαμαχώ και Κομίνη Ολιβέρε από τι 2 Ιουλίου του 2019 λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της ε, εκλογικής, ε, Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της 3ης Ιανουαρίου 2020 της Ισπανίας και μετά από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας της 9 η Ιανουαρίου του 2020 το Κοινοβούλιο ε, δηλώνει ότι παραμένει καινή η θέση του κυρίου Οριόλ Γιουνκέρα από τις 3 Ιανουαρίου του 2020 σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού, μέχρι να ε, επαληθευτούν οι εξουσίες τους και να αποφασιστεί κάτι σε σχέση με πιθανές ενστάσεις. Οι κύριοι Αντώνη Κομίνη Ολιβέρες και Πουίτς Μονικά Σαμαχώ θα είναι μέλη πλήρη του Κοινοβουλίου και των οργάνων του με όλα τους τα δικαιώματα αφού δηλώνεται ότι δεν υπάρχει καμία, κανένα πρόβλημα συμβατότητας με το ρόλο του Ευρωβουλευτή η κυρία Ελίζαμπετ Χάρις, η κυρία Ανοντσιάτα Μέρι Ρισμόγκ και ο κύριος Τζον Λόγγουερθ εγκατέλειψαν τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές και εντάχθηκαν στην ομάδα ECR από τις 10 Ιανουαρίου του 2020. Οι ευρωβουλευτές έτσι Μονίκα Σαμαχώ και Κομίνη Ολιβέρες θα ενταχθούν στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές η Επιτροπή Γιούρη αποφάσισε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις δύο οργανικές ε, εν ώψη της πρώτης ανάγνωσης του Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ιστορικού κανονισμού, οι θέσει που έχει οθετήσει το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση, που αποτελούν τι εντολέ για τι εν λόγω διαπραγματεύσει, είναι διαθέσιμε στην ιστοσελίδα τη Ολομέλεια και οι τίτλοι του θα δημοσιευτούν στα πρακτικά της, Συνόδου. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί στην τακτική διαδικασία. Θα ήθελα να ενημερώσω την Σύνοδο ότι την Τετάρτη. Μπορείτε να καθίσετε παρακαλώ κύριε Ευρωβουλευτή. Καθίστε, δεν θα συζητηθεί εδώ κάτι. Παρακαλώ, μείνετε ήρεμοι. Ήθελα να ενημερώσω την Ολομέλεια ότι την Τετάρτη θα υπογράψω δυνάμει του άρθρου 79 του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου δύο πράξεις που εγκρίθηκαν ε, στην, ε, με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Οι τίτλοι θα δημοσιευτούν λεπτομερώς στα πρακτικά της παρούσας συνόδου. Για όλα αυτά δεν γίνεται φυσικά συζήτηση. Όπω ήθεστε. Περάσω, ας περάσουμε στις εργασίες μας. Το τελικό σχέδιο ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ καθίστε. Κύριε Βουλευτά, μείνετε, να είστε ήσυχο. Το τελικό σχέδιο ημερήσια διάταξη όπω εγκρίθηκε από την διάσκεψη των Προεδρών στις 9 Ιανουαρίου ε, δυνάμει του σχετικού άρθρου έχει διανεμηθεί. Ας δούμε τώρα κάποιες προτάσεις ε, για τροποποίησεις. Μετά από διαβουλεύσεις με τις πολιτικές ομάδες θα ήθελα να υποβάλω ε, στη συνέλευση εδώ την ακόλουθη πρόταση αλλαγής του τελικού σχεδίου ημερησίας διαταξής όσον αφορά την Πέμπτη. Ο τίτλος της συζήτησης ε, θα, για τον Μπουρούντι, ειδικότερα η περίπτωση των κρατουμένων δημοσιογράφων, αλλάζει σε Μπουρούντι ειδικότερα ελευθερία έκφρασης. Υπάρχουν ενστάσεις. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, εγκρίνεται η τροποποίηση. Όσον αφορά τη Δευτέρα, η ομάδα του ΕΛΚΑ ζήτησε ο τίτλος της δήλωσης της Επιτροπής για το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα και οι επιπτώσεις του στην ελεύθερη κυκλοφορία να αλλάξει σε διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα και οι επιπτώσεις του στην ελεύθερη κυκλοφορία η περίπτωση του Μάλμε και της Κοπενχάγης. Κύριε Τομπέ, θέλετε να παρουσιάσετε την πρόταση αυτή, παρακαλώ. Sweden has uh, uh, τη Σουηδία έχουμε σοβαρά προβλήματα. Βία σε σχέση με εργονομένο έγκλημα. Ιδίω έχει θυγεί η πόλη του Μάλμε, βόμβε, ανταλλαγή πυροβολισμών. Αυτά είναι καθημερινά φαινόμενα στην ε, πόλη αυτή. Πέρσι η Δανέζικη κυβέρνηση ξεκίνησε συνοριακού ελέγχου μεταξύ των δύο χωρών για να προστατεύσει του Δανού από τι συμμορίε από την Σουηδία. Πρόκειται για μια μοναδική απόφαση γιατί καμία άλλη κυβέρνηση ε, στην Ευρώπη δεν έχει ξεχωρίσει έτσι κάποιες ε, ε, γειτονικέ συμμορίες και αυτό να είναι πρόφαση για συνορικού ελέγχου. Έχει κλεμακωθεί επομένω στο Μάλμο και στην Κοπενχάγη αυτή η ε, έκφραση βία. Αυτό θα πρέπει να τα βάλουμε στον τίτλο του ψηφίσματος και επίσης ζητούμε ονομαστική ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Οι σοσιαλδημοκράτες δεν θέλω να φέρουν τα προβλήματα του μάλλον στον ε, τίτλο. Αυτό είναι πολύ απογοητευτικό. Να ευκαιρία αυτό το κοινοβούλιο να δράξει είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για Σουηδία, Δανία και για Ευρώπη. Ευχαριστούμε κύριε Τομπέ. Θα ήθελε κάποιος να παρέμβει ε, με την αντίθετη άποψη. Παρακαλώ κύριε Ιράς. Αυτό που εγώ θεωρώ εξαιρετικά λυπηρό είναι να χρησιμοποιούμε ε, αυτή την ε, ολομέλεια που επιτρέπει να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη για τρίτη συνεχή φορά για να κερδίσουμε μια ψηφοφορία που χάθηκε δύο φορές ήδη. Γιατί δύο φορές το ΕΛΚ προσπάθησε να μεταφέρει το θέμα αυτό στη διάσκεψη των Προέδρων και οι υπόλοιπε ομάδες τους είπαμε απερίφραστα ποια είναι η θέση μας. Εάν το κρίνεται απαραίτητο να το ξαναπούμε. Θεωρούμε πως είναι σημαντικό να μιλάμε για τους κινδύνους του οργανωμένου εγκλήματος, χωρίς όμως να χρειάζεται να ποινικοποιούμε ένα θέμα και να ε, ε, ε, καταδικάζουμε μια ολόκληρη πόλη όπως κάνετε σε αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να επιμένετε, αλλά να ξέρετε πως η στάση των υπόλοιπων πολιτικών ομάδων θα παραμείνει η ίδια. Λοιπόν, σε ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία έρχεται η ψηφοφορία για το αίτημα αυτό. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Λοιπόν, πάμε. συνεχίζουμε με τη Δευτέρα. Η ομάδα ID ζήτησε ο τίτλος της δήλωσης της Επιτροπής ε, για τις καταστροφικές πυρκαγιές ε, στην Αυστραλία και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα εξαιτία της κλιματικής αλλαγής να αλλάξει σε καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία ενεργοποίηση του προγράμματος Rescue. Δίνω το λόγο στην κυρία Μέλα για να παρουσιάσει το αίτημα της ομάδας ID. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πραγματικός ε, εφιάλτης για μία Ήπειρο να καίγονται και να γίνονται καπνός και στάχτες, ζώα, φυτά. Είναι μία τεράστια απειλή και χρειάζεται να αντιδράσουμε συλλογικά. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε ε, δείχνοντας πως εμείς στην Ευρώπη έχουμε αλληλεγγύη προς αυτή τη φίλη χώρα, την Αυστραλία. Και το πρόγραμμα Rescue, παρόλο που σε θεωρητικό επίπεδο περιορίζεται στα κράτη-μέλη, μας επιτρέπει να το κάνουμε. Να στείλουμε δηλαδή στην Ήπειρο αυτή επιχειρησιακές δυνάμεις έτσι ώστε να καταστήλουν τις φλόγες. Και αυτό που ζητώ είναι να κάνουμε μια τροποποίηση στη δήλωση της Επιτροπής μας για αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, Ευχαριστούμε για την αντίθετη άποψη. Δίνουμε τον λόγο στον κύριο Κόκαλη, παρακαλώ. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, Δυστυχώς αυτός ο εφιάλτης της Αυστραλίας δεν έγινε από μόνο στο γενελό της ε, αλλαγή του κλίματο. Και συμφωνήσαμε για την αλλαγή του τίτλου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύουμε ότι είναι η ηθική μα ευθύνη να χρησιμοποιηθεί το Rescue παντού με κάθε μέσον. Οπότε εμείς δεν έχουμε καμία ένσταση να μπει αυτό στον τίτλο. Δεν θέλουμε όμως να απαλληφθεί η μνήμα της κλιματικής αλλαγής από τον τίτλο. Ακούσαμε λοιπόν τις δύο προτάσεις. Το αίτημα θα ψηφιστεί τώρα τις χειρός. Ποιος συμφωνεί με την πρόταση της κυρίας Μελά. Παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας. Ποιος είναι κατά. Παραμένει λοιπόν χωρίς αλλαγή ημερήσια διάταξη. Για την Τετάρτη η ΓΚΟΕ ζήτησε να προσθεθούν δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την υπερβολική χρήση βίας από τις αρχές επιβολής του νόμου σε ειρηνικές διαδημαρτυρίες και διαδηλώσεις ως δεύτερο σημείο για το απόγευμα. Θα πρέπει να καταλήξει η συζήτηση σε ένα ψήφισμα το οποίο θα ψηφιστεί την Πέμπτη. Η κυρία Ανσοφή Πελετιέ, θέλετε να παρουσιάσετε το αίτημα της ομάδας Γκουε. Ευχαριστώ πολύ. Πριν από ένα χρόνο ψηφίσαμε εδώ κατά της αστυνομικής βίας στις ευρωπαϊκές χώρες. Και παντού όσοι συγκεντρώνονται και διαδηλώνουν στην Ευρώπη περνάνε δύσκολα στα χέρια της αστυνομίας και σκεφτούμε ιδιαίτερα τους Έλληνες, τους Γάλλους, τους Βέλγους παρόλες τις καταδίκες από την Amnesty International, από τις ΜΚΟ, από ε, τους ε, όσοι υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, από το δικαστήριο. Είδατε τι συνέβη ε, αυτή την εβδομάδα με μία κοπέλα την οποία ε, στρίμωξε και έσπρωχνε η αστυνομία. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να απαγορεύεται η χρήση χημικών όπλων, για παράδειγμα, όπως ε, επίσης ε, και εξοπλισμού ΜΑΤ, όπως απαγορεύεται σε κάποιες από τις ευρωπαϊκές χώρες. Και το λέω αυτό γιατί στο κείμενο που μιλάει για τις θεμελιώδεις ελευθερίες αυτή την εβδομάδα, ε, κρίνουμε πως και η ελευθερία του να διαδηλώνει είναι μία από τις θεμελιώδεις ε, ευρωπαϊκές ελευθερίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριο Σκέμπ την αντίθετη άποψη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία μου, νομίζω ότι αναφέρεται και στη δική μου χώρα, την Πολωνία. Εκεί είναι πάρα πολύ νυφάλιες οι διαδηλώσεις και δεν υπάρχει καταστολή από την αστυνομία αλλά για την Γαλλία θα πρέπει να σεβαστούμε την επικράτηση του κράτους ε, δικαίου. Από πλευράς του ΙΣΙΑΡΑ, Πρόεδρε, να μας επιτρέψετε να ζητήσουμε να, προ... συζητηθεί το δικό μας ψήφισμα την Τετάρτη. Ψηφίζουμε για την πρόταση της κυρίας Πελέτια με ονομαστική ψηφοφορία, αρχιτή ψηφοφορία. Πρέγω. Παρακαλώ, κύριε Γκαρσία Πέρες. Κύριε Γκαρσία Πέρες. Κύριε... Μήπως γίνεται να ζητήσουμε χωριστή ψηφοφορία γιατί από ό,τι γνωρίζουμε ε, έχει προταθεί συζήτηση με ψήφισμα. Εμεί συμφωνούμε να γίνει συζήτηση, αλλά όχι ψήφισμα. Αν είναι δυνατόν επομένως να γίνει διαχωρισμό στην ψηφοφορία και εμεί συμφωνούμε για τη συζήτηση. Πρόεδρος. Λοιπόν, πρώτη ψηφοφορία για την πρόταση Πελέτχε για συζήτηση χωρίς ψήφισμα. Ποιος είναι υπέρ. Ψηφίζουμε άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παραμένει λοιπόν χωρίς αλλαγή ημερήσια διάταξη. Σα ευχαριστούμε. Τετάρτη η ομάδα ECR ζήτησε προσθήκη ως δεύτερο θέματο μια δήλωση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου στη Γαλλία και ειδικότερα περιπτώσει βία κατά δικηγόρων που διαμαρτύρονται που διαδηλώνουν θα καταλήξει αυτό σε ένα ψήφισμα που θα ψηφιστεί την Πέμπτη. Κυρία Κέμπα, θα παρουσιάσετε εκ ονόματος της ε, ομάδας ECR την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Όταν συζητάμε τη χρήση βίας κατά ανυπεράσπιτων ε, ε, ε, δικηγόρων στο Παρίσι, όταν προσπαθούν να καταπνίξουν τα κίτρινα γυλαίκα τη στιγμή που διαδηλώνουν, ε, νομίζω τότε θα πρέπει να γίνει συζήτηση ε, και ψήφισμα για το κράτος δικαίου στη Γαλλία. Το δικαίωμα του να διαδηλώνει και το δικαίωμα του να εκφράζει ελεύθερα είναι θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρώπη. Και το λέει και το άρθρο 12 ε, της Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καθένας από εμά πρέπει να έχει το δικαίωμα του συνέρχεσθε, της διαδήλωσης, της ελεύθερης έκφρασης και καταλαβαίνετε πως ε, τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία είναι ε, διαφορετικά από όσα έχουμε στην χάρτα όπως επίσης και στην θήκη της Λισαβόνας. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γαλλία για παράδειγμα, θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτές τις αρχές, γιατί αυτό που γίνεται δεν είναι σωστό. Οι διαδηλωτές δεν θα πρέπει να καταστέλλονται με τον τρόπο αυτό. Ονομαστική ψηφοφορία λοιπόν, έτσι ώστε όλοι να εκφραστούμε ε, και να εκφραστούμε κατά της χρήση βίας εναντίον ανυπεράσπιτων δικηγόρων. Ποιο έχει αντίρρηση, λέει ο Πρόεδρο. Κανένας δεν θέλει να παρουσιάσει αντεπιχείρημα. Έτσι λοιπόν ας ψηφίσουμε διάνατα χειρός την πρόταση της κυρίας Κέμπα. Ποιος συμφωνεί με την κυρία Κέμπα, σηκώστε το χέρι σας. Ποιο είναι κατά. Απορρίπτεται η πρόταση. Έτσι οριστικοποιείται η μερική διάταξη. Ας περάσουμε τώρα στην πρώτη συζήτηση που αφορά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία. Diamo la parola Σέρκοβιτς. Ο Επίτροπος κύριος Σεύκοβιτς, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank Αξιότιμα μέλη. Θα περιμένω λοιπόν λιγάκι έτσι ώστε να ηρεμήσει η κατάσταση στην αίθουσα. Ένα λεπτό πριν ξεκινήσει η συζήτηση, αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ λοιπόν όσοι από εσά δεν θέλουν να συμμετάσχουν να αποχωρήσουν από την αίθουσα με ησυχία σας παρακαλώ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη δήλωση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δασοπυρκαγιές στην Αυστραλία και, τις άλλες, ε, και τα άλλα ακραία φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις μπλε κάρτες με τη συνήθη διαδικασία αλλά και με το ηλεκτρονικό σύστημα. Έχετε οδηγίες στην είσοδο μπαίνοντα θα ήθελα τώρα λοιπόν να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Σεφκοβίτς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Παρόλες τις δραματικές και ίσως ε, τραγικές στιγμές στις οποίες θα αναφερθούμε, είναι η πρώτη φορά που βλεπόμαστε μετά τα Χριστούγεννα, γι' αυτό θα ήθελα παρόλα αυτά να σας ε, ευχηθώ σε όλους και σε όσους εκπροσωπείτε καλή χρονιά. Καλή χρονιά και καλό 2020. Θα είναι μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις. Και πραγματικά χαίρομαι που το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι αυτή η επίγουσα συζήτηση για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία. Ξέρετε κι εσείς πως οι συνάδελφοι ε, υπουργοί έρχονται από Λουξεμβούργο στο Στρασβούργο που ορκίζονται στο ΔΕΚ και γι' αυτό έχω τη χαρά να τους εκπροσωπήσω εγώ σήμερα το απόγευμα εδώ στην Ολομέλεια. Ξέρετε κι εσείς πως αυτό που μας επιβεβαιώνει η Αυστραλία είναι αυτό που πιστεύουμε κι εμείς. Δεν έχουν ξαναυπάρξει τέτοιες πυρκαγιές. Έχουν καταστρέψει μικρές κοινωνίες, έχουμε τεράστια απώλεια σε νοικοκαιριά, έχουν χαθεί ζωές και ίσως και πάνω από ένα δισεκατομμύριο ζώα, κάποια τα οποία είναι πραγματικά μοναδικά στην πλάση. Έχουμε καταστροφή ε, δασών, γεών, ε, ζώων, οικοσυστημάτων και επίσης οι πυρκαγιές αυτές ε, προκαλούν βλάβη και σε άλλες περιοχές, για παράδειγμα στην Καμπέρα, η ατμοσφαιρική ρήπανση ήταν 20 φορές ε, πιο ψηλά από το όριο όπου θεωρείται ε, επικίνδυνη. Θέλουμε να εκφράσουμε λοιπόν στήριξη και λιγή καταρχήν προς την Αυστραλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να βοηθήσει τους Αυστραλούς. Την Κυριακή ο Επίτροπος Λέναρτσης μίλησε με τους Αυστραλούς και τους επανέλαβε την προθυμία μας να βοηθήσουμε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή. Επίσης, ενημέρωσε ε, τους Αυστραλιανούς Υπουργούς για τη δυνατότητα του να στείλουμε πυροσβέστες μια και έχουμε πια το μηχανισμό πολιτικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκφράστηκαν με ευγνωμοσύνη για την προθυμία μας και την ετοιμότητα να βοηθήσουμε, αλλά ο υπουργό ο Αρμόδης μας είπε πως αυτή τη στιγμή δεν χρειάζονται επιπλέον βοήθεια. Αξιότιμα μέλη. Η επιστήμη το λέει δυνατά και βροντερά. Η κλιματική ανάγκη θα ε, αυξήσει το ρυθμό αυτών των ακραίων φαινομένων και θα μας επηρεάζουν με όλο και περισσότερες επιπτώσεις, με όλο και μεγαλύτερη ένταση. Χρειάζεστε κι άλλες αποδείξεις πως η αλλαγή του κλίματος, η καταστροφή του περιβάλλοντος ε, θα πρέπει να καταπολεμηθούν απαραίτητα πως θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ε, εξισορροπήσουμε αυτές τις καταστροφές που συμβαίνουν στην Αυστραλία και αλλού. Εδώ και πολλούς μήνες συζητάμε τη σημασία που έχει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγετικό ρόλο στα θέματα κλίματος παγκοσμίως. Στόχοι από το Παρίσι, ε, Green Deal, Πράσινη Συμφωνία και Σύμφωνο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έχουμε τα εργαλεία για να αντιμετωπίζουμε αυτή την παγκόσμια κλιματική πρόκληση μαζί με τις χώρες εταίρους, με τις οικονομίες των G20 που παράγουν τρία τέταρτα των παγκόσμιων εκπομπών. Εμείς εκτιμάμε ιδιαίτερα την μακρόχρονη σχέση που έχουμε με την Αυστραλία και θέλουμε να κάνουμε διάλογο μαζί τους για τα όσα μπορούμε να κάνουμε για το περιβάλλον στα πλαίσια της Συμφωνίας Πλαίσιο. Ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο που ξεκίνησε αυτή την επίγουσα συζήτηση και που καταλαβαίνει ότι το κλίμα επήγει. Σας ευχαριστούμε γιατί υπό αυτές τις περιστάσεις πρέπει να φωτίσουμε την ανάγκη για παγκόσμια δράση. Αυτό αποδεικνύει για μια φορά ακόμα πως εμείς έχουμε τη φιλοδοξία ε, να καταπολεμήσουμε από ηγετική θέση την ε, κλιματική αλλαγή. Εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τώρα εκ μέρου των πολιτικών ομάδων για ένα λεπτό εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Η κυρία Μπέντελε παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Σεύκοβιτ, ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Δύο παρατηρήσει θέλω να κάνω. Πρώτον, δεδομένη τη νέα επιτροπή και τη κατάσταση τη Πράσινη Συμφωνία και τη διάσκεψης στη Μαδρίτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αλλάξει σαφώ την εξωτερική τη πολιτική και να συμπληρώσει τη διάσταση του κλίματο. Δεν γίνεται να έχουμε συνόδου κορυφή ε, και διασκέψει διπλωματικέ ε, που να αναφέρονται στην ε, τήρηση των στόχων χωρίς να γίνεται τίποτα. Η ευρωπαϊκή διπλωματία για το κλίμα πρέπει να ενισχυθεί και θεσμικά ούτω ώστε να καταστεί σαφές ότι στο μέλλον και δύσκολοι εταίροι όπως η Αυστραλία θα συμφωνήσουν μαζί μας γρήγορα. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο τρόπος καταπολέμησης των πυρκαγιών είναι εμφισβητήσιμος. Ο τρόπος ε, πυρόσβεσης στην Αυστραλία είναι από τους καλύτερους στον τρόπο. Παρ' όλα αυτά ε, ήταν πιο δυνατή η πυρηνή Ε, θα αφήσει ακατοίκητες ε, πολλές περιοχές στο μέλλον. Το 2018 είχαμε στην ε, Ελλάδα 100 νεκρούς. Τα φυτά στην Αυστραλία τέτοια φυτά όπως στην Αυστραλία υπάρχουν σε πολλές περιοχές του, κόσμου και μπορεί να έχουμε παρόμοια προβλήματα το επόμενο καλοκαίρι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει για την πρόληψη και να ενισχυθεί η κλιματική διπλωματία της Ευρώπης. Παρακαλώ να τηρείτε τις χρονοθυρίδες αγαπητοί συνάδελφοι. Δίνουμε τώρα το λόγο ε, εκ μέρους της ομάδας των σοσιαλιστών ε, στην κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ πολύ. Θα θεωρούσαν ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν γίνονται σε μια μεγάλη ήπειρο, μακριά από την Ευρώπη. Όμως αυτό με τίποτα δεν ισχύει. Ε, έτσι έχουμε τώρα περισσότερο διοξίδιο στην ατμόσφαιρα και έτσι τώρα έχουμε τοξικότητα στον αέρα. Αυτός ο καπνός από τις ε, πυρκαγιές είναι κακός για όλο τον ε, πλανήτη. Μόνο στο Queensland έχουμε 106 εκατομμύρια τόνους που εξελίθησαν όσον αφορά το διοξίδιο. Και τώρα έχουμε βοήθεια ε, αυτό προκαλεί επίσης και κυκλώνες και έχει γίνει μεγάλη καταστροφή ε, καταστράφει η γη όσο είναι το Βέλγιο και η Ολλανδία μαζί πάνω από ένα δις ζώα εκτός από τους ανθρώπους και πρόκειται για μια κρίση βιοπικιλότητας έχει πάρα πολλά ε, είδη που υπάρχουν μόνο στην Αυστραλία περίπου στα 200. Επομένως δεν θα πρέπει αυτά να τα βλέπουμε ε, με αδράνεια, θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε πρωτοπόροι στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Είδατε τι έγινε, τι έκανε η κυβέρνηση, τι δεν έκανε όταν είχε φωτιά στον ε, Αμαζόνιο. Δισταγμός ε, επικράτησε αυτούς τους μήνες για να συνδέσουμε το φαινόμενο με την αντικλιματική αλλαγή. Θα πρέπει επομένως εμείς να αποφύγουμε τέτοια λάθη και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά για τα οποία δεσμευθήκαμε στο Παρίσι. Όπως ε, λέμε τώρα, ε, θα, αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι φωτιές και τελικά πρόκειται να αλλαγή το κλίματος. Ε, χέρι-χέρι θα αντιμετωπίσουμε αυτά, γι' αυτό και η κυβέρνηση θα πρέπει να αναγνωρίσει την κλιματική αλλαγή αιτία, θα πρέπει να τιμήσουμε τις δεσμεύσεις των Παρισίων πριν να είναι πολύ αργά. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους του Renew Europe για δύο λεπτά η κυρία Μίλλερ παρακαλώ εκ μέρου τη ε, αντιπροσωπεία για τι σχέσει με την Αυστραλία και την Ζηλανδία, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω τη λύπη μου για τα θύματα των πυρκαγιών στην Αυστραλία. Αυτέ τι δύσκολε ημέρε ε, όπου χάθηκαν τόσε ζωέ, ε, τόσα σπίτια, τόσα ζώα, τόσους φυσικός πλούτος στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τον λαό της Αυστραλίας. Ε, η σκέψη μας πηγαίνει στους συγγενείς και τους φίλους των ε, τραυματιών, των νεκρών και θέλουμε να εκφράσουμε τη φιλία μας προς αυτούς και τη στήριξή μας και προς τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Φυσικά τίθενται ερώματα για τους λόγους αυτών των καταστροφικών πυρκαγιών. Γενικά είναι ζεστό και ξηρό το κλίμα στην Αυστραλία και οι πυρκαγιές ε, είναι κομμάτι χαρακτηριστικό της Αυστραλιανής φύσης και βοηθούν ε, και στην ανανέωση ορισμένων φυσικών πόρων. Οπότε, ε, το, ωστόσο το κλίμα, η κλιματική αλλαγή οδήγησε σε ξηρότερες ε, εποχές στην Αυστραλία με αποτέλεσμα αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ποιες είναι οι συνέπειες. Πρέπει να ελέγξουμε να δούμε κατά πόσο ο μηχανισμός που υπάρχει για την καταπολέμηση είναι επαρκής. Αυτό πρέπει να το δούμε και εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για του δικού μα μηχανισμού, ούτω ώστε εάν προκύψουν τέτοιε εξαιρετικέ περιπτώσει σε άλλε χώρε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ε, παράσχουμε βοήθεια. Φυσικά θα πρέπει να τηρήσει του κλιματικού στόχου η Αυστραλία και θεωρούμε δεδομένο ότι οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν και λόγω των τεράστιων δυνατοτήτων που μα προσφέρουν οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ο Πρωθυπουργό, ο κ. Μόρσεν, χθε το είπε στον τύπο. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ήδη το Φεβρουάριο πρόκειται να ταξιδέψει στην Αυστραλία και εκεί επί τόπου μεταξύ άλλων θα διαπιστώσει ποιες ήταν οι συνέπειες των πυρκαγιών και ε, πώς έχει προοδεύσει η διαδικασία προστασίας του κλίματος. Θα κάνουμε ε, εκτενή συζήτηση με τους βουλευτές και με την κυβέρνηση και πρέπει να πούμε τώρα ότι ε, αυτές τις δύσκολες στιγμές προσφέρουμε την υποστήριξή μας στους Αυστραλιανούς φίλους ώστε και είμαστε στο πλευρό τους για την καταπολέμηση αυτής της τεράστιας φυσικής καταστροφής. Thank you very much. Now, on of the... Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των Πρασίνων, για ένα λεπτό, ο κύριος Χολγκριν. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σας πω πως αυτή τη στιγμή η Αυστραλία περνάει το πιο ζεστό καλοκαίρι ποτέ, όπως επίσης και το πιο ξηρό καλοκαίρι ποτέ. Μέση θερμοκρασία για το Δεκέμβριο, 4 βαθμοί πάνω από τη συνηθισμένη. Αυτό είναι ακραίο. Και έχουν εξεπερέσει κατά 1,7 βαθμού το τελευταίο ρεκόρ που ήταν ο περσινός Δεκέμβριος. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως εδώ βρισκόμαστε στο σενάριο για το οποίο μας είχαν προειδοποιήσει οι εμπειρογνώμονες. Τι σημαίνει η αλλαγή κλίματος, περισσότερη ξηρασία, περισσότεροι καύσονες, περισσότερες περιπτώσεις δάσοπυρκαγιάς. Και η πολιτική για το περιβάλλον που ακολουθούμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φτάνει. Και αυτό ισχύει και για τη ΣΥΠΑ, την Κίνα, την Αυστραλία και για το λόγο αυτό εμείς αντιμετωπίζουμε όλο και υψηλότερες θερμοκρασίες. Και το καλοκαίρι αυτού του τύπου θα θεωρείται πλέον φυσιολογικό καλοκαίρι. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς στην Ευρώπη πολύ περισσότερα και πολύ πιο σύντομα. Όχι το 2050, όχι το 2030. Φέτος. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της ID, για ένα λεπτό, η κυρία Λίμερ. Παρακαλώ. Αυτό που με ενοχλεί σε αυτή τη συζήτηση είναι αυτή η αυτοικανοποίηση της αριστεράς των πρασίνων ε, να καταγγέλνουν αυτές ε, τις ε, φρικτές πυρκαγιές και λένε αυτή είναι επιπλέον η απόδειξη της κλιματικής αλλαγής. Ντροπή σας. Διαρκώς πάντα υπήρχαν τέτοιες πυρκαγιές οι οποίες είναι κομμάτι του οικοσυστήματος της Επίρου το 85, το 93 το 75, άλλες ε, πολλές χρόνιες τέτοιες ε, και ε, ετησίως βρέχει και περισσότερο παντού. Βασικά, βάσει των στατιστικών στοιχείων, να συμβαίνει αυτό τα τελευταία 120 χρόνια. Ο λόγος για τις πυρκαγιές, μεταξύ άλλων, μπορεί να είναι και ο εμπρισμός διότι με την πολιτική προστασία του κλίματος ε, υπάρχουν διάφορες ε, συνέπειες καταστρεπτικές. Αυτά τα γεγονότα δεν ε, απαλύνουν τον πόνο των πληγέντων, ούτε το δράμα που βλέπουμε στο ζωικό βασίλειο. Ευχαριστούμε. Εκ μέρου ε, του ECR για ένα λεπτό η κυρία Βυσνιεύσκα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κοιτάξτε τι γίνεται στην Αυστραλία. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση και θα δείτε πως οι πυρκαγιές αυτές επηρεάζουν ολόκληρη την Ήπειρο και κρατάνε εβδομάδες. Έχουν καταστρέψει όλη τη χώρα, ε, ενδιαιτήματα, βιοπικιλομορφία, άνθρωποι, ζώα, περιουσίες. Καταλαβαίνετε πως μας έχει συγκινήσει ιδιαίτερα η κατάσταση αυτή με μια ξηρασία η οποία διαρκεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και βεβαίως ισχύουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι ε, αναζωπυρώνουν αυτές τις φυρές. Αλλά ξέρετε πως αυτές οι πυρκαγιές σε θαμνόδεντρα και σε θαμνόδε εκτάσεις στην Αυστραλία δεν είναι κάτι καινούριο, συμβαίνουν κάθε χρόνο. Και αν ακούσετε κάποια από τα σχόλια τα οποία γίνονται κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θα δείτε πως ναι, μεν ανησυχούμε εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κλιματική αλλαγή, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι έχουμε κάνει εμεί. Μια φορά το μήνα ταξιδεύουμε για το Στρασβούργο και οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι τεράστιες. Και βεβαίως το κόστος της διατήρησης της έδρα μας εδώ. Ε, εκατοντάδες ε, εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν μην το ξεχνάμε και αυτό. Εκ μέρους λοιπόν ε, εκ της ΓΚΟΕ ο κύριος Κόκαλης. Mr. Vice President, in Australia είναι χωρίς προηγούμενα αυτές οι φωτιές, αυτές οι πυρκαγιές, αλλά ήταν κάτι το προσδόκιο το 2008 δεν έγινε τίποτα και είχε ε, προβλεφθεί ότι θα κρατήσει περισσότερο εξήρα περίοδος και έτσι θα είχαμε την αύξηση αυτών των πυρκαγιών και ότι τα πράγματα έτσι θα γίνουν και από το 2020 και από το GOC το 2018 ελέγχεται το ίδιο, μεγαλύτερο καλοκαίρι, μεγαλύτερες τέτοιες ε, εκτάσεις, μεγαλύτερες πυρκαγιές, αλλά και στη Νότια Ευρώπη. Ακόμη και με το καλύτερο σενάριο, ε, η προβολή, η, η, προ, τα προγνωστικά για το μέλλον αποκλειπτικού χαρακτήρα και τι κάνει η κυβέρνηση, ε, δεν προσυπογράφει την συνδικία το κλίμα και Κύριε Πρόεδρε, δεν θα πρέπει εμείς να κάνουμε το ίδιο λάθος με την κυβέρνηση της Αυστραλίας. Θα πρέπει να κάνουμε αυτά τα οποία ε, ζητούν οι επιστήμονες και τα παιδιά μας. Προσαρμογή, προστασία και να είμαστε πρωτοπόροι σε αυτή την ε, προσπάθεια μέσα από το New Green Deal. Η ε, πρόεδρος, τους μη γεγραμμένους. Ένα λεπτό. Κυρία Εύη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι πυρκαγιές που καταστρέφουν την Αυστραλία από το Σεπτέμβριο έχουν έναν τραγικό απολογισμό. Το βλέπουμε 25 νεκροί, πάνω από 10 εκατομμύρια εκτάρια καταστράφηκαν, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ζώα σκοτώθηκαν. Η πρωτεύουσα η Κανμπέρα με τους 500.000 κατοίκους της έχει τη χειρότερη ποιότητα αέρα στον κόσμο. Έφτασαν οι καπνοί μέχρι τη χιλή για την Αργεντινή. Είναι απαράδεκτος ο απολογισμός δεν είναι παρά ένα ακραίο φαινόμενο που προστίθεται στα υπόλοιπα ε, που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Οι δραματικές εικόνες όμως της πυρκαγιάς δεν αρκούν για τον ε, Πρωθυπουργό της Αυστραλίας. Όχι μόνο καθυστέρησε να αποκριθεί, αλλά δήλωσε ότι η κυβέρνησή του, η συντηρητική, δεν πρόκειται να ενισχύσει τι πολιτικέ ε, καταπολέμησης τη κλιματική αλλαγή. Η Αυστραλία επίση ήταν μία από τι χώρε που μαζί με τη Βραζιλία παρεμπόδισε σημαντικά τις διαπραγματεύσεις ε, στην τελευταία COP25 στη Μαδρίτη. Η Επιτροπή αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών με την Αυστραλία. Πώς θα δράσετε ώστε να εισαχθούν στόχοι βιωσιμότητας και προστασίας του περιβάλλοντος ε, στο κεφάλαιο βιώσιμης ανάπτυξης και να περιλαμβάνονται και κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστούμε για ένα λεπτό. Ο κύριος Βιέζικ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Το πρόβλημα δεν είναι οι πυρκαγιές. Αυτό είναι κομμάτι της φύσης. Ε, αυτές οι θαμνώδεις περιοχές και η συγκεκριμένη χλωρίδα και πανίδα μπορούν να επανέλθουν. Το ζήτημα είναι οι συνθήκες ε, αυτά τα χρόνια ε, ξηρασίας με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που ξεπερνάνε κατά τέσσερις βαθμούς την φυσιολογική για την εποχή. Ε, όλα αυτά μας ε, ε, δημιουργούν ανησυχίες για το μέλλον γιατί θα γίνονται οι συνθήκες αυτές όλο και πιο συνηθισμένες αν δεν μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αν δεν προσαρμοστούμε. Διαφορετικά αποτελεί ένα κουδούνι που χτυπάει για μας η Αυστραλία και χρειάζεται μια παγκόσμια πρωτοβουλία που θα μεταμορφώσει τις εθνικές πολιτικές, γιατί ε, εντάξει, μπορεί να μας φαίνεται πως είναι μακριά και εξωτική και μικρή η Αυστραλία, αλλά μην νομίζετε, δεν είναι τόσο μακριά από εμά τελικά. Η κυρία πήρε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Τέσσερις τεράστιες φωτιές ε, καίνε στη χώρα μήνες. Από το Σεπτέμβριο 28 άτομα έχασαν τη ζωή τους, χιλιάδες νοικοκυριά καταστράφηκαν. Οι πυροσβέστες κινδυνεύουν τη ζωή τους για να σώσουν ζωές. Εμείς ε, εκφράζουμε τη συμπάθειά μας για τον λαό της Αυστραλίας ε, αυτή τη δύσκολη στιγμή, όπου βρέχει στάχτες, όχι νερό, και ξέρετε πως αυτές οι ακραίε πυρκαγιέ δεν μπορεί να είναι κάτι ε, που να το βλέπουμε αποσπασμένο από την κλιματική αλλαγή. Δεν είναι φυσική καταστροφή απλώς, είναι κλιματική επίγουσα ανάγκη. Αυτή η καταστροφική πυρκαγιά ίσως ε, συνετίσει κάπω την πολιτική ε, του, του συντηρητικού Πρωθυπουργού κ. Μόρισον που δεν έχει κάνει τίποτα για να συμμορφωθεί με τι υποχρεώσει του για το κλίμα και να σας πω πως ε, συναντήθηκε με την ε, Σαουδική Αραβία και την Βραζιλία για να ε, παρακολύσει τις προσπάθειες ε, μέτρων για την κλιματική αλλαγή. Μα πώ είναι δυνατόν αυτό ο Πρωθυπουργό να θεωρεί πω η κλιματική αλλαγή, τα μέτρα για την κλιματική αλλαγή είναι πιο τρομακτικά από την κλιματική αλλαγή την ίδια και αυτά που προκαλεί. Καταλαβαίνετε πώ αποτελεί αυτό μια τεράστια παγκόσμια πρόκληση για την οποία είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Οι καταστροφικέ αυτέ πυρκαγιέ υπογραμμίζουν το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργεί η αδράνειά μας σε επίπεδο COP25 και το κάνει ακόμα πιο σημαντικό να αναλάβουμε εμεί ηγητική δράση και να είμαστε πρότυπο για τους υπόλοιπους. Η Ευρωπαϊκή πράσινη, ε, το, το Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο, το Green Deal δεν φτάνει. Η κλιματική πολιτική θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όλων των συμφωνιών που υπογράφουμε παντού στον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Θα πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα και θα πρέπει όλοι οι εταίροι να μας ακολουθήσουν για να έχουμε κοινή πολιτική που θα αντιμετωπίσει την κρίση στο περιβάλλον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ακούτε τις κραυγές από την Αυστραλία. Μπορούμε να αισθανθούμε την οδύνη των θυμάτων και τον πόνο αυτών που τέχασαν όλα από την πυρκαγιά. Ένα δισεκατομμύριο ζώα έγιναν στάχτη. Πρόκειται για ένα σήμα κινδύνου συγκλονιστικό. Πρόκειται για ένα καμπανάκι κινδύνου για όλο τον πλανήτη. Έτσι θα πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτά το έγιναν στην Αυστραλία. Να, ε, γιατί κάνουμε το New Green Deal και έχουμε 300.000 Ευρωπαίους εκεί σε Αυστραλία, Νέα Καλλιδονία, Νέα Ζηλανδία. Αυτή ήταν η πρώτη μάρτυρα της μεγάλης καταστροφής. Σήμερα στην Ευρώπη θα πρέπει να κινητοποιηθούμε, να είμαστε αλληλέγγυοι. Βεβαίως. Όμως θα πρέπει με ευθεία να αντιδράσουμε, να κινητοποιηθούμε σε πολιτικό επίπεδο ε, αφού έχουμε κηρύξει κατάσταση ανάγκης για το κλίμα γιατί πώς δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται ε, με την ε, απορρίθμιση που είναι εις βάρος του κλίματος αυτό που έπαθε σήμερα η το πάθει αύριο ο πλανήτης δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν ακόμα σκεπτικιστές σε όλο τον κόσμο και εδώ δεν καταλαβαίνουν το ότι η οικολογία δεν έχει ε, σύνορα. Στην ε, Χιλή έφτασε ένα τέτοιο τοξικό σύννεφο, πέρασε τον ε, ωκεανό, 80% της πανιδεχλωρίδας μας προέρχεται από την άλλη μεριά της υδρογείου επομένως για το New Green Deal θα πρέπει να καλύψουμε και αυτές τις ε, υπεράκτες, υπερπόντιες ε, πτήσει. Η κυρία Καβατσίνη για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι εφιάλτης η πυρκαγιά στην Αυστραλία και διαρκώς λέμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ε, ως Ευρωπαίοι. Είναι σαφές η αλληλεγγύη μας πρέπει να δοθεί στην Αυστραλία, αλλά δεν φτάνει η αλληλεγγύη. Πρέπει να δούμε πώς ε, η οικονομική μας σχέση με την Αυστραλία θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Ο Πρωθυπουργό Μόρισαν ε, μάλιστα είπε ότι υπάρχει ε, σχέση μεταξύ της προστασίας του κλίματος και των πυρκαγιών. Πρώτο παράδειγμα, θα έχουμε τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών φέτος με την Αυστραλία. αυτή η συμφωνία θα οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών βάσει ανάλυσης της Κομισιόν. Θα αυξηθεί η παραγωγή κρεάτων στην Αυστραλία και άλλα προϊόντα τα οποία θα στέλνουν σε ολόκληρο τον κόσμο και αυτό θα θερμανεί περισσότερο τον πλανήτη. Δεύτερο παράδειγμα, γνωρίζουμε όλοι ότι πρέπει να βγούμε το συντομότερο δυνατόν από τον άνθρακα, αλλά η Αυστραλία έχει από τη μεγαλύτερη παραγωγή άνθρακα στον κόσμο, μαζί τα οποία εξάγει στη Siemens, στην Ευρώπη και η Αυστραλία και... Ε, δεν τηρεί τους ε, στόχους του Παρισιού. Χρειαζόμαστε μια κλιματική αλλαγή στην οικονομική μας πολιτική και στην, στην εμπορική μας πολιτική στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα για ένα λεπτό η κυρία Μπρούνα. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τα φρικτά γεγονότα στην Αυστραλία έχουν οδήγησει στο θάνατο 28 ανθρώπων, καταστροφή δασικών περιοχών ίσης έκτασης με την Αυστραλία και εξαφάνιση πάνω από ένα δισεκατομμύρια ζώα. Θα χρειαστούν πολλές, πολλοί αιώνε για να ξαναβρεθεί αυτή η βιοπικιλότητα. Και οι ζημιές που έχουν γίνει είναι μερικές ανεπανόρθωτες. Να θυμίσουμε ότι η ελεύθερη συναλλαγή που ετοιμάζεται να συνάψετε θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης. Ε, ε, ε, στην προπαγάνδα του μάλιστα παρακινεί σε δασικές πυρκαγιές επίσης. Οι ειδικοί από την Ευρώπη σε θέματα πυρόσβεσης καθυστέρησαν να φτάσουν στην Αυστραλία. Ας βοηθήσουμε την Αυστραλία και ας ενισχύσουμε για να αποφύγουμε μελλοντικά δράματα το μηχανισμό Risk e εκ μέρους της Ευρώπης ας οργανώσουμε μια διακριτική ομάδα που θα μπορεί να σταλεί για να αντιμετωπίσει μεγάλες πυρκαγιές εκτός της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα για ένα λεπτό η κυρία Πελετιέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά ποτέ σε επίπεδο τετραγωνικών χιλιόμετρων, σε στάχτες, σε ζώα που χάθηκαν, σε ανθρώπους που μετακινήθηκαν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που να μπορούμε να το συγκρίνουμε. Είναι απερίγραπτο, δεν έχει προηγούμενο. Είναι κάτι το οποίο όμω θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Η υπεύθυνη όμω δεν είναι ούτε η κακοτυχία, ούτε οι περιστάσει, ούτε ο συνδυασμό αυτών. Γιατί έχουμε αυτούς του οποίου προτιμούν την ανάπτυξη από το περιβάλλον, που φτωχοποιούν μονοπολούντας τα κοινά αγαθά. Όσο αυτή τη στιγμή πνίγεται και καίγεται η ε, Αυστραλία πουλά παρόλα αυτά ε, το νερό η κυβέρνησή της. Τι συμβαίνει λοιπόν με τις δικές μας συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Πότε θα συμπεριλάβουμε σε αυτές υποχρεώσεις κλιματικές. Πότε θα το κάνουμε. Την Τρίτη ε, θα ψηφίσουμε και θα ανοίξουμε την πόρτα στα λόμπι που ρηπαίνουν. Άρα λοιπόν το φιλελεύθερο σύστημα το οποίο ε, λατρεύεται έφερε την κλιματική αλλαγή και θα φέρει την κλιματική καταστροφή ε, στο μέλλον και οι αγορές σας δεν πρόκειται να σας σώσουν. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό. Ο κύριος Πεντιτσίνη παρακαλώ. Ανεξαρτητός. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι μόλις μάθαμε την είδηση για τις τραγικές πυρκαγιές στην Αυστραλία, αμέσως μάθαμε ότι συλλήθηκαν και περίπου 200 πυροναμείς που ενδέχεται να προκάλεσαν αυτές τις πυρκαγιές. Αυτό αποδυναμώνει, αρνείται τη σχέση μεταξύ ε, θέρμανσης του πλανήτη και πυρκαγιών. Αλλά το θέμα εδώ δεν είναι να πούμε ποιες ήταν οι αιτίε των πυρκαγιών αυτών, αλλά να πούμε ποιες ήταν οι αιτία που δια, διαδόθηκαν τόσο γρήγορα. Είναι σαν να μην βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο ε, συμβαίνει ταυτόχρονα παντού. 50 βαθμοί ήταν η θερμοκρασία όταν συνέβησαν όλα αυτά και κατά ηρωνικό τρόπο όλα αυτά γίνονται σε μια χώρα που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας άνθρακα παγκοσμίω και που αρνήθηκε τις συμφωνίες για το κλίμα. Είναι ηρωνικό που ε, εκεί έχει αυξηθεί περίπου 1,5 βαθμό, 1,5 βαθμό η θερμοκρασία εκεί ε, φέτος το καλοκαίρι στην Αυστραλία. Οπότε φανταστείτε τι μπορεί ακόμα να συμβεί. Ευχαριστώ η κυρία Ευχαριστώ. Το 2020 είναι η χρονιά της βιοποικιλότητας και αυτές οι πυρκαγιές οι οποίες ε, χτύπησαν την Αυστραλία ε, είναι κάτι το κατεπίγον θα πρέπει να κάνουμε. Έχουμε πάνω από ένα δις ζώα τα οποία χάθηκαν στις ε, φλόγες και έχουμε πάρα πολλά από αυτά τα ζώα που ήταν ζώα που εξαφάνισε, τα κοάλα, τα καγκουρό, ε, οι εικόνες αυτές ήταν ε, κάτι που σόκαρε τον κόσμο, πρόκειται για ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Ε, είναι κάτι το οποίο αφορά τη βιοπικιλότητα. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Αυτό θα είναι πράξη αυτοκτονίας, οι διατροφές, το οξυγόνο, το πρόεδρο τι σύλλες, το κλίμα. Είναι όλα αυτά το που αφορούν το ε, κλίμα και δεν θα πρέπει να τα καταστρέφουμε, θα πρέπει να τα διασώσουμε και θα πρέπει να δούμε ε, ποιες από τις υποσχέσεις μας ε, τηρήσαμε. Ας ξυπνήσουμε να αντιστρέψουμε αυτήν την ε, τάση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι θα πρέπει να επικεντρωθεί ε, σε αυτήν την πολιτική για την βιοποικιλότητα την στρατηγική 2020 και έτσι να μπορέσουμε να πετύχουμε στους στόχους που έχουμε τάξει. Θα πρέπει να αναλάβουμε δράση η Πρόεδρος. Για ένα λεπτό και μισό, κυρία Γκούτελαντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η δεκαετία ξεκίνησε με κακά μαντάτα για την Αυστραλία με αυτές τις ε, πυρκαγιές που κάτεγαψαν την ε, χώρα σε εκτάσεις ε, όσο κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θέλουμε να εξασφαλίσουμε να είναι βιώσιμος ο πλανήτης μας για εμάς τους ανθρώπους για μας, για τα ζώα, ε, δεν θα πρέπει η γη να γίνει ήλιος από την ε, άλλαγη του κλίματος. Όμως, ε, ξεκίνησε μια εποχή με σκοτάδι, γιατί έχουμε συζητήσει για το κλίμα, οπότε ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Η υπόθεση που είναι κατεπίγουσα, η αλλαγή του κλίματος αποτύχαμε κατά την τελευταία δεκαετία. Τάξαμε στην Μαδρίτη κάποιους φιλόδοξους στόχους. Οι πολιτικοί που δεν ε, τηρούν αυτούς τους στόχους ε, μας δημιουργούν απογοήτευση. Οι νέοι μας λένε εσείς στο κοινοβούλιο δείξτε υπευθυνότητα. Να τηρήσετε αυτά για τα οποία δεσμευθήκατε στο Παρίσι. Έχω ένα παιδί 7 ετών και μου είπε να, τι γίνεται ε, με το κλίμα, δεν φταίνε οι εξατμίσεις, ε, τα καυσαέρια των αυτοκινήτων. Ένα παιδί το είπε αυτό. Τα παιδιά μας παρακαλούν να είμαστε πιο φιλόδοξοι, πιο τολμηροί με την στρατηγική μας για το κλίμα. Τόρβολτ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε δάση ευκαλύπτων που κάηκαν στην Αυστραλία, που είναι πολύ ιδιαίτερα. Το λέμε, είναι η βιοπικιλότητα, είναι ε, η ιδιαιτερότητα της Αυστραλίας που απέχει ε, και έχει ένα διαφορετικό ενδιέτημα και που ε, βασίζεται στους ευκαλύπτους για όλη την βλάστηση που περιβάλλει αυτούς. Εκεί μέσα ζουν ζώα, έντομα, άλλη βλάστηση. Γιατί λοιπόν τα δάση ευκαλύπτουν είναι τόσο σημαντικά. Γιατί αν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς, τότε χάνεται ε, η υγρασία και είναι εκρηκτική η πυρκαγιά, κάτι το οποίο έχουμε δει και σε άλλες ε, πυρκαγιές, όχι μόνο στην Αυστραλία. Τι κάνει λοιπόν η Αυστραλιανή κυβέρνηση. 5% της, ε, του μείγματος ενέργειας στην Αυστραλία είναι από ΑΠΕ. Όλα τα υπόλοιπα είναι από ρηκτά ε, καύσιμα. Νομίζω αυτό είναι αρκετό. Για ένα λεπτό ο κύριος Νινίστο. Οι φρικτές σκηνές στην Αυστραλία αποδεικνύουν πως η βιοπικιλότητα που χάνεται και η κλιματική αλλαγή ε, πάνε χέρι-χέρι. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ζώα, για ένα μεγάλο κομμάτι της πολύ ιδιαίτερη φύσης ε, και των ενδιατημάτων στην Αυστραλία που πια χάθηκαν. Η κλίμακα της καταστροφής είναι κάτι το οποίο πρέπει να ε, κατανοήσουμε, γιατί αν δεν προσαρμοστούμε δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι καταστροφές που θα φέρει η κλιματική αλλαγή και στην Ευρώπη. Πρέπει τις πυρκαγιέ αυτές σε δάση στην Ευρώπη να τις αντιμετωπίζουμε καλύτερα, να είμαστε πιο φιλόδοξοι για το κλίμα και να κάνει ό,τι χρειάζεται και ε, να κάνουν ό,τι χρειάζεται και χώρε όπως η Αυστραλία. Είναι σημαντικό ε, να δείξουμε αλληλεγγύη προ το λαό της Αυστραλίας, Εμεί, οι Ευρωπαίοι, και να τονίσουμε το τρόπο με τον οποίο θα αντιστρέψουμε αυτές τις απώλειες στην Αυστραλία. Να τους βοηθήσουμε σε αυτό, αλλά στην κλιματική πολιτική χρειάζεται να τους δώσουμε και μια σκουδιά. Ευχαριστούμε τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Χακεράιναν. Ευχαριστώ. Το κέριο ερώτημα είναι να μάθουμε τι προκάλεσε αυτές τις πυρκαγιές. Αυτές δεν προκλήθηκαν από την κλιματική αλλαγή. Πυρκαγιές ε, τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε σχεδόν παντού στον κόσμο. Ναι, μεν, υπάρχει αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά το κατά πόσο αυτό ήταν η αιτία για αυτές τις πυρκαγιές είναι αμφισβητήσιμο. Οι πυρκαγιές συχνά προκαλούνται από τον άνθρωπο, εσκεμένα ή όχι. Στην περίπτωση της Αυστραλίας ε, είχαμε εμπρισμούς από ανθρωπογενείς εμπρισμούς. Εδώ λοιπόν ε, πάσχουμε από ιστερία νομίζω. Ουσιαστικά επιβάλλουμε πεπιθήσεις εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό η κυρία Χάζεκαμπ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι συγκλονισμένη από τις πυρκαγιές στην Αυστραλία. Εκατομμύρια εκτάρια έχουν χαθεί ε, ζώα όπως τα καγκουρό, κοάλα. Δεν, τους δόθηκε καμία ευκαιρία ε, να επιζήσουν σε αυτή την πύρινη λέλαπα. Είναι καταστροφή για τον άνθρωπο, για το περιβάλλον, για τα ζώα. Πόσε καταστροφέ χρειαζόμαστε για να αλλάξουμε επιτέλου ε, κατεύθυνση. Στα τελευταία 100 χρόνια έχει αυξηθεί η θερμοκρασία κατά 1,5 βαθμό. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το καταπολεμήσουμε αυτό και να στραφούμε και κατά της κτηνοτροφίας επιτέλους ε, η καταστροφή των δασών, η αποψήλωση των δασών, η αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα σε τεράστια κλίμακα συμβάλλουν στην κλιματική κρίση που επιδεινώνει τις πυρκαγιές αυτές. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του πλανήτη μας ε, και το πυρούνι μας ε, είναι το πιο σημαντικό όπλο για να βοηθήσουμε ε, στην, κλιματική, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να καταργηθούν οι γεωργικές επιχορηγήσεις και να τρώμε λιγότερο κρέας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λόβ, παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι βέβαιος ότι όλοι εδώ θα συμφωνήσουν μαζί μου να στείλουμε ευχές ε, και την αλληλεγγύη μας ε, στο λαό της Αυστραλίας ε, σε αυτή την εθνική καταστροφή. Με απογοητεύει που κατηγορούμε την κλιματική αλλαγή ω κύρια αιτία για αυτέ τι πυρκαγιέ. Τόσο εδώ στο Κοινοβούλιο και άλλου διάφορου υποτιθέμενου εμπειρογνώμονε του κλίματο. Αυτή η θρησκεία τη κλιματική αλλαγή προχωρά χωρί να υπάρχουν πραγματικά στοιχεία που να το αποδεικνύουν. Η λογική μας λέει ότι η κλιματική αλλαγή δεν έχει πολλά να κάνει με αυτή τη φυσική καταστροφή. Η μεγαλύτερη ε, πυκνότητα του πληθυσμού σημαίνει ότι πολύ περισσότερο κόσμο πετά τα τσιγάρα του, πολύ περισσότερε πίθε υπάρχουν από ηλεκτρικά καλώδια, ε, πολύ περισσότεροι ανάβουν φωτιά στην άγρια φύση όταν κάνουν κάμπινγκ και φυσικά υπάρχει και ο εμπρισμό. Ε, δεν υπάρχει καμία κατανόηση των συνεπειών αυτών. Εδώ στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουμε κάτι να... και για να μειώσουμε τη δική μας, το δικό μας ανθρωπικό αποτύπωμα όταν έχουμε ε, τα κτίρια μας σε τρεις ε, διαφορετικές περιοχές του πλανήτη δεν πρέπει να κρίνουμε τους άλλους ε, να κάνουμε και εμείς αυτά που πρεσβεύουμε αντί να στεκόμαστε εδώ ως υποκριτές. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε. Δέχεστε μια επερώτηση από τον κύριο Κόκαλη. Μπλε κάρτα. Κύριε Κόκαλη, έχετε το λόγο. Thank ε, ευχαριστώ. Στην Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή σας ε, η άποψη για την πυκνότητα του πληθυσμού και τις γόπες. Τι λέτε όμως ε, για το ότι έχουμε άνοδο ε, θερμοκρασίας χωρίς προηγούμενο. Οπότε έχουμε πάρα πολύ λίγη υγρασία. Όλο ένα και λιγότερη. Και έτσι έχουμε ε, αυτές τις ε, πυρκαγιές παρά τις Γόπε. πάρα πολύ απλή είναι η απόψή μου. Δείτε την ιστορία. Τέτοιε πυρκαγιέ στην Αυστραλία υπάρχουν ε, τα τελευταία χρόνια, χιλιάδε χρόνια. Συγγνώμη, συνάδελφε. Ε, σας έδωσα τον λόγο και σα υπενθυμίζω ότι έχετε μισό λεπτό, μισό λεπτό, έχετε τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ο κύριο Λόβ, και κατά τη γνώμη μου όλα αυτά είναι άσχετα με την ξηρασία ή την ε, άνοδο της θερμοκρασίας, όπως λέτε εσείς. Τελικά όμως πάρα πάρα πολλούς αιώνες και δυστυχώς πάρα πολλές φορές είναι αυτά. Τα περισσότερα έγιναν το 1974 1975 τότε όμως είχαμε τις περισσότερες βροχές ε, που είχε ποτέ η Αυστραλία. Και γι' αυτό φύτρωσαν πάρα πολύ θάμνη και έτσι είχαμε τις σχετικές πυρκαγιές. Ε, έχουμε αυτές τις παραδόσεις των ε, γηγενών που ε, εάν δεν τους αφήσουν να κάνουν αυτές τους, τις, να κάψουν αυτούς τους θάμνους που χρειάζεται να κάψουν όταν ξέρουν ότι πρέπει, τότε έχουμε τα προβλήματα. Ο κύριος και ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι κοιτώντας στην Αυστραλία βλέπουμε τι μορφή έχει πραγματικά η καταστροφή. Τεράστιες περιοχές έχουν Καταστροφή από τις πυρκαγιές ε, τεράστιοι καύσονες. Ε, η ρήπανση του αέρα στην Καμπέρα ήταν 25 φορές περισσότερη από το επιτρεπόμενο όριο. Ένα δισεκατομμύριο ζώα χάθηκαν σε αυτές τις πυρκαγιές. Αυτές είναι οι πραγματικές σκηνές της κόλασης. Θα ήθελα να εκφράσω την ελληνική μας και τη συμπόνια μας ε, στο λαό της Αυστραλίας και σε όσους επλήγησαν, όσους έχασαν τα σπίτια τους και τους αγαπημένους τους. Αλλά τώρα θα πρέπει να ρωτήσουμε και την ε, Αυστραλιανή κυβέρνηση τι θα κάνει για να αναλάβει τις ευθύνες της, γιατί προς το παρόν δεν κάνει απολύτως τίποτα για να μειώσει τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα. Ταυτόχρονα εξάγουν τα αποθέματικά τους ε, άνθρακα. Ας κάνουμε λοιπόν επιτέλους πιο υγιή τον πλανήτη. Για 1,5 λεπτό η κυρία Βαν Μπρέμπτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Ακούσαμε πολύ ακραίες απόψεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά νομίζω πως τούτη τη φορά μπορούμε να πούμε με ασφάλεια πως η κλιματική αλλαγή, η υπερθέρμανση του πλανήτη έχουν συνέπειες. Αυτές οι πυρκαγιές που ξεσπάνε κάθε χρόνο είναι πλέον μια φυσική, ανθρωπογενής και ανθρωπιστική καταστροφή. Είναι σημαντικό εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδείξουμε πως είμαστε υπεύθυνοι. Έχουμε το καινούριο Green Deal. Έχουμε τη βούληση να κινηθούμε ε, με τρόπο που θα οδηγηθούμε σε μια κοινωνία και σε μια οικονομία η οποία σέβεται το κλίμα. Τώρα που μιλάμε, υπογράφουμε μια νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Αυστραλία. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτή την επιρροή ως μοχλό για να περάσει η Αυστραλία από την πλευρά ε, των όσων κάνουν το σωστό δεν είναι σωστό να θέλει να έχει πρόσβαση στην αγορά μας η Αυστραλία και παρόλα αυτά να μην μας ακολουθεί στις δράσεις που κάνουμε υπέρ του κλίματος. Οι επόμενε λοιπόν εμπορικές συμφωνίες που θα υπογράψουμε στο μέλλον είτε με την Αυστραλία είτε με κάποιον άλλον θα πρέπει να ε, επαναλαμβάνουν τις διατάξεις από τη σύμβαση ε, του Παρισιού ε, και νομίζω πως θα πρέπει να μετακινηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα να ε, δώσουμε το καλό παράδειγμα και στη συμφωνία με την Αυστραλία να τα λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Δέχεστε την μπλε κάρτα από τον κύριο Μπάουτ. Ωραία. Κύριε Μπάουτ, ο λόγος είναι σε εσά. Σας παρακαλώ, μπορείτε να σηκωθείτε όρθιος και σας δίνω και 30 δεύτερα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω την εξή ερώτηση στη συνάδελφο και κυρίως να σχολιάσω. Πιστεύετε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω Εάν θέλουμε να επηρεάσουμε την παραγωγή, έχουμε τα πράσινα πιστοποιητικά. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένας ολόκληρος βιομηχανικός κλάδος. Ε, θέλετε λοιπόν να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, γιατί αυτό τι θα σημάνει. Ε, αυτή τη στιγμή εισάγουμε 10 ε, εκατομμύρια τόνους χάλιβα από τη Βραζιλία, ενώ μειώνουμε την παραγωγή στις δικές μας χαλιβουργίες. Τι σημαίνει αυτό για τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή μειώνουμε τι δικέ μα και εισάγουμε από χώρε οι οποίε δεν μειώνουν τι δικέ του εκπομπές. Τι άποψη έχετε κυρία μου. Έχετε το λόγο κυρία Φομπραντ. Ο συνάδελφος ε, έθεσε ένα θέμα το οποίο είναι ακριβώ περιγράφει αυτό που λέω για την εμπορική μα πολιτική. Δεν έχει κανένα μα κανένα νόημα εμεί εδώ στην Ευρώπη να είμαστε ουδέτεροι ε, κλιματικά και να επιτρέπουμε προϊόντα από άλλα μέρη του κόσμου όταν τα μέρη αυτά δεν έχουν ούτε τους ίδιους στόχους, ούτε τις ίδιες και ρηπαίνουν πολύ περισσότερο. Να χρησιμοποιούμε ακριβώς για το λόγο αυτό την εμπορική μας πολιτική έτσι ώστε η κλιματική μας πολιτική να ευνοηθεί. Κλιματική ουδετερότητα προστατεύοντας δε και τη βιομηχανία μας. Ευχαριστώ πολύ για ένα λεπτό η κυρία Τουσά. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Μετά από την Αμαζονία τώρα καίγεται η Αυστραλία. 10 εκατομμύρια εκτάρια καταστράφηκαν από τις φλόγες. 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από ένα δισεκατομμύριο ζώα χάθηκαν. Οι επιστήμονες ε, έχουν πει ότι υπάρχει σχέση αδιαμφισβήτητη μεταξύ, αδιαμφισβήτη μεταξύ του κλίματος και αυτών των πυρκαγιών και όσοι αμφισβητούν συνεχίζουν. Ε, και αυτοί είναι ουσιαστικά υπερομανής. Ε, η χώρα ίδια, η κυβέρνηση η ίδια εξάγει κάρβουνο, υπερασπίζεται ε, τις ε, βιομηχανίε παραγωγή άνθρακα, ο τρόπος κατανάλωσης. Το να θέτουν σε κίνδυνο ε, τη φύση εκεί, θέτει σε κίνδυνο τη φύση σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσω τη αδράνεια, η οποία είναι εγκληματική. Θα πρέπει επιτέλου να κάνουμε κάτι για αυτή την καταστροφή, ε, να αναγνωρίσουμε τα περιβαλλοντικά εγκλήματα, να ξαναδούμε τι οικονομικέ μα συνθήκε, ε, τι συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών βάσει των κλιματικών παραγόντων. Καίγεται ο πλανήτη σα, μην περιμένουμε την τελευταία πυρκαγιά να καταστραφεί το τελευταίο δέντρο πριν δράσουμε. Ευχαριστούμε. Τώρα για ένα λεπτό η κυρία Μελάν παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι άμεσε συνέπειε των πυρκαγιών στην Αυστραλία είναι αυτέ που είπα στην αρχή όταν ζήτησα να αλλάξει ο τίτλο τη συζήτηση. Θα ήθελα να προσθέσω την ιδέα των δραματικών συνεπειών. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα χαθεί η βιομάζα, ε, περισσότερη ξηρασία και τεράστιες πιέσεις στη φύση σε μια χώρα όπου ήδη το νερό σπανίζει. Φυσικά οι πυρκαγιές σχετίζονται με, την, ε, με το ιδιαίτερο θερμό καλοκαίρι στην Αυστραλία, αλλά προφανώς υπάρχει ε, η ανάγκη να δοθούν άμεσες και συγκεκριμένες απαντήσεις. Γι' αυτό ήθελα να αλλάξουμε το τίτλο ε, της συζήτησης. Προφανώς για λόγους πολιτικούς το Κοινοβούλιο αρνήθηκε την πρότασή μου να συμπεριλάβουμε το πρόγραμμα Rescue το οποίο θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί για να βοηθήσουμε τους Αυστραλούς. Και αντί γι' αυτό, ακόμα αυτά που μόλις άκουσα τώρα, τεράστιες δηλώσεις για την κλιματική αλλαγή, αλλά ας μην κάνουμε τίποτα, ε, καμία πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ρόλαν, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τραγικές αποτρόπες πυρκαγιές. Για άλλη μια φορά τις ε, εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι. Ε, αυτοί που όλα τα θέλουν ανθρωποκεντρικά και ακριβώ το έχουν ως πρόφαση ενώ το φαινόμενο αυτό έχει περίπλοκες ε, αιτίες ε, και έχουμε τους εμπρισμούς έχουμε την πολυνομία, αλλά υπάρχουν κάποιοι ζηλωτές οι οποίοι δεν ε, περιορίζουν ε, τα δέντρα σε μερικά σημεία ή τους ε, θάμνους που βοηθούν την πυρκαγιά. Δεν στη δεκαετία του 1920 αλλά και σε άλλες περιόδους υπήρχε πάλι πάρα πολύ μεγάλη επισύλλες θερμοκρασίες και ξηρασία Επομένως, να σκεφτούμε ότι αυτή η πράσινη ιδεολογία είναι μια φενάκη και θα πρέπει να σταματήσουμε να μεταχειριζόμαστε αυτές τις ε, τραγωδίες για να προγάγουμε αυτό μας το θεματολόγιο. Πρόκειται για προσπάθειες που πέφτουν στο κενό γιατί δεν κάνουν τίποτα για τον θερμοστάτη της ε, υδρογείου. Η Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Ζέμτσα. Την δέχεστε. Μάλιστα. Κύριε Ζέμτσα, έχετε μισό λεπτό. Ευχαριστώ. Είναι ενδιαφέρον οι αιτίε αυτών των πυρκαγιών. Πρόκειται για την αλλαγή του κλίματος, της θερμοκρασίας, αλλά συγκεκριμένα θέλω να ρωτήσω, είπατε ότι είχαμε και νομοθετικές μεταβολές στην Αυστραλία όσον αφορά δηλαδή τις αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και είπατε ότι τώρα την αρμοδιότητα την έχουν οι τοπικές αρχές. Πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος των πρασίνων. Δεν θέλουν παρεμβάσεις. Έτσι μου είπανε, εσείς το επιβεβαιώνετε, έχετε κι εσείς ε, μισό λεπτό να απαντήσετε κύριε. Έχει δίκιο ο αξιότιμος φίλος και έκανα κάποια έρευνα την περασμένη εβδομάδα και φάνηκε πως το λόμπι των, ε, ε, του περιβάλλοντος ακριβώς αυτό απέφυγε. Δηλαδή μετακίνησε την πολιτική προς το ομόσπονδο επίπεδο και εκεί Έχουμε το λόμπι που δεν επιτρέπει ούτε ε, κοπή, ούτε ε, ε, να καίγονται μικρές ε, εκτάσεις που υπάρχει λόγος. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό όντως να επιστρέψει η επικουρικότητα, έτσι το λέγαμε, έτσι ώστε οι τοπικές αρχές να μπορούν να αποφασίζουν ήδη τι είναι καλύτερο και να κυβερνάνε ήδη στη δική τους περιοχή. Για ένα λεπτό η κυρία Περέιρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί Ευρωπαίοι πολίτες, να σας πω τα εξή, Η βία με την οποία οι πυρκαγιές αυτές κατέστρεψαν την Αυστραλία αφήνουν μία και μοναδική εντύπωση φρίκης και θρήνου για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, για το δασικό πλούτο που χάθηκε, για τη βιοπικιλότητα που χάθηκε, για τα νοικοκυριά που καταστράφηκαν, για το φόβο που έζησαν οι Αυστραλοί και θα πρέπει να τους στηρίξουμε με αλληλεγγύη. Εμείς στην Πορτογαλία δυστυχώς το πρόβλημα το γνωρίζουμε. Έχουμε υποφέρει και εμείς με ανθρώπινες ζωές, με ε, πολλά δασικά ζώα που χάθηκαν τα τελευταία χρόνια η καταστροφή αυτή ε, δεν αντιστρέφεται. Η πολιτική ζητά δράση και στην Ευρώπη εμείς προχωράμε με τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής και θέλουμε να είμαστε μια ήπειρος ουδέτερη σε εκπομπές δεξιοδίου του άνθρακα, να είμαστε οι πρώτοι παγκοσμίω. Και αυτό αποδεικνύουν οι πυρκαγιές σε Καλιφόρνια, Αυστραλία, Πορτογαλία. Δεν μπορούμε ε, παρά να ανοίξουμε τα μάτια μας και να δούμε πως ο πλανήτης καταστρέφεται. Θα ζητήσουμε από όλα τα κοινοβούλια και τους λαούς να συστρατευτούν μαζί μας και να δείξουμε και απόλυτη αλληλεγγύη στο λαό της Αυστραλίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης. Φορά που η Αυστραλία πλήττα από πυρκαγιές. Όμως σε συνεχιζόμενη ξηρασία και υψηλέ θερμοκρασίες που έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ το μήνα Δεκέμβριο επιδίνωσαν σημαντικά την κατάσταση. 28 άνθρωποι έχουν πεθάνει και σπάνια είδη πανίδας κινδυνεύουν από εξαφάνιση μια έκταση μεγαλύτερη από το βέλγιο και τη δανία μαζί έχουν γίνει στάχτη. είναι εντυπωσιακά παράλογο βέβαια πω οι χώρε με τι μεγαλύτερε πυρκαγιέ αυστραλία βραζιλία ηνωμένε πολιτείε με μπροστάρι τον κύριο τραμπ δεν θέλουν να υλοποιηθεί η συμφωνία των παρισίων και βέβαια με συνοδοιπόρου κάποιου συναδέλφου εδώ σήμερα οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν επηρεάζεται η κλιματική αλλαγή από ανθρωπογενή αίτια. πραγματικά ο τρόπο σκέψη θυμίζει αυτούς που κυνηγούσαν το γαλιλαίο αιώνες πριν. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Εμείς πρέπει να αγωνιστούμε για να υλοποιηθεί η Συμφωνία των Παρισίων και συγχρόνως να βρεθούν τα απαραίτητα χρήματα ώστε το rescue που είμαι εισηγητής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι έτοιμο από το 2021 ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και στην Ευρώπη αλλά και στον τρίτο κόσμο. Ένα λεπτό, η κυρία Μπρικμό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το 87 το αυστραλέζικο συγκροτήμα, Midnight Oil έγινε διάσημο με το τραγούδι Beds Are Burning. Τα καυτά κρεβάτια και είχαν καταγγείλει την καταστροφή του περιβάλλοντος. Αυτό μετά από 30 χρόνια παραμένει επίκαιρο είναι η κατάσταση τέτοια, οπότε έλεγε τότε πώς να χορέψουμε όταν γυρίζει η γη, όταν καίνε τα κρεβάτια. Και ακριβώ ε, αυτό είναι μια εικόνα του πώ θα είναι ο κόσμος αν δεν τηρήσουμε τη Συμφωνία των Παρισίων. Ε, χρειάζεται ελεγγύη και φέτο θα κάνουμε την συμφωνία με την Αυστραλία. Ελεύθερο εμπόριο. Επομένως χρειάζεται να υπάρχει κάτι που να έχει σχέση με βιώσιμη ανάπτυξη και δύο πλευρές ε, έχει επικυρώσει συνδική των Παρισιών η χώρα και το θέμα τι γίνεται με τις εξορίξεις είναι πάρα πολύ βασικό αυτό για τη χώρα 10% αλλά πρέπει να δούμε πώς θα προστατευτούν και οι, οι και έχουν όμως την Αυστραλία μαζί με την Σαουδική Αραβία πάρα πολύ διοξιδίου του άνθρακα θα πρέπει να γίνουν αυτά που λέει το Green Deal θα πρέπει να υπάρχει κλιματική, περιβαλλοντική διπλωματία και θα τα περάσουμε ως Ένωση μέσα από την εμπορική πολιτική. Ευχαριστούμε για να το τώρα κυρία Σπυράκη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αντιπρόεδρε Σεύκοβιτς, αν κάποιος αναζητήσει τρεις όρους για να περιγράψει τα αίτια της τραγωδίας στην Αυστραλία, θα μπορούσε να μιλήσει για αδράνεια, υπερεκμετάλλευση και κινησμό στην αυστραλία το δεκέμβριο του 2018 οι ετήσιες εκπομπές των ρήπων του θερμοκηπίου αυξήθηκαν κατά 558 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμους του διοξιδίου του άνθρακα. η αυστραλία επιμένει να αρνείται στην πράξη την κλιματική αλλαγή και γι' αυτό η παραγωγή του ηλεκτρικού της ρεύματος προέρχεται κατά 60% από άνθρακα. υπάρχουν άνθρωποι και μέσα εδώ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο που αρνούνται την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγή, ευτυχώ όμως για όλους είναι περιθωριοποιημένοι η τραγωδία στην αυστραλία μπορεί να είναι καταλήτη στις εξωτερικές μας σχέσεις ως ευρωπαϊκή ένωση. ως πρωτοπόροι στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής οφείλουμε να διευρύνουμε και να στηρίξουμε τη συμμαχία των προθήμων χωρών περιφερειών βιομηχανιών που εργάζονται για την εφαρμογή της συμφωνίας του παρισιού. το green deal μπορεί να είναι το νέο εργαλείο αλλά και το βαρύ οικονομικό μας όπλο. είναι η ώρα να δράσουμε στο όνομα των πολλών προλαβαίνοντα άλλη μια τραγωδία και δίνοντας προοπτική νέας ανάπτυξης με νέες βιώσιμες δουλειές που θα υποστηρίξουν τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό, κυρία Βάης. Ευχαριστώ. Οι άνθρωποι που μπορούν να ξεπεράσουν μόνοι του τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν είναι ισχυρότεροι. Είδαμε ε, αυτές τις ε, σοβαρότατες πυρκαγιές ε, στην Αυστραλία. Πριν από αυτές είχαμε τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο και φυσικά κάτι παρόμοιο μπορεί να συμβεί και στην Ευρώπη. Και αυτό θα επηρεάσει φυσικά τη γεωργία μας. Έχουμε δει ότι λιώνουν οι πάγοι στους πόλους, ε, όλα αυτά, όλα αυτά πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε ως πολιτικοί. Δεν μπορούμε απλά να λέμε ότι ανησυχούμε, πρέπει να δράσουμε, πρέπει να λύνουμε τα προβλήματα, να φέρουμε αποτελέσματα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει εμείς ως πολιτικοί να εγκαταλείψουμε τους δισταγμούς μας, ε, να αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο τα προβλήματα αυτά. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, θα πρέπει να επιτύχουμε και αποτελέσματα άμεσα. Πρέπει να δίνουμε λοιπόν το παράδειγμα μπροστά στους λαούς της Ευρώπης και στις νεότερες γενιές ειδικότερα πρέπει να αποδείξουμε ότι εμεί ως πολιτικοί μπορούμε να συνεργαστούμε, μπορούμε να δράσουμε και προληπτικά και να εστιαστούμε στα αποτελέσματα όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τις δυσκολίες που συνεπάγεται. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελα να συμβάλλει σε αυτό και θα ήθελα και οι άλλες ομάδες εδώ να μας βοηθήσουν σε αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Η διαδικασία κάτω λοιπόν θα ξεκινήσει και παρακαλώ τους συναδέλφους να σεβαστούν το όριο του ενός λεπτού, διαφορετικά θα σας διακόπτω. Πρώτος ομιλητής, η κυρία Σόντροβα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. μαζί με τους χιλιάδες πολίτες, έτσι κι εγώ αισθάνομαι ανυπεράσπιστη όταν βλέπω να χάνονται ζωές, να καταστρέφεται η φύση, να χάνονται ζώα. Αλλά προσπαθώ να το αντιμετωπίζω λογικά. Αποτελεί λογική συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Και μιλώ τώρα στους συναδέλφους εξ αριστερών. Γιατί η ξηρασία αυτή η ακραία ή οι ακραίες αυτές θερμοκρασίες δεν είναι πράσινη ιδεολογία, γιατί αν ήταν πράσινη ιδεολογία θα ξέραμε πώς θα την ανταπίσουμε. Είναι επίπτωση της κλιματικής αλλαγής που προκύπτει από τα γνωστά, από τις γνωστές πηγές και προκαλούν υψηλές θερμοκρασίες και φοβερή ξηρασία. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κύριο Σεύκοβιτς που προσφέρει στήριξη στην Αυστραλιανή κυβέρνηση, γιατί βέβαια οι πολίτες συνεισφέρουν ε, μέσω δωρεών, μέσω χρημάτων, αλλά πολλοί ψηφοφόροι έχουν έρθει και με έχουν ρωτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνουν. Και η απάντηση που δίνω είναι το Green Deal και ελπίζω πως θα βοηθήσει ο κ. Κασάρης για ε, ένα λεπτό. Αγαπητή Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω ε, πραγματικά τα συλληπιτήριά μου για τα όσα έχουν συμβεί στην Αυστραλία. Ας σκεφτούμε πάλι τι σημαίνει κλιματική αλλαγή. Ξέρετε πώ με αυτέ οι πυρκαγιέ εκπέμπει περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα η Αυστραλία από ότι όλο το χρόνο το Ηνωμένο Βασίλειο. Χρειάζεται να βάλουμε μέτρα σε τροχιά με μια στρατηγική για το κλίμα και για το δάσο. και να μην μεταφέρουμε τα όσα συμβαίνουν εκεί στη χώρα μα: στην Πορτογαλία, στη Γαλλική, στην Ελλάδα έχουμε φυτίες ευκαλύπτων που είναι μόνο καλλιέργειες που ε, μπορούν να καούν με τον ίδιο τρόπο που καίγονται οι ευκάλυπτοι στην Αυστραλία. Μην τους διευκολύνουμε. Όταν έχουμε συνθήκες πάνω από τους 30 βαθμούς, με κάτω από 30% υγρασίας και πάνω από 30 χιλιόμετρα άνεμο την ώρα, μπορεί να καεί ένα δάσος. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε τα διδάγματα της Αυστραλίας, έτσι ώστε να μην συμβούν στην Ευρώπη αυτά και να έχουμε στρατηγική πρόληψη που θα είναι ρεαλιστική, επειδή ακριβώς πλησιάζει η αλλαγή στο κλίμα. Ευχαριστώ πολύ για ένα λεπτό. παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί. Χάθηκαν τα κοάλα, δεν υπάρχει νερό στην Αυστραλία. Εκατομμύρια πολίτε επλήγησαν. Θέλω να εκφράσω την υποστήριξή μου προ την Αυστραλιακή κυβέρνηση για το εξαιρετικό του έργο και για του Αυστραλού πολίτε τόσο δύσκολε εποχέ. Θα ήθελα λοιπόν να ενθαρρύνω εδώ τα θεσμικά όργανα να είναι ανοιχτό μυαλί για να βοηθήσουν την Αυστραλία με οικονομικούς και άλλους πόρους για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό καλωσορίζω την προσφορά του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για παροχή αρρωγής και το να στείλουν ε, αντλίες πολλά κράτη-μέλη. Ήθελα να συγχαρώ ε, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τον Μηχανισμό Κοπένικου που παρήχε τόσο μεγάλη βοήθεια για τι πυρκαγιέ στην Αυστραλία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για ένα λεπτό η κυρία Τσόμς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Επιτρόπε, συνάδελφοι. Η πρώτη συζήτηση αφορά την κλιματική αλλαγή και αυτό έπρεπε να είναι έτσι γιατί φέτος πρέπει να είναι χρόνια που επιτέλους θα δράσουμε για το κλίμα με τις σημερινές πολιτικές ε, έχουμε τρεις ε, βαθμούς ε, θα υπερθέρμανση του πλανήτη και βλέπουμε τα αποτελέσματα στις τραγικές πυρκαγιές στην Αυστραλία και οι βουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες αναγνωρίζουν τα αποδεικτικά στοιχεία ότι η κλιματική αλλαγή είναι η αιτία που έχουμε πιο συχνά και πιο σοβαρά τέτοια φαινόμενα. Όχι μόνο οι ίδιες οι πυρκαγιές είναι τραγικές, τραγικό είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολιτικοί με μεγάλη επιρροή στην Αυστραλία που εθελοτυφλούν ε, πάνω από ανθρακοριχεία και αρνούνται ότι υπάρχει τέτοια σχέση. Ε, αντίθετα με όσους ε, καταπολεμούν με πόνο στην Αυστραλία αυτές τις πυρκαγιές και στεκόμαστε στο πλευρό σας με αλληλεγγύη προς όσους στην Αυστραλία μάχονται για να αναγνωρίσουν η κρατική λειτουργή, οι κυβερνήσεις τους, η κυβέρνησή τους, το δράμα αυτό, στεκόμαστε στο πλάι τους. Και σε όσους πρόκειται να συνάψουν ε, συμβάσεις τέτοιες που θα επιδεινώσουν το κλίμα, ξανασκεφτείτε το. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό η κυρία Ντέλιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό που βλέπουμε στην Αυστραλία σίγουρα είναι καταστροφή. Τίποτα φυσικό δεν έχει. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι οι καταστρεπτικές πυρκαγιές που μένονται σε ολόκληρη την Αυστραλία σχετίζονται άμεσα με την αδράνεια και την άρνηση της κλιματικής αλλαγής από την συντηρητική κυβέρνηση της Αυστραλίας. Οι καλύτερες συμβουλές και η υποστήριξη που μπορούμε να δώσουμε στο λαό της Αυστραλίας είναι να το αναγνωρίσουμε. Δεν είναι τυχαίο που η Αυστραλία υποστηρίζει την παραγωγή άνθρακα. Δεν είναι τυχαίο που εξακολουθεί να προσφέρει επιχορογή την βιομηχανία άνθρακα και ότι είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και υγροποιημένο φυσικό αερίο. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει ε, να μας αφυπνίσει όλους. Είναι καταστρεπτική αυτή η πολιτική, χρειάζεται αλλαγή. Δεν μπορεί να γίνεται ε, ε, ότι διατάσσουν τα βιομηχανικά λόμπι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νικολάου Λαβάνος για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η επίκληση της κλιματικής αλλαγής σαν αιτία των πυρκαγιών που στήχησαν δεκάδες ανθρώπινες ζωές και ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές καταστροφές στην Αυστραλία αποκρύπτει ότι υπάρχει επιστήμη και τεχνολογία σήμερα ικανές να περιορίζουν προλαμβάνουν και καταστέλουν τι συνέπειε φυσικών φαινομένων. δεν μπορεί να αποτελούν δικαιολογία οι όποιε αλλαγέ στο κλίμα αντίθετα θα έπρεπε εκείνες να σημαίνουν ακόμη περισσότερε πολιτικέ ευθύνε στι κυβερνήσει που όχι μόνο δεν παίρνουν τα αναγκαία μέτρα αλλά αντίστροφα αποδυναμώνει την πολιτική προστασία και πυρόσβεση. η αυστραλία αντιμετωπίζει αυτή την καταστροφή χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό με λιγοστό προσωπικό 80% είναι εθελοντές πυροσβέστες με μέσα δανεικά από άλλες χώρες. ανάλογο σχεδιασμό προβλέπει και το resceu για τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης. οι περικοπές με βάση το απαράδεκτο κριτήριο Κόστου ωφέλου, που δεν περιορίζονται στην αυστραλία αποτελούν κατεύθυνση τη ευρωπαϊκής ένωσης και των κυβερνήσεών της να μην συμβιβαστεί ο λαό με τι φυσικέ καταστροφέ με το σύνολο τη αντιλαϊκής πολιτική. η λαϊκή οργή πρέπει να γίνει οργανωμένο αγώνα για περιβάλλον και γη λαϊκή περιουσία για μέτρα ασφαλεία και προστασία του λαού. Δεν είπε. Γερμανικά μόνο. Γιώργο. Θέλω να εκφράσω τη συμπονία μου προ όλου του Αυστραλού και την ελεγγύη μου που υποφέρουν από τι πυρκαγιέ. Φυσικά αυτό είναι συνέπεια τη κλιματική αλλαγή. Είναι κάτι που δεν θα συμβεί μόνο στην Αυστραλία, συμβαίνει και στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη θα το δούμε. Θυμάστε την Πορτογαλία, τη Σουηδία και όλα τα προβλήματα που είναι σοβαρότατα. Πρέπει οπωσδήποτε να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή, αλλά πρέπει να εξοπλίσουμε και σωστά τι υπηρεσίε ε, καταπολέμηση, πυρόσβεση και διάσωση. Έχουμε ασχοληθεί με το πρόβλημα αυτό στην Ευρώπη και στην Ευρώπη οι δυνάμεις πυρόσβεσης μπορούν να δράσουν καλά, να αντιδράσουν καλά σε τέτοιες ε, περιπτώσεις ε, πλημμυρών, πυρκαγιών και αυτό που είναι σημαντικό είναι στις προσπάθειες αυτές κατά της κλιματικής αλλαγής ε, να μην παραμείνουμε μόνοι Επί παραδείγματι, δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε τη γεωργία στην Ευρώπη όπως έγινε στην Βραζιλία. Αυτό θα ήταν λάθος μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ. Για ένα λεπτό, η κυρία Φαϊόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υποστηρίξει την Αυστραλία σε αυτή την κρίση με τις πυρκαγιές. Δεν αρκεί να περιμένουμε να έρθει βοήθεια ε, από τον Αυστραλό Πρωθυπουργό η Αυστραλία δεν είναι σε θέση, είναι σαφές. Ένας οροκόσμος έχασε τη ζωή του. Ε, τέθηκαν σε κίνδυνο πόσες ανθρώπινες ζωές, ε, ζώα, κοάλα. Και στην Ευρώπη ε, έχουμε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για να προσφέρουμε βοήθεια στην Αυστραλία οι διαθέσιμες ε, δυνάμεις που υπάρχουν, οι υπηρεσίες διάσωσης θα πρέπει να πάνε εκεί. Θα πρέπει να τις προσφέρουμε και απευθύνω έκκληση προς την Κομισιόν να σχεδιάσει κοινέ ε, επιχειρήσεις. Μην χάνουμε άλλο χρόνο. Α στείλουμε τους πυροσβέστες μας στις υπηρεσίες διάσωση εκεί για να είμαστε οι πρώτοι στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωή μας, να αναλάβουμε ευθύνη, να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Για ένα λεπτό, η κυρία Φάκου, μας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, να σταθούμε δύο λεπτά και να ξεκινήσουμε με συλληπιτήρια και αλληλεγγύη προς την Αυστραλία. και επίση να εκφράσουμε το θαυμασμό μας για τους πυροσβέστες που μέρες τώρα μάχονται τις φλόγες. Είναι εξαιρετικά συγκινητικές οι προσπάθειες που κάνουν. Η κόρη μου μόλις υιοθέτησε ένα κουάλα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Να του στείλουμε ό,τι μπορεί να βοηθήσει. Δορυφορικές εικόνες, για παράδειγμα, που θα βοηθήσουν την Αυστραλία και να σας πω πως η κλιματική αναλλαγή όντως είναι θέμα εδώ. Θα πρέπει να μετακινηθούμε προς το Green Deal, προς τη Συμφωνία των Παρισίων. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως τα ψηφίσματα τα οποία εγκρίναμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, ε, έκτακτη ανάγκη που δημιουργεί το κλίμα θα ληφθούν υπόψη με τα απαραίτητα μέτρα που θα μας επιτρέψουν να υπερασπιστούμε και την υπόλοιπη ε, πλάση και την Αυστραλία. Wallis, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η κλιματική αλλαγή δεν δημιουργεί πυρκαγιές στα δάση, αλλά τι, χειροτερεύει τις πυρκαγιές αυτές. Ριζικά. Είναι από τους βασικούς παραγωγούς άνθρακα και εξαγωγής άνθρακα η Αυστραλία. Επίσης, ε, υγροποιημένου αερίου. 29 δις επιδόσεις στη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων, σύμφωνα με το Δουνουτού. Ο Πρωθυπουργός Μόρισον ε, όταν ρωτήθηκε για την κακή του επίδοση στο, στη μείωση ε, των εκπομπών, είπαν δεν θέλουμε στόχους οι οποίοι καταστρέφουν την οικονομία. Δηλαδή, είπε πως η οικονομία είναι πιο σημαντική από το μέλλον του πλανήτη. Η Ευρώπη λέει πως δεν θα υπογράφει εμπορικές συμφωνίες με όσους δεν συμπεριφέρονται σωστά και δεν σέβονται τη συμφωνία των Παρισίων. Ε, ήταν απέσια η στάση της Αυστραλίας στη Μαδρίτη. Παρακαλώ λοιπόν όχι συμφωνίες αν οι άνθρωποι αυτοί δεν αλλάξουν στάση και δεν θέλουν να σεβαστούν τη συμφωνία που υπεγράφει στο Παρίσι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Χαϊσέλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όντως όντως αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο, την πιο καταστροφική δασική πυρκαγιά που έχει φανεί ποτέ. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά. Ε, πρόσφατα στον Αμαζόνιο είχαμε παρόμοια φαινόμενα και πριν από αυτό τεράστιε τεράστιες πυρκαγιές στη Σιβηρία. Ήφτασε η αποκάλυψη. Και είναι καλό που έχουμε τον Green Deal μπροστά μας, αλλά χρειάζεται και άλλοι μεγάλοι παίκτε να συνταχθούν μαζί μας. Οι Κινέζοι, οι Αμερικάνοι, οι, Βραζιλιάνοι, οι Αυστραλοί, ε, είναι δημοκρατικά καθεστώτα με τους οποίους ε, διαπραγματευόμαστε εμπορικές συμφωνίες. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι οι δημοκράτες σημαντικοί παίκτε από αυτού να συμμαχήσουν μαζί μα και να μειώσουμε όσο μπορούμε τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, ίσως κατά 10%. Διαφορετικά να δημιουργήσουμε ε, μια ισχυρή διπλωματία και να πιέσουμε, γιατί διαφορετικά θα καταστρέψουμε τον πλανήτη για όλου μα. Είναι πολύ καλό που θα διαπραγματευτεί μαζί του η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα τους βοηθήσει, αλλά αφού τους βοηθήσουμε θα πρέπει να τους πιέσουμε στην Αυστραλία να αλλάξουν στάση. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο η κυρία Ward. Για ένα λεπτό. Το θέαμα αυτών των πυρκαγιών όλους μας τρομοκράτησε και το Δεκέμβριο του 2015. Είχαμε στην ε, Κάμπρια, την περιφέρειά μου, φοβερές ε, πλημμύρες. Ε, πρόκειται για φυσικά φαινόμενα, όντως, αλλά ο βαθμός στον οποίο αυτά σοβούν στέλνει να μην το είναι πραγματικό γεγονός η αλληλεγγύη του κλίματος, χτυπάει τον κόσμο παντού και όπως πολλοί από εσά θυμάμαι ένα ε, ντοκιμαντέρ που έλεγε πώς σκοτώνονται έτσι τα ζώα, τι γίνεται με ε, τα παγόβουνα και έχουμε πάρα πολλούς και το UKIP που αρνούνται την άνοδο της θερμοκρασίας. Είδατε τι λέει το κόμμα του Brexit, του που πήγανε τώρα, τι λένε συντηρητικοί θα πρέπει να ανησυχήσουμε για την πολιτική των συντηρητικών στην Αγγλία για το περιβάλλον. Ο κύριος Πισμόκ επίσης ε, έχει οργανώσει αυτά τα δίκτυα, ε, έχει ε, εκθέσει και αποκαλύψει το τι κάνει με διάφορες οργανώσεις και λόμπι ο Μπόρις Τζόνσον, η πρόεδρος. Και πάλι ο Αντιπρόεδρος Σεύτσοβιτς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Ναι, πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Κάτι το, δραματικό και εντυπωσιακό για την πρώτη συνεδρίαση με την καινούργια χρονιά. Αλλά όπως σας είπα και στην αρχή, Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι έχουμε πει ότι θα βοηθήσουμε την Αυστραλία. Θα είμαστε αλληλέγγυοι ακριβώ όπως τόνισε η κυρία Σόιντροβα. Είναι σημαντικό αυτό το μήνυμα να φτάσει παντού. Στην χώρα που τώρα έχει πληγεί από αυτό το οποίο έγινε τονίσατε ότι αυτά τα πηγαίνοντας στην Αυστραλία είναι συνέπεια της ε, αλλαγής του κλίματος σε όλο τον πλανήτη. Πρόκειται για μια ε, κατάσταση που εμείς οι άνθρωποι την δημιουργήσαμε. Άρα χρειάζεται να προσπαθήσουμε εμείς όλο τον κόσμο για να κάνουμε κάτι. Και η κυρία Τάλη, ο κύριος Μπιζού και άλλοι ε, είπαν ότι θα πρέπει η Επιτροπή αλλά και όλοι οι εταίροι μας όλο τον κόσμο κάτι να κάνουμε. και να είμαστε συνεπείς στην περιβαλλοντική μας πολιτική. Να εξασφαλίσουμε την παγκόσμια εφαρμογή όλων των ε, ισχυρών χωρών. Ε, ε, η Συμφωνία των Παρισίων είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει η μετάβαση στην Ευρώπη, αυτό να γίνει με δίκαιο κοινωνικά τρόπο, να δείξουμε ότι είναι δυνατόν να περιορίσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου και αυτό θα γίνει, να γίνει πάντων με δίκαιο τρόπο. Θα πρέπει βέβαια όλος ο κόσμος να ακολουθήσει του ίδιου ρυθμού όπω ε, να βρούμε νέου μηχανισμού που να σπρώξουν τι χώρε στην κατεύθυνση, ακόμα και αν καταρχήν δεν έχουν ανταποκριθεί, αλλά να έχουμε μηχανισμού όπως ε, το μηχανισμό προσαρμογή των εκπομπών του άνθρακα, <clears throat> ούτω ώστε η βιομηχανία να είναι καθαρή από τέτοιες εκπομπές. Να κάνουν και άλλοι αυτό που κάνουμε και εμείς. Βέβαια οι τραγωδίες από την αλληλή του κλίματος είχαμε και στην Ευρώπη. Δεν την γλιτώσαμε. Θυμηθείτε τα τραγικά γεγονότα αυτά που θυμήσατε τις πυρκαγιές στην Πορτογαλία, στην Σουηδία και στην Ελλάδα. Όχι, δεν θα κάνουμε πίσω. Θα είμαστε σε ετοιμότητα. Όλο ένα και περισσότερο κάθε χρόνο. Οπότε θα εξασφαλίσουμε την βελτίωση της διαχείρισης των δασών, καλύτερους μηχανισμούς αντιμετώπισης των ε, πυρκαγιών και πρόληψη αυτών και επίσης τα άμεσα μέτρα να συνδυαστούν με μακρόπνες προσπάθειες προσαρμογής. Η στρατηγική της Ένωσης που αφορά αυτήν την πολιτική που έχει ορίσει το 2030 είναι για να έχουμε περισσότερη ανθεκτικότητα στο μέλλον, να εντοπίσουμε τις επιπτώσεις αλλαγής του κλίματος και ιδίω αυτό εκεί που τα πράγματα είναι πιο ευάλωτα όπως ας πούμε σε σχέση με τα δάση. Νέα στρατηγική. Ε, για μας είναι σημαία τα σχετικά προγράμματα όπως και για σας ε, και συγκεκριμένα το New Green Deal. Αναφερθήκατε και στο πρόγραμμα Κοπέρνικος. Εμείς είμαστε η βασική παροχή για τα σχετικά δεδομένα, ούτως ώστε να τρέχει το πρόγραμμα και έτσι να καταπονούμε τις πυρκαγιές από Καλιφόρνια μέχρι η Αυστραλία οπότε θα αναπτύξουμε περαιτέρω το σύστημα και τα συστήματα της προειδοποίησης ε, και το σύστημα για τις στην Ευρώπη πολύ σημαντικό αυτό για την κλιματική κρίση όπως ελέγχθη βελτιώσαμε την πολιτική προστασία αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο και σύμφωνα με την κυρία Μίλλερ τον κύριο Κόκαλη επίσης ότι θα πρέπει παγίως να αναζητούμε τρόπους για να βελτιωθούμε όσον αφορά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών για κάθε τέτοια, κάθε κατάσταση που μπορεί να έρθει. Η καλύτερη αντίδραση για αυτή την κρίση είναι το να προσέξουμε, να είμαστε αποφασιστικοί όσον αφορά το New Green Deal και έτσι να δείξουμε και στον υπόλοιπο κόσμο ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, ξέρουμε πώς να τα καταφέρουμε και ότι είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την εμπειρία μας μαζί τους. Και βέβαια για τις προσπάθειές μας υπολογίζουμε στην βοήθεια του Κοινοβουλίου. Και σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, εμείς ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρο. Κλείνει εδώ η συζήτηση και πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης ε, δήλωση της Επιστροπής ε, για το διασυνεριακό οργανωμένο έγκλημα και τις επιπτώσεις του στην ελεύθερη κυκλοφορία. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να ζητήσετε κατσδιά και μπλε κάρτες χρησιμοποιώντας τόσο τον ε, συνηθή τρόπο εγγραφής όσο και το ηλεκτρονικό σύστημα. τη οδηγίες θα τις βρείτε στην είσοδο του ημικυκλίου. Δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντιπρόεδρε Σεφτσοβιτς, έχετε το λόγο και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Από το ένα δύσκολο θέμα περνάμε στο επόμενο. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, διότι το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ. Το διασυνοριακό έγκλημα, το οργανωμένο έγκλημα επηρεάζει τι ζωέ και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, την οικονομία τη Ευρώπη, την εμπιστοσύνη τη κοινωνία στου θεσμού. Η αξιολόγηση του οργανωμένου εγκλήματος το 2017 στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι πάνω από 5.000 ε, ομάδες οργανωμένου εγκλήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί αύξηση άνω του 15% σε σχέση με τα νούμερα του 2013. Τα κέρδη τους εκτιμώνται σε 110 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, μόνο το 1% αυτών των κερδών κατασχόνται η δυσκολία δημιουργίας μιας ολιστικής ε, ολοκληρωμένης προσέγγισης ε, νομοθετικά και επιχειρησιακά είναι αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα για να καταπολεμήσουμε τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος. Ε, πρέπει να δείξουμε θάρρος για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά. Είχαμε κάνει έκκληση για μια στρατηγική για το οργανωμένο έγκλημα και την διαφθορά. Τα αναφέραμε ως ευρωπαϊκά προβλήματα που απαιτούν ευρωπαϊκές λύσεις. Έτσι λοιπόν καλωσορίζω την πολύ επίκαιρη συζήτηση αυτή. Το 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ένα νομικά δεσμευτικό όργανο που απαιτεί από τα κράτη-μέλη να θέσουν εκτός νόμου την συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, να την ποινικοποιήσουν. Τότε παρατηρήθηκαν κάποιες ελλείψεις ε, όπως η μη εναρμόνιση του ορισμού του παραπτώματος, ε, τη συμμετοχή ε, του εγκλήματο, ε, τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, το οποίο σημαίνει στην πρακτική ότι πολλά κράτη-μέλη δεν ποινικοποιούν την απλή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Απαιτούν αντιθέτω να αποδειχθεί εγκληματική πράξη. Εμεί ω νομοθέτε πρέπει να κλείνουμε παραθυράκια. Είναι καθήκον μα στην νομοθεσία μια επόμενη μελέτη θα γίνει για αυτό το ζήτημα για το οργανωμένο έγκλημα πολύ ε, σύντομα. Το να ακολουθούμε το χρήμα πρέπει να είναι ε, η γραμμή που θα ακολουθούμε για το οργανωμένο έγκλημα. Η οδηγία για την πρόσβαση των αρχών επιβολή του νόμου σε οικονομικέ πληροφορίε θα τεθεί, τέθηκε σε ισχύ 1η Αυγούστου του περσινού έτου. Ε, μπορεί να χρειαστούν επιπλέον μέτρα, ούτω ώστε οι αρχέ επιβολή του νόμου να μπορούν να πραγματοποιήσουν αποτελεσματικέ έρευνε διασυνοριακά να διαπιστώνουν την διασύνδεση ε, τις διασυνδέσεις και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση οι αρχές επιβολής του νόμου για να μπορούν να πραγματοποιούν τις έρευνες. Γραφεία κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων έχουν δημιουργηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη και η οδηγία για τις σχετικές διαδικασίες ε, κατάσχεσης και ε, δέσμευσης ε, των εσόδων και των περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από κλιματικές δραστηριότητες έχουν εναρμονιστεί, εναρμονιστεί πλέον σε όλη την Ευρώπη. Η δέσμευση και η δίμευση ισχύουν από το θα ισχύσουν από τον Δεκέμβριο του 2020 συμπληρωματικά προς το νομοθετικό πλαίσιο, ωστόσο πρέπει να γίνουν περισσότερα. Η κατάσχεση του 1% δεν είναι τίποτα η Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να παρουσιάσει μια έκθεση για την υλοποίηση της ε, οδηγίας ε, ε, κατάσχεσης που θα μας βοηθήσει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ιχνηλάτηση, την κατάσχεση και τη δίμευση των περιουσιακών στοιχείων που προερχόνται από κλιματικέ δραστηριότητε. Υπάρχει ένα έγγραφο που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο, η έκθεση του 2017 της Ευρωπόλ έδειξε πώς η διαφθορά βοηθά το έγκλημα η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2019 έδειξε σημαντική αύξηση στα ανώτερα επίπεδα και στι θετικέ δραστηριότητε ε, των εγκληματικών ομάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει τα κράτη-μέλη να εξοπλιστούν κατάλληλα για να καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Η ικανότητα καταπολέμηση διαφθορά θεωρείται ότι είναι μια από τι βασικέ πτυχέ του νέου κράτου δικαίου και του νέου κύκλου ε, αναθεώρησης για το κράτο δικαίου που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2020 θα χρειαστεί να συμμετέσχει και η αρχή ε, που βοηθά ε, στην ελεύθερη κυκλοφορία ε, να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να δημιουργηθούν συνέργειες, να υπάρξει συνεργασία με άλλους οργανισμούς όπως η Ευρωπόλ και η Eurojust στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την εμπορία ανθρώπων. Η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως την προσέγγιση της Ευρωπόλ για την καταπολέμηση των εγκληματικών ομάδων με την ε, εξουδετερώση των βασικών φορέων, ε, των βασικών παικτών. Θα πρέπει να κατασχεθούν τα παράνομα ε, περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτήσει τέτοιοι εγκληματίες. Οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα θα πρέπει να συμπληρώνει τον κύκλο πολιτική ε, για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματο. Η καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών θα είναι προτεραιότητα για την επόμενη Επιτροπή. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθηση ε, Ναρκωτικών ε, και εθισμού στα ναρκωτικά δείχνει ότι αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία μα. Οι ποσότητε ηρωίνη και κοκαίνη που έχουν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανευπροηγουμένου και σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης η παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών αυξάνεται. Η σημερινή στρατηγική για τα ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελειώνει και θα πρέπει η Κομισιόν να εξετάσει τι νέα δράση απαιτείται δεδομένου του επίγοντος της κατάστασης αυτής. Το impact, ο νέο ε, κύκλο πολιτική ε, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο έχει αλλάξει τον τρόπο συνεργασία των κρατών μελών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο, για την ε, περίοδο 2018-2021 υπάρχουν 10 προτεραιότητες μεταξύ των οποίων το κυβερνοέγκλημα, η διακίνηση ναρκωτικών, η διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης, η εμπορία ανθρώπων. Είναι μόνο μερικά από αυτά οι αριθμοί. Είναι συγκλονιστική. Το 2018 η εμπορία ανθρώπων ε, ε, για την εμπορία ανθρώπων έγιναν 1.200 έρευνες με πολλούς ε, χιλιάδες ανθρώπους ε, που ανακρίθηκαν ε, και πολλές συλλήψεις στο απάτη στο φόρο καταναλώσεις. Ε, πολλά εκατομμύρια ευρώ φοροδιαφυγής ε, προλήφθηκαν. Βλέπουμε λοιπόν ότι η δυσκολία είναι τεράστια. Το πρόβλημα είναι τεράστιο και αυτό πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφού είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Πρέπει να βρεθεί ευρωπαϊκή απάντηση λοιπόν. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω να ευχαριστήσω την κυρία Πρόεδρο που ε, πρότεινε αυτό το θέμα για τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Θα ακούσουμε πολύ προσεκτικά τι απόψει των αξιότιμων μελών και θα επανέλθουμε με συγκεκριμένε προτάσει στο μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Τώρα εκ μέρου των πολιτικών ομάδων από το ΕΛΚ θα δώσω το λόγο για δύο λεπτά στον κύριο Τομπέ. Έχετε το λόγο. Ε, ε, Αγαπητέ κύριε Σεύκοβιτς, η βία η οποία σχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό για την Ευρώπη. Και στη δική μου τη χώρα, τη Σουηδία, η κατάσταση έχει ε, κλιμακωθεί γιατί πέρσι 40 άτομα ε, πυροβολήθηκαν, ε, έγιναν 200 εκρήξεις και είδαμε πιο πολλά από αυτά τα επεισόδια να σημειώνονται στην πόλη του Μάλμο μία γυναίκα σκοτώθηκε την ώρα που είχε στα χέρια της το παιδί της. Πυροβολήθηκε. Αυτά λοιπόν τα επεισόδια είναι πια τόσο συχνά στη Σουηδία που η κυβέρνηση της Δανίας χρειάστηκε να βάλει ε, ελέγχου στα σύνορα με τη Σουηδία έτσι ώστε να προστατεύσει τους πολίτες της. Τώρα δεν είναι η εποχή ε, της άρνησης και της υποβάθμισης των προβλημάτων ε, με, το έγκλημα των συμμοριών στην Σουηδία. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και σε εσωτερικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να έχουμε περισσότερη ασφάλεια στην Ευρώπη έτσι ώστε να ε, λειτουργήσει και η ελεύθερη μετακίνηση μεταξύ Δανίας και Σουηδίας. Είναι τραγικό να βλέπει κανείς πως ε, οι σοσιαλδημοκράτες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπάθησαν να μειώσουν ε, τη σημασία του φαινομένου. Δεν θέλουν να το συζητήσουμε και θα πρέπει να φανούμε πιο όριμοι. Είναι πρόβλημα για τη Σουηδία, αλλά είναι πρόβλημα και για όλη την περιοχή και θα έλεγα και για όλη την Ευρώπη. Παρακαλώ λοιπόν να παρουσιάσετε τρεις προτάσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Europol περισσότερους πόρους και θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στη Σουηδία. Και επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσετε πως θα ε, καταπολεμήσετε το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Επίσης θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να απελάσουμε ε, τα μέλη των συμμοριών ακόμα και αν είναι με ε, Ευρωπαίοι πολίτες. Μαζί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να αυξήσουμε την ασφάλεια στην Ευρώπη και στη Σουηδία. Ευχαριστώ. Thank you very much. Now, on of... Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 1,5 λεπτό η κυρία Φρίτσον έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε. Το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικά όλο και περισσότερο έχει γίνει περίπλοκο και πιο διασυνοριακός ο χαρακτήρας και χρειαζόμαστε και διασυνοριακή λύση συνεπώς. Εμείς οι δημοκράτες πιστεύουμε ότι αυτό το θέμα είναι σημαντικότατο και το παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Στις χώρες μας θα πρέπει πραγματικά να αυξήσουμε τα μέτρα μας, να καταπολεμήσουμε το έγκλημα αλλά και τι ρίζε του εγκλήματο, τα αίτια του εγκλήματο. Και πράγματι αληθεύει, η κατάσταση είναι άκρο ανησυχητική σε πολλέ από τι χώρε μα και πολλέ από τι πόλει μα. Το Μάλμο είναι μια πόλη που ξέρω πολύ καλά. Είναι μια υπέροχη, φανταστική πόλη. Ταυτόχρονα όμω είναι μια πόλη που έχει πληγεί σκληρά από τη βία και από πυροβολισμού. Και αυτό είναι γεγονό. Το βλέπουμε αυτό, αλλά μπορούμε να δούμε επίση ότι η κυβέρνηση κατέβαλε προσπάθειε, η σουηδική κυβέρνηση κατέβαλε προσπάθειε και αυτό έχει δώσει καρπού. Δείτε τα στατιστικά των αστυνομικών αρχών τα πρόσφατα. Είδαμε μια μείωση του αριθμού των πυροβολισμών και νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά σημαντική δουλειά. Ε, το τελευταίο επεισόδιο στη Σουηδία ήταν στο Στοκχόλμη. Ε, στην πατρίδα του κυρίου Τομπία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό πραγματικά να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν ευθύνη ε, να επομιστούν χρειάζεται συνεργασία και χρειάζεται και συνεργασία μεταξύ Σουηδία και Δανία, αλλά χρειάζεται και μεγαλύτερη προσπάθεια πλευρά του Europol, χρειάζεται αποτελεσματικότερη συνομική συνεργασία, θα πρέπει να έχουμε ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των χωρών μα. Θα πρέπει να πούμε εμεί οι Δημοκράτε ότι πάντα θα πολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα, πάντα θα το πολεμάμε, πάντα διότι οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα πρέπει να μπορούν να ζουν σε ασφάλεια στι μεγάλε αστικέ περιοχέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκ μέρου τη ομάδα New Europe, η κυρία Καλσμπρού. Για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η ασφάλεια είναι η ελευθερία. Όταν δεν αισθανόμεθα ασφαλής, η πραγματικότητα συρρυκνούται και κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Εμείς στη Σουηδία με θλίψη ακούσαμε για διάφορα φρικτά εγκλήματα που διεπράχθησαν το τελευταίο έτος και σχετίζονται με την αύξηση της εγκληματικότητας. Ανάμεσα στα θύματα ήταν μια έγκυος μητέρα η οποία πυροβολήθηκε σε ένα δρόμο. Πρέπει να εγγυθούμε την ασφάλεια των ανθρώπων. Αυτό είναι βασικό στοιχείο καθήκον για κάθε κράτος μέλος. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί το έγκλημα και να προληφθεί. Όμως επί μακρόν υποτιμούσαμε το πώς εγκληματικότητα ε, και τα ναρκωτικά έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και ρέουν σε διασυνοριακό επίπεδο. Δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό. Η ελευθερία τη κίνηση θα πρέπει να αυξήσει την ελευθερία μα. Δεν θα πρέπει αντιθέτω να αποτελεί δικείμενο κατάχρηση και να καταστρέψει την ελευθερία μα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνεργασία διασυνοριακή. Η συνεργασία αστυνομική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Europol, είναι πολύ αδύναμη και δεν έχει επιχειρησιακέ εξουσίε. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και αν θέλουμε πραγματικά να πνίξουμε το διασυνοριακό έγκλημα, θα πρέπει να αυξήσουμε τι εξουσίε που δίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι φιλελεύθεροι θα θέλουν να δουν μια ανάπτυξη τη Europol, να γίνει μια ευρωπαϊκή FBI, ένα ευρωπαϊκό FBI, να έχει επιχειρησιακέ δυνατότητε και να μπορεί να ασκεί δική του δράση με διασυνοριακέ συμμορίε. Το ε, ΕΛΚ και οι μετριοπαθεί τη Σουηδία πήραν μια πρωτοβουλία για τη συζήτηση και λέω ότι είναι κατεπήγον θέμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θα πρέπει να δούμε τι πράγμα κουβεντιάζουμε. Θα πρέπει να συζητήσουμε τις λύσεις. Αυτό απαιτεί πόρους και αυτό απαιτεί νέους τρόπους ε, συνεργασίας. Ελπίζω ότι όλα τα κόμματα εδώ απόψε είναι έτοιμα να αυξήσουν τη συνεργασία τους κατά του διασυνοριακού εγκλήματος και αυτή η συζήτηση να μην είναι μόνο κενός λόγος. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και για την ανθρώπινη ελευθερία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της ομάδας των Πρασίνων για ένα λεπτό, η κυρία Όκεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον Επίτροπο. Σας ευχαριστώ για την απάντηση, ήταν πολύ ικανοποιητική. Θέλω να δω το θέμα από άλλη οπτική γωνία, διότι τα μέσα που υθετούμε σε πολλές χώρες, όπως και στη Δανία, ήταν η συνοριακή έλεγχη. Και η συνοριακή έλεγχη μπορεί να είναι χρήσιμη σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά ε, είναι πολύ επαχθές μέτρο. Ευτυχώ, ο μεθοριακό έλεγχο μεταξύ Σουηδία και Δανία δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν ενοχλούμε του πολίτε όπω κατά το παρελθόν. Και πάση περιπτώσει, οι μεθοριακοί έλεγχοι δεν βοήθησαν πολύ. Και έχουμε μεθοριακού ελέγχου και στα σύνορα Δανία-Γερμανία. Φέτο έχουμε την εγκοτατεία από την Ένωση τη ε, ε, Νότια Δανία με τη Δανία και το γιορτάζουμε και χαιρόμαστε που δημιουργήσαμε αυτή την υπέροχη δυσυνορική συνεργασία στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι οι δανέζικε αρχέ θεσπίζουν μεθοριακού ελέγχου. Αυτό είναι σπατάλι χρημάτων, είναι κάτι που εμποδίζει την κίνηση των πολιτών μα. Παρ' όλα αυτά, όμω, έγινε. Είναι εξίσου ανόητο μέτρο όπω εκείνοι οι φράχτε που έχουν χτιστεί. Μα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνουν καμία διαφορά αλλά είναι μια απόπειρα να δημιουργηθούν κάποια σύμβολα που δίνουν την εντύπωση ότι κάτι γίνεται. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλή πρόταση. Ευχαριστώ εκ μέρου του ID. Για ένα λεπτό, ο κύριος Χακαράινεν έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, η ελεύθερη μετακίνηση οδηγεί στην ε, υπέρβαση των συνόρων από πλευρά του οργανωμένου εγκλήματος. Το οργανωμένο εγκλήμα μετακινείται όπως θέλει. Και όταν δεν υπάρχουν πλέον εμπόδια για το οργανωμένο έγκλημα, ουσιαστικά ο καθένας μπορεί να πάει όπου θέλει. Ως εγκληματίας, ως μετανάστη. Και πώς αντιδρά λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση στο φαινόμενο με αυτό λέει καλώς ορίσατε, περάστε. Πλήρη πρόνοια να σας δώσουμε. Πώς να σας βοηθήσουμε. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση. Χρειαζόμαστε μια άμυνα. Αυτό το εξασφαλίζαμε με τα σύνορα. Πιστεύουμε ότι η πολυπολιτισμικότητα με τη μορφή που λαμβάνει η χώρα σήμερα στην ε, Μέση Ανατολή και στην ε, Αφρική Ποιο πιστεύει ότι αυτό δεν αποτελεί κίνδυνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ από την ομάδα του ECR, ο κύριο Βέιμερς. Για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Η δανεική κυβέρνηση των Σοσιαλδημοκρατών ε, εισήγαγε μεθοριακούς ελέγχους στα σύνορα με την Σουηδία γιατί τους απασχολεί το οργανωμένο έγκλημα και οι Ισλαμιστές στη Σουηδία μετά την, τον βομβαρδισμό των ε, κτηρίων, των κυβερνητικών κτηρίων της Δανίας, οι Σουηδοί σοσιαλδημοκράτες δεν μπορούν καν να εκδώσουν οι μάμητες που έχουν εξακριβωμένους συνδέσμους με το τρομοκρατία και έχουμε μόνο το 2019 πάνω από 200 βόμβες και χτες ακόμα δύο βόμβες στην Ούψαλα Θέλουμε λοιπόν να ξέρουν όλοι οι Σουηδοί ότι η επικέντρωση των σοσιαλδημοκρατών για σήμερα για το οργανωμένο έγκλημα δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την αύξηση του κατακεφαλή ποσοστού των βομβαρδισμών ε, στην Σουηδία σε ποσοστά ανάλογα με το Μεξικό. Να πούμε λοιπόν στους ε, σοσιαλδημοκράτες, στους Δανούς, να πάνε στην Κοπεχάγη να διδαχθούν από τους Δανούς, γιατί επί σειρά ετών καταδικάζατε τους ε, Δανούς ως ξενόφοβους. Αλλά ίσως τελικά μπορείτε κάτι να μάθετε για αυτούς και πάνω απ' όλα η μετανάστευση. Όταν τα πράγματα πάνε άσχημα, ακόμα και στη Σουηδία, ξέρουμε ότι πραγματικά πηγαίνουν άσχημα τα πράγματα. Ας σταματήσουμε να ασκούμε πιέσεις, λοιπόν, ε, στις ε, αρχές επιβολής του νόμου. Θα πρέπει να είναι εξάρτητες. Θα πρέπει να μην ασκείται πίεση σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των εκθέσεων τους. Και θα πρέπει η αστυνομία να μπορέσει να δείξει στις συμμορίες αυτές ποιος είναι τελικά ο αρμόδιος. Να γίνει ένα ξεκαθάρισμα στους αυτού αυτούς μάμιδες που μισούν την Σουηδία. Και αν αρχίσουμε να είμαστε ειλικρινεί με τον λαό τη Σουηδία. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, α παρατηθούμε λοιπόν. Ευχαριστώ για ένα λεπτό από τους μη εγγεγραμμένους, ο κύριος Τόπνη. Ευχαριστώ. Το 1992 οι Ευρωπαϊκοί ηγέτες μαζεύτηκαν και υπεγράψαν την πιστοποιητικό γέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή τη φρικόδη συνθήκη που ουσιαστικά ήταν και η καταδίκη σε θάνατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς, λοιπόν, καταδικάζεται την συνθήκη αυτή γιατί αρνείστε τη δημοψήφισμα από τους Βρετανούς και στη συνέχεια ο Τόνι Μπλερ υπογράφει για την διεύρυνση με 10 ευρωπαϊκά κράτη και πάλι δεν ζητήθηκε η το γνώμη του Βρετανικού λαού. Και τελικά καταλήγουμε να πλημμυρίζεται η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου από εκατομμύρια α, μετανάστες για λόγους εργασιακούς. Και έτσι λοιπόν ήταν ήδη εκεί τα ψήγματα του Brexit που ε, μέλουν να καταδικάσουν και να καταστρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν ε, το 2015 δόθηκε ε, καθεστώς άσυλο σε εκατομμύρια μετανάστες και ετούντες άσυλο, επιτέλους οι Βρετανοί αντίδρασαν και χτες ζητήθηκε να υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση ως τμήμα του Brexit. Κύριε Μπαρνιέ, αυτό που έχω να σας πω Αφίντερζεν και εδώ πέρα η πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Ζητώ συγγνώμη. Δεν έχετε άλλο χρόνο. Επόμενο ομιλητής για ένα λεπτό, ο κύριος Σαρσαλέχος. Κυρία Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η συζήτηση. Είναι η μοναδική γνωστή περίπτωση κατά την οποία θεσπίζονται εκ νέου έλεγχοι στα σύνορα λόγω κλιμάκωσης οργανωμένου και βίου εγκλήματος. Η διασυνοριακή εγκληματικότητα θα έχει ως μόνη απάντηση τη διασυνοριακή συνεργασία και όταν πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία, τα σύνορα δεν προστατεύουν την εθνική κυριαρχία. Τα σύνορα προστατεύουν μόνο τους παραβάτες, τους εγκληματίες. Η Ευρώπη πρέπει να πρέπει να είναι ένας χώρος ελευθερίας για τους πολίτες της και όχι ένας χώρος κινητικότητας για τους παραβάτες. Γνωρίζουμε τα προβλήματα, γνωρίζουμε τι οφείλουμε να πράξουμε. Να μιλήσουμε για πιο αποτελεσματική δίμευση και πάγωμα στοιχείων ενεργητικού, για έλεγχο της νομιμοποίησης παράνομος προσόδων, για πρόσβαση στις δικαστικές διαδικασίες, για εναρμόνιση, εναρμόνιση των νομοθεσιών, για συνεργασία ε, με τα εργαλεία σύλληψης και παράδοση των υποδίκων, δηλαδή πρέπει οι πράξεις μας να ακολουθούν κατά γράμμα τα λόγια μας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής για 1,5 λεπτό, η κυρία Σαλντεμόζε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μας παρουσιάσατε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Προκλήσεις όλο ένα και πιο σημαντικές, όλο ένα και πιο απαιτητικέ. σε ό,τι έχει να κάνει με την εγκληματικότητα, το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ που μας είπατε τι πρέπει να κάνουμε και στο μέλλον. Συμφωνώ απολύτω γιατί πρέπει να πράξουμε πολύ περισσότερα πράγματα ώστε να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια ο Ευρωπαίος πολίτης. Το οργανωμένο έγκλημα έχει πολύ σοβαρές, πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Δεν έχουμε κανένα φόβο. Γνωρίζουμε τις προκλήσεις. Θέλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Είδαμε την ένταση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Σουηδική κοινωνία αλλά και οι υπόλοιπε σκανδιναβικές χώρες. Και αυτό ισχύει και στις δικές μας χώρες επίσης. Πρέπει να συνεργαστούμε. Πρέπει να είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε. Ε, το έχουμε πράξει. Η Δανία και η Σουηδία συνεργάζονται ήδη. Και το έχουμε κάνει γιατί θέλουμε να θετήσουμε ένα κοινό τρόπο δράσης για την καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος. Θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων μόνο αν δράσουμε από κοινού, όλοι μαζί. Ίσως θα πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα, όχι μόνο η έλεγχη στα σύνορα, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το θέμα. Εμείς αναλάβαμε δράση και περιμένω με μεγάλη αγωνία και με μεγάλη ανυπομονησία να δω τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους επόμενους μήνες για να βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση στη Δανία, στη Σουηδία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Παγκασάρου Ουρτουντούα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία ε, Πρόεδρε. Επίτροπε Σεύκοβιτς, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, το οργανωμένο έγκλημα τον 21ο αιώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κλίμα της διαφθοράς, το ε, έγκλημα της διαφθοράς, ε, το οργανωμένο έγκλημα, το έγκλημα εναντίον των κρατών έχει φτάσει σε επίπεδα πολύ ψηλά, πολύ εκλεπτισμένα, πολύ ανεπτυγμένα. Είναι απαραίτητο να έχουμε μεγαλύτερη δικαστική και αστυνομική συνεργασία. Πρέπει να εναρμονιστούν οι ορισμοί των αδικημάτων και αυτό θα είναι καθοριστικό για τη βελτίωση τη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολή του νόμου, δικαστικών και αστυνομικών. Διότι, ιδαλλιώ, όσοι παραβάτε έχουν και τα μεγαλύτερα οικονομικά μέσα, αυτοί θα ξεφεύγουν από την δικαιοσύνη, θα παίζουν με τα δικαστικά συστήματα και θα επιτυχάνουν την ασυλία και την ατιμορρησία του δηλαδή. Έχουμε πολύ σοβαρά δικήματα από το οργανωμένο έγκλημα που στρέφονται ενάντια ενάντια στο, κάθο, στο κράτος δικαίου και αξιοποιούν ε, τις γκρίζες ζώνες του κάθε δικαστικού συστήματος και χειραγωγούν ε, τις διάφορες διατάξεις και υποπεριπτώσεις για να ξεκλειστρήσουν από τα χέρια των αρχών, ε, από την αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Το είπατε κι εσείς, ότι πρέπει να είμαστε πολύ καλά εξοπλισμένοι, να βασίζεστε στη δική μας βοήθεια για να καταπολεμήσουμε όλο αυτό το φαινόμενο. Θα έχετε την αμέριστη στήριξη και συμπαράστασή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για ένα λεπτό. Η κυρία Τόμασιτς έχει το λόγο. Σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει, περίπου 90% των παράνομων μεταναστών έρχονται στην Ευρώπη, που έρχονται στην Ευρώπη ήρθαν σε επαφή με διακινητές που τους μετέφεραν για ένα τμήμα της διαδρομής τουλάχιστον. Είναι σαφές από την πρώτη μέρα ότι η ανοχή όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση ενισχύει αυτό το είδος του οργανωμένου εγκλήματος και άλλες μορφές αυτού, όπως είναι η πορνεία, το ελευθερμπόριο ναρκωτικό, το εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων, η τρομοκρατία. Είναι κατανοητό ότι θέλουν απελπισμένα να βρουν λύσει οι άνθρωποι. Για να... Αυτοί οι άνθρωποι, μάλλον, έρχονται στην Ευρώπη να βρουν μια καλύτερη ζωή. Δεν είναι όμω ε, κατανοητό το να θέτουν σε κίνδυνο με τη συμπεριφορά του αυτού ε, ε, αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται που κάνουν παρανομίες και έρχονται άλλοι παράνομοι μετανάστες και δημιουργούνται και νέα παιδεία για τον παράνομο κόσμο. Θα πρέπει να θέσουμε κάποια τάξη στην Ευρώπη προ όφελο όλων των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και εκείνων που θέλουν να γίνουν πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να είναι πραγματικά ενταγμένοι οι νέου ερχόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να σέβονται τα σύνορά μα, του νόμου μα και τον τρόπο διαβίωσή μα, τη ζωή μα. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό, ο κύριο Χιτβέγγι έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα είναι ο μεγάλος αριθμός βιαίων εγκλημάτων που διαπράττονται στη Σουηδία, στο Μάλμο και άλλες πόλεις που έφτασαν σε τέτοιο επίπεδο που οι πολίτε τώρα πρέπει συνεχώς να ζουν υπό το φόβο. Αυτό είναι πονίδιστο και εξωφρενικό. Η προσπάθεια τη ελίτη αριστεράς και του τύπου είναι να καλυφθεί ε, το υπόβαθρο αυτού του φαινομένου. Ξέρουμε ότι το 2015 η Σουηδία έχει δεχτεί τους περισσότερους μετανάστες κατά αναλογία του πληθυσμού. Έκτοτε, ο αριθμός των εκρήξεων, των πυροβολισμών, βιοπραγιών και παρενοχλήσεως γυναικών έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Η, η είσοδο των μεταναστών ήταν κάτι καταστροφικό στη Σουηδία και δεν έχουν ενταχθεί καθόλου. Είναι εξωφρενικό το πώ η Σουηδική και η Ευρωπαϊκή Αριστερά κάνουν τα πάντα για να αποκρύψουν αυτά τα στοιχεία. Το πραγματικό πρόβλημα με το κάτω δικαίου είναι όταν μια χώρα δεν μπορεί να προστατεύσει του πολίτε τη πλέον και ο τύπος δεν παρουσιάζει την πραγματικότητα αλλά γίνεται εργαλείο της αριστερής ε, δικτατορίας όσον αφορά τη διαμόρφωση της γνώμης. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά, η κυρία Φαγιών έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο χώρος ε, Σέγγεν, χωρίς εσωτερικά σύνορα, θα πρέπει να εγγυάται σε κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμα στην ελεύθερη διακίνηση και διαμονή είναι από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και είναι ένα στοιχείο της πραγματικής ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσωποποιεί τη συνεργασία, τη συμφιλίωση, την ειρήνη, την ανοχή, την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια. Και αυτό δοκιμάζεται πολύ σοβαρά τα τελευταία τέσσερα χρόνια και έξι από τα κράτη-μέλη που ανήκουν στο χώρο Σέγγεν έχουν, έχουν θεσπίσει και αυξήσει τους εσωτερικούς ελέγχους των συνόρων χωρίς νομική βάση. Πρέπει να διαρωτηθούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ήδη έχουμε φτάσει στο τέλος της εποχής του Σέγγεν. Ε, τι θα πρέπει να κάνουμε για να αναζωογονήσουμε τον χώρο Σέγγεν. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε κάποια μέτρα παραθέτοντας πράγματα, πάντα μάλλον το πρόβλημα του οργανωμένου εγκλήματος και τη δυσκολία καθορισμού ποσοστώσεων. Θα πρέπει να καθορίσουμε, να λύσουμε τα προβλήματα με ασφαλή εξωτερικά σύνορα, να καταπολεμήσουμε τους διακινητές και να βοηθήσουμε τις χώρες προέλευσης να επιλύσουν τα προβλήματα που είναι και η ρίζα των μεταναστεύσεων. Θα πρέπει επίσης να έχουμε καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δικαστικών μας φορέων και θα πρέπει να ενισχύσουμε και το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών μελών. Θα πρέπει επίσης να έχουμε περισσότερους σαφείς κανόνες για όλους, να είναι εύχριστοι οι κανόνες. Και στα εσωτερικά μας σύνορα αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση που δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε εδώ και μερικά χρόνια. Βέβαια, δεν θα μπορούμε πάντα να λύνουμε όλα τα προβλήματα ακόμα και όταν εφαρμόζουμε ελέγχους όλα μας τα σύνορα. Αλλά το πρόβλημα πιστεύω είναι η έλλειψη προθυμίας, πολιτικής βούλησης των ηγετών μας. Και αυτή είναι μια νέα πρόκληση για όλους μας. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στις διαπραγματεύσεις για αυτό το θέμα. Πριν είναι πολύ αργά. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό η κυρία Στρουγκάριο έχει το λόγο. Για να είμαστε ειλικρινείς, για κάποια πράγματα. Η καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια συντονισμένη δράση. Και η συνεργασία προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές ε, θα συνεργάζονται σωστά χρειάζεται απόλυτη εμπιστοσύνη. Το να κλείνουμε τα σύνορα δεν επιλύει τι αιτίε του προβλήματο. Ουσιαστικά μόνο το σύμπτωμα αντιμετωπίζει. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε ποιε είναι οι βαθύτερε αιτίε του προβλήματο. Κατά δεύτερον, το Σέγγεν αποτελεί έναν χώρο ελευθερία, μετακίνηση και ασφάλεια. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο αν αφενό οι εθνικέ αρχέ κάνουν τη δουλειά του και μάλιστα με πραγματικό τρόπο και αφετέρου αν υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή και πιο πολλή συμμετοχή σε ό,τι αφορά την νομοθετική δεν αρκεί να λαμβάνουμε μέτρα, όπως φάνηκε και στην ακρόαση της 3ης Δεκεμβρίου και όπως είπατε και εσείς άλλωστε κύριε Επιτροπέ. Θα πρέπει το θέμα της διασυνοριακής εγκληματικότητας να το κοιτάξουμε με πιο σοβαρό τρόπο. Δεν, μπορέσουμε, δεν θα μπορέσουμε. Γιατί Μάλλον δεν μπορούμε να δώσουμε ικανοποίηση σε αυτού που θέλουν να περιοριστεί η ελευθερία μετακίνηση. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ο κύριο Βόρμπορν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί πλέον ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώ η Σουηδία είναι το παράδειγμα προς αποφυγή. Η κατάσταση λοιπόν είναι τόσο σοβαρή που έχουν επανεισαχθεί συνοριακοί έλεγχοι από πλευρά τη Δανία. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στους μικρομεσαίους ε, επιχειρηματίες που ανησυχούν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ίδιο τη εγκληματικότητα αυτή, ε, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τους αγρότες, ε, του επιχειρηματίε, που αντιμετωπίζουν τέτοιε συμμορίε κάθε εβδομάδα. Αυτέ οι κλιματικές λοιπόν συμμορίε, οι οποίε ε, έχουν ως θέματα τους ε, εστιατόρε, απλού επιχειρηματίε. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να βοηθήσει, γιατί η Σουηδική κυβέρνηση των Σοσιαλδημοκρατών έχει χάσει τον ελεγχό τη στην κατάσταση. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται ε, στα Τελωνία, να ε, υπάρχει μεγαλύτερη επέκταση της, ε, των σχετικών ευρωπαϊκών υπηρεσιών και η ελευθερία μετακίνησης δεν πρέπει να ισχύει για τους εγκληματίες. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό, ο κύριος Κέρνερ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμε, κύριε Επιτροπέ, η ποινική δίωξη συχνά, ακόμα σήμερα, δυστυχώς έχει προβλήματα σε ό,τι αφορά τα σύνορα των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά η ευρωπαϊκή ενοποίηση προχωρά εδώ και καιρό και κάθε μέρα που δεν υπάρχει σωστή αστυνομική συνεργασία, κάθε μέρα που δεν υπάρχει σωστή εναρμόνιση στον ευρωπαϊκό χώρο, αυτό επιτρέπει στους εχθρούς της Ευρώπης να εκμεταλλεύονται τη βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ελευθερία ελευθερία μετακίνηση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πιο θαραλέοι, πιο τολμηροί ω Ευρωπαίοι και σε ό,τι αφορά θέματα δικαστική και αστυνομική συνεργασία, επιτέλου να προχωρήσουμε με αποφασιστικό τρόπο. Θα πρέπει να βγούμε εκτό των εθνικών νοοτροπιών. Χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό FBI, το οποίο θα καταπολεμά την ευρωπαϊκή, την, ε, το οργανωμένο εγκλήματο και χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των σχετικών αρχών. Αλλά κυρίω ένα πράγμα πρέπει να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε την ελεύθερα σύνορα στην Ευρώπη και την ελεύθερη μετακίνηση. Μία από τις πιο βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Να προχωρήσουμε με τη διαδικασία Catch the Eye. Και συνάδελφοι, να σας υπενθυμίσω ότι έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας. Παρακαλώ να σέβεστε τα χρονικά όρια, ιδάλλως θα σας διακόπτω. Ε, ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Μπόκοβιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το διασυνορικό έγκλημα είναι σε εξέλιξη. Οι εγκληματίε δεν γνωρίζουν σύνορα. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κοινή λογική και την αμοιβαία συνεργασία ω απάντηση στο φαινόμενο αυτό. Υπάρχουν πολλέ μορφέ οργανωμένου εγκλήματο. Εκπόρνευση, ε, ε, ναρκωτικά και άλλες τέτοιες ε, μορφές εγκλήματος οι οποίες ε, αναπτύσσονται. Τώρα λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα κλειστά σύνορα της Δανίας γιατί με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να πολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα αλλά θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι κάθε τέτοιο πρόβλημα το οποίο ανακύπτει στα σύνορά μας θα πρέπει να μελετάτε σωστά, θα πρέπει να γνωρίζετε ω βασικό πρόβλημα και να εξετάζετε ποιε είναι οι βαθύτερε αιτίε. Δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και να τα περνάμε όλα αυτά παρατηρητά, γιατί έτσι δεν επιλύονται τα προβλήματα και έτσι δεν κερδίζουμε και την εμπιστοσύνη του κόσμου. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε διαδικασίε σωστέ στην κοινωνία μα, να μην εθελοτυφλούμε όταν ερχόμαστε αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Να έχουμε καλύτερη συνεργασία και να θεωρήσουμε ως βασική αξία την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων. Ε, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, λέει ο κύριος Χαϊζελ. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή η συζήτηση αυτή. Έρχεται σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο χανομένο έγκλημα, έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις υποθέσεις που σημειώθηκαν στη Δανία και στη Σουηδία. Αυτό είναι πολύ θετικό. Είναι πολύ φυσικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Δανίας υιοθέτησε αυτό το προσωρινό μέτρο της επανεισαγωγής και επαναθέσπισης ελέγχων στα σύνορα εντός του χώρου Σέγγεν. Γίνεται για να καταλαγιάσει λίγο η κατάσταση και νομίζω ότι εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε υπεύθυνοι πολίτες και πρέπει να διατηρήσουμε το, τη θετική αφήγηση του Σέγγεν και να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις παρατηρήσεις του Επιτρόπου Σεύκοβιτς. Δηλαδή να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να αξιοποιήσουμε περισσότερο την Europol, να ενισχύσουμε την αστυνομική και άλλη συνεργασία μεταξύ χωρών μελών Αυτά ισχύουν και τα προσυπογράφω 100%. Να κατανοούμε όμως και τη θέση ε, της κυβέρνησης της Δανίας και να μην αξιοποιούμε αυτό το μέτρο για να μπούμε σε πολιτικές αντιπαραθέσεις στήρες. Ας ε, επιδείξουμε λίγη κατανόηση. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε. Η ασφάλεια είναι στόχος για όλους μας λέει η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίγα όμως θα πρέπει να πετύχουμε και άλλους στόχους. Ναι, να συντονιστούμε και να αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες πληροφορίες και τους διαφόρους πόρους. Με την ιστορία του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη έχουμε δει ξανά και ξανά ότι όταν δεν μοιραζόμαστε πληροφορίες και στοιχεία, όταν περιθροποιούμε ε, υπηρεσίες οι οποίες είναι πραγματικά πολύ ικανές, δημιουργούνται πολλά προβλήματα και μας στοιχίζει σε ανθρώπινη ζωή. Πρέπει να έχουμε καλύτερο συντονισμό, ένα ευρωπαϊκό σύστημα συλλογή πληροφοριών, δημιουργία και ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών τεχνολογιών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, εφαρμογών και άλλου είδους τεχνολογικών επιτευγμάτων. Να μην ε, υποχωρήσουμε στις αντιδραστικές δυνάμεις που θέλουν να καταστήχουν ενόχους όλους όσοι φτάνουν στην Ευρώπη. Αυτή η ρητορική του μίσους θα πρέπει να αποφευθεί, να έχουμε ουσιαστική συνεργασία για να ε, αποφύγουμε τις επιμέρους ευθύνε και να εφαρμοστεί σωστά ο νόμος. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό, ο κύριος Βόλας, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην Ιρλανδία το οργανωμένο έγκλημα δεν έχει καμία σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων και οι μετανάστες έχουν διαδραματίσει πολύ θετικό ρόλο στην Ιρλανδική κοινωνία. Από το 2009 και την τραπεζική κρίση αυτό το οποίο έχουμε δει είναι ένα θεσμοθετημένο και ένα νομοποιημένο οργανωμένο έγκλημα στο τραπεζικό μα κλάδο και στο Bad Bank, στην κακή τράπεζα την ΆΜΑ η οποία δημιουργήθηκε για να ασχοληθεί με τα στοιχεία ενεργητικού τα οποία ήταν επισφαλή. Όμω η κυβέρνηση έκανε τα για όλα αυτά. Το οργανωμένο έγκλημα στην Ιρλανδία έχει να κάνει με τα ναρκωτικά. Η καταπολέμηση των ναρκωτικών έχει αποτύχει. Ο πόλεμος εναντίον των ναρκωτικών απότυχε. Όπως επίσης και ε, διάφορες άλλες τέτοιες πολιτικές. Αδυνατό να καταλάβω γιατί η Ευρώπη συνεχίζει να μην εναρμονίζει την προσέγγιση της σε ό,τι έχει να κάνει με, τη, ε, με τα ναρκωτικά. Το μόνο που κάνει είναι να πλουτίζει τους εγκληματίες. Η, η διχαστική αυτή προσέγγιση δεν λειτουργεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κοκαλάρη, η επόμενη μιλήτρια για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τους τελευταίους μήνες συζητήσαμε στο Κοινοβούλιο διάφορα σοβαρά περιστατικά που συνέβησαν σε διάφορα κάτι μέρη μεταξύ άλλων την ποινικοποίηση της, ε, ποινικοποίηση της εκπαιδεύσεως και σεξουαλικά θέματα στην Πολωνία. Είχαμε δολοφονία της δημοσιογράφου στην ε, Μάλτα. Και όταν όμως ε, ήθελα να αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα πυροβολισμών και εκρήξεων στο Μάλμο στη Σουηδία, οι σοσιαλιστέ έθεσαν τροχοπέδι στη συζήτηση. Πώ το ερμηνεύω, Ότι βρίσκονται σε δύσκολη θέση, προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν το πρόβλημα. Εγώ απευθύνω έκκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προ τον Επίτροπο, πραγματικά να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση τη ασφαλείας στην Ευρώπη και στη Σουηδία. Έχασε τον έλεγχο η κυβέρνηση η Σουηδία. Χρειάζεται ενίσχυση η Σουηδική αστυνομία από τη Europol. Χρειάζεται συνεργασία. Δεν θέλω να ξυπνήσω ξανά διαβάζοντα ότι είχαμε σοβαρή έκρηξη βόμβα, όπω σήμερα το πρωί στην πατρίδα μου στη Στοκχόλμη και στην Ούψάλα. Η κατάσταση έχει ε, φτάσει σε πολύ δύσκολα επίπεδα και πρέπει να κινηθούμε. Ευχαριστώ για ένα λεπτό. Η κυρία Γκραπίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βέβαια, πρόκειται περί δικοτά του θέματο που απασχολεί όλου του Ευρωπαίου πολίτε. Παρουσιάζεται ενσυχητική κατάσταση, κύριε Επίτροπε. Έχουμε 5.000 ομάδε εγκληματικέ και ο αριθμό αυξήθηκε κατά 50% εν συγκρίση με το 2013. Και διαρωτώ με ποιε είναι οι λύσει, οι διαθέσιμε που έχουμε μπροστά μα. Διότι και η Europol λέει ότι έχει αυξηθεί η διαφθορά. Έχουμε οικονομική κλιματικότητα, πορνεία, ναρκωτικά, εμπόριο όπλων και απώλεια ανθρώπινων ζώων. Uh, και όχι, όχι μόνο αυτό, έχουμε και πυροβολισμού στου δρόμου. Έχουμε πυροβολισμού σε καταστήματα και σε καφενεία και εστιατόρια και πρέπει να βρούμε λύση. Είπατε ότι σχεδιάζετε να κάνετε μια ανάλυση της καταστάσεως, αλλά θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν συμφωνώ με την κατονομασία της Σουηδίας ή ε, της Δανίας πιο συγκεκριμένα. Μας ενδιαφέρει κάτι άλλο, να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών για να εξαρθρώσουμε αυτά τα δίκτυα που επηρεάζουν έτσι τη ζωή των ανθρώπων. Ευχαριστώ. κύριος Μάντερς είναι επόμενος που έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο για την συνεισφορά του. Μου λείπει, Πρόεδρε, για το Συμβουλίο, βέβαια. Αυτό είναι κρίμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην οικονομική συνεργασία και στην ελευθερία. Και συχνά βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που καταχρούνται τι ε, ελευθερίε αυτή και στρέφονται στο οργανωμένο έγκλημα. Το κόμμα μα υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ωφελήσει τον Ευρωπαίο πολίτη. Αλλά στην παρούσα φάση κάνουμε πάρα πολλά χρήματα και εισοδήματα από το οργανωμένο έγκλημα και δεν μπορούν πλέον να τα καταπολεμήσουν όλα αυτά επαρκώ οι αστυνομικέ και δικαστικέ δυνάμει. Καλό λοιπόν τα θεσμικά όργανα στην επόμενη συνθήκη να φροντίσουν το ποινικό δίκαιο και η καταπολέμηση του οργανωμένου έγκληματος να καταστεί ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Στην παρούσα φάση λοιπόν λόγω της εμ, επικουρικότητας τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να τα επεξέλθουν και υπάρχει υπερβολικά μεγάλη κατάχρηση των ελευθεριών τις οποίες ε, προασπιζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα πρέπει να λάβει ένα τέλος. Να φροντίσουμε να μην χάνουμε τόσα πολλά χρήματα ε, λόγω του οργανωμένου εγκλήματος με διάφορες ευφύης ιδέε και ελπίζω να καταλήξουμε σε μια πολιτική η οποία πραγματικά θα καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα. Ευχαριστώ. Και τελευταία σου λέει πρόεδρος για ένα λεπτό είναι η κυρία Λέιτο. Δεν είναι παρούσα, είναι απούσα. Θα δώσω το λόγο αμέσως στον Αντιπρόεδρο Σεύσοβιτς για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, ευχαριστώ και εσάς και τα αξιότιμα μέλη. Πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση τονίζει το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως Ευρωπαίοι. Αντιμετωπίζουμε το οργανωμένο έγκλημα και τη βία. Και αυτό μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικά είναι αυτά τα θέματα για τους πολίτες μας και πόσο δραματική είναι η κατάσταση. Πολλοί από εσά αναφέρατε συγκεκριμένα πράγματα. Την κατάσταση στο Μάλμο, στη Σουηδία, στη Δανία, και είδαμε σκανδιναβικές χώρες αυτό το φαινόμενο, αλλά θα έλεγα εν γέννη σε όλη την Ευρώπη. Το οργανωμένο έγκλημα αυξάνει τη δράση του, το αθεμπόριο ναρκωτικών έχει αυξηθεί και είδαμε μεγάλο αριθμό εγκληματικών ομάδων που χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τη βία Αναφερθήκατε σε στοιχεία για τη Σουηδία. Συμφωνώ. Είναι εντυπωσιακά. Σας διαβεβαιώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διερευνήσει όλες τις δυνατότητες να δούμε πώς εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλληδικοί φορείς μας όπως η Europol και το Eurojust μπορούν να βοηθήσουν τη Σουηδία. Και άλλες σκανδιναβικές χώρες ή οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που χρειαστεί βοήθεια. Αρκετοί από εσά ρωτήσατε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Στα αρχικά μου σχόλια επανέλαβα κάποια από τα μέτρα που θα θέλαμε να προτείνουμε. Το σημαντικότερο είναι να καλύψουμε τα νομικά κενά να μην υπάρχει διαφοροποιημένη εφαρμογή των νόμων. Οι αστυνομικές μας δυνάμεις θα πρέπει να συνεργάζονται με μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Να κλείσουν έτσι τα σύνορα για τους εγκληματίες και να είναι ανοιχτά τα σύνορα για τους νομοταγείς μας πολίτες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τομπέ, την κυρία Φρίτσα και την κυρία Χάουκεν που ζήτησαν να διερευνήσουμε κάθε δυνατότητα για την αύξηση των δυνατοτήτων που διαθέτει η Europol και να δώσουμε κίνητρα και στα κράτη-μέλη και στις αστυνομικέ δυνάμεις για στενότερη διασυνορική συνεργασία. Είναι ύψιστη προτεραιότητα μας, σας διαβεβαιώ, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δούμε πώς θα αντικατοπτρίζεται αυτό σε ένα πρόγραμμα εργασιών που ελπίζουμε να σας παρουσιάσουμε πριν το τέλος του μήνα. Κάποια από εσά, η κυρία Σαντεμόζα, η κυρία Φαγιών, αναφερθήκατε στην προσωρινή ε, επαναφορά των μεθοριακών ελέγχων από πλευρά Δανία. Να υπογραμμίσω ότι κάτι μέλη έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν τους ελέγχους στα σύνορα αν απειλείται η εσωτερική τους ασφάλεια και γενικά η δημόσια ασφάλεια και η πολιτική τους αναφέρθηκε ο κίνδυνος που δημιουργείται από τη διασυνοριακή εγκληματικότητα που προέρχεται από τη Σουηδία. Να σε ενημερώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει τα διάφορα θέματα. Χρειάζεται αναλογική απάντηση. Ξέρουμε πώς το Σέγγεν είναι σημαντικό για τους πολίτες. Να δούμε αναλογικά τα μέτρα επαναφοράς των συνόρων. Είναι ένα σύμβολο το Σέγγεν ε, τη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και πρέπει να προστατευτεί. Θα πρέπει να αποφύγουμε τα αίτια που οδήγησαν στην προσωρινή επαναφορά των συνοριακών ελέγχων. Κλείνοντας, συμφωνώ με όλους σας που είπατε ότι πράγματι είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και χρειάζεται ευρωπαϊκή λύση. Γι' αυτό είναι κρίσιμη σημασία όλοι μας, όλοι οι φορείς, να συνεργαστούμε σε αυτή την μάχη κατά του εγκλήματος και να υπογραμμίσω το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σας στηρίζει συνεχώς σε αυτή τη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επιτροπέ και έτσι ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το θέμα αυτό. Η επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα των κοινών φορτιστών για τις ε, κινητές ε, συσκευές. Και εδώ πέρα θα δώσω το λόγο λοιπόν και πάλι στον Επίτροπο κ. Σερτσοβίτσα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, το θέμα αυτό θα είναι λίγο πιο ελαφρύ, αν και πολύ σημαντικό επίση για του πολίτε μα. Και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω πραγματικά για την ευκαιρία που μου δίνετε να εξηγήσω τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα αυτό σε ό,τι αφορά του κοινού φορτιστέ. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω καταρχά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την εναρμόνιση των φορτιστών για τα κινητά τηλέφωνα και παρόμοιε συσκευέ και ξεκίνησε μια τέτοια εκστρατεία από το 2009 ήδη. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι χάρη στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κλάδος εθελοντικά ε, ακολούθησε κάποιες συστάσεις και το θέμα αυτό λοιπόν άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη σημασία έκτοτε και μιας και κάνουμε τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, μια βιώσιμη πολιτική για τα προϊόντα είναι βασική προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Πράσινο Deal, το σύμφωνο αυτό, το οποίο υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σας δώσω λοιπόν λίγο μια εικόνα του που βρισκόμαστε, να σας υπενθυμίσω ότι το 2009 λοιπόν είχαμε πάνω από πάνω από 30 φορτιστές, Σήμερα έχουμε τρει βασικέ τέτοιε δυνατότητε. Αυτή η εθελούσια λοιπόν προσέγγιση ήταν πολύ αποτελεσματική. Μειώθηκε ο κατακαιρματισμό της αγορά και έδωσε μία μεγαλύτερη άνεση στον καταναλωτή και πιο πολύ φιλικές λύσει προ το περιβάλλον. Να τονίσουμε επίση ότι τα ηλεκτρονικά απορρίμματα απόβλητα αποτελούν ένα βασικό ακόμα θέμα και πρόβλημα και άρα είναι πολύ σημαντική αυτή η ενιαία διαμόρφωση των φορτιστών. Από το 2014 και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μεγάλες προσπάθειες για να προωθήσει αυτό το εθελούσιο σύστημα. Ακόμα δεν έχει γίνει όμως το τελικό βήμα. Από το 2014 και μετά που σταμάτησε αυτή η εθελούσια ε, συμφωνία έχουν ε, δύο νέες τεχνολογίες USB-C και τις ασύρματες μορφές ε, φόρτιστες και διάφορες άλλες μορφές ταχείας φόρτισης και έτσι στο πλαίσιο των ταχαίων αυτών τεχνολογικών εξελίξεων θεωρούσαμε ότι η εθελούση αυτή η προσέγγιση ήταν η καλύτερη μορφή προώθησης ε, των στόχων μας χωρίς να παρεμποδίζουμε και την καινοτομία. Συζητήσαμε λοιπόν με τον κλάδο την ανάγκη εξέβρεσης λύσεων που θα ε, ικανοποιούν τους εξή στόχους. Άνεση για τον καταναλωτή, ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των φορτιστών και μείωση των ηλεκτρονικών απορριμμάτων το, το Μνημονίο Συμφωνία του 2014, ωστόσο δεν ανταπεξελτέ στι προσδοκίε μα. Ε, ο κλάδο εξακολουθεί να επιτρέπει ιδιαίτερε ε, λύσει ανά μάρκα, αντί να επιβάλλει ένα ενιαίο μοντέλο. Και άρα το πόσο άνετη τελικά είναι η χρήση για τον καταναλωτή και πόσο μειώθηκε ο αντίκτυπο για το περιβάλλον δεν μα ικανοποιεί. Και έτσι δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε φορτιστές κοινούς και για άλλες κινητές συσκευέ. Και μιας και αυξάνεται διαρκώς η χρήση των πόρων σε ό,τι αφορά και τους στόχους μας για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε και άλλες δυνατότητες. Μια μελέτη η οποία θα δημοσιευτεί επίσης τις επόμενες ημέρες θα μας βοηθήσει. Για παράδειγμα, μια λύση, μια τάξη για τις ε, ραδιοσυσκευές ε, και τη σχετική νομοθεσία. Αυτό δεν θα αποτελούσε ενδεχομένω τη βέλτιστη λύση και βασικά θα σημαίνει κατάργηση των συγκεκριμένων ε, λύσεων για φορτιστές συγκεκριμένα από συγκεκριμένε μάρκε, με περιορισμένο όμω όφελο για τον καταναλωτή. Θα πρέπει να πετύχουμε βασική μείωση και των απορριμμάτων και των ε, αερίων του θερμοκηπίου. Για να το πετύχουμε λοιπόν αυτό χρειάζονται επιπρόσθετα μέτρα. Για παράδειγμα, να δοθεί εντολή σε ό,τι αφορά τη χρήση κινητών και τους φορτιστές τους. Κοιτάμε λοιπόν διάφορες λύσεις πολιτικής, ρυθμιστικά και μη ρυθμιστικά μέτρα για να πετύχουμε τους στόχους που αναφέραμε. Η μελέτη επίσης αξιολογεί κατά πόσον είναι δυνατόν να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή και πέρα από τα τηλέφωνα, τα smartphones ε, και να λαμβάνουμε υπόψη και τεχνικά ζητήματα όπως και διαφορετικές ε, ανάγκε. ισχύω. Σε ό,τι αφορά λοιπόν οποιαδήποτε καινούργια λύση θα ήταν ε, καλή αρκεί να αποτελούσε μια κοινή λύση για τη φόρτιση. Θα πρέπει να επίσης να εξασφαλίσουμε ε, την τεχνολογία αυτή και θα πρέπει οι καταναλωτές να έχουν την αίσθηση ότι μπορούν να επιλέξουν. Ιδιαίτερα αν οι, παραγωγοί μπορούν να απολούν τις συσκευέ και τις φορτιστές ε, ξεχωριστά. Για να τα πετύχουμε αυτό θα πρέπει να υπάρξουν ευρείες εκστρατείες ενημέρωσης του καταναλωτή και σε ό,τι αφορά τις ε, τιμές που θα πρέπει να μειωθούν για τι μεμονωμένε συσκευέ. Θα πρέπει επίση να υπάρξει σωστότερη και γρηγορότερη μετάβαση για να υπάρξει ένα μοντέλο βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε δεσμευτεί να κινητοποιήσουμε τον κλάδο για να υπάρχει καθαρή και κυκλική οικονομία. Για να υπάρχει και βιώσιμο σχεδιασμό των προϊόντων με προτεραιότητα στη μείωση τη χρήση των πόρων πριν από την ανακύκλωση. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να κάνει τα επόμενα βήματα για να υπάρξει πραγματικότητα των κοινών φορτιστών και θα σας ε, τηρήσουμε ενήμερους ανάλογα με τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε και τώρα από το, την ομάδα του ΕΛΚ, η κυρία Τούν Φων Χόνστεν. Και να σας επισημάνω, λέει η πρόεδρος, κάτι το οποίο θα το έχετε αντιληφθεί, ότι α, από εδώ και πέρα το ρολόι μετράει ανάποδα. Αν ε, φτάσατε λοιπόν στα κόκκινα ψηφία, θα ξέρετε ότι είναι η ώρα να ολοκληρώσετε την ομιλία σας. Ευχαριστώ. Thank you, President. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και κυρίως αγαπητοί συνάδελφοι από την Επιτροπή ΙΜΚΟ. ΙΜΚΟ. Κύριε Επίτροπε, καλώς ήλθατε. Εδώ και δέκα χρόνια ζητούμε να βρεθεί λύση σε αυτό το απλό πρόβλημα. Πάρα πολλά καλώδια παράγονται, πάρα πολλοί φορτιστές παράγονται και όλα αυτά πετάγονται κάθε χρόνο. Και ο όγκος των απορριμμάτων αυτών είναι απαράδεκτος. Εάν έχει κανείς ταμπλέτα, ψηφιακή κάμερα, έχει ε, κινητό και διάφορε άλλες ψηφιακές συσκευασίε θέλει διαφορετικούς φορτιστές για κάθε μία από αυτές τις συσκευές. Αλλάζουν συνήθως συσκευή κάθε δύο χρόνια οι Ευρωπαίοι και κάθε φορά είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν νέους φορτιστές παρόλο που οι παλιοί λειτουργούν μια χαρά ανα, ανεβαίνει η ζήτηση, έχουμε εξάντληση των φυσικών πόρων, πνιγόμαστε σε έναν ωκεανό ηλεκτρονικών αποβλήτων και απορριμμάτων. 50 εκατομμύρια είναι τα απορρίμματα που δημιουργεί ε, η Ευρώπη, με πάνω από 6 κιλά ανά πρόσωπο, ανά άτομο. Στην Ευρώπη είναι 16 κιλά ανά άτομο, 6 κιλά παγκοσμίω. Μιλώ για τα ηλεκτρονικά απορρίμματα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ο στόχο δεν είναι αρκετός. Περιμένουμε τρεις συγκεκριμένε δράσεις να αναλυφθούν. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να επιδείξει πνεύμα ηγεσία και να σταματήσει να αφήνει τις εταιρείε που είναι γίγαντες στο χώρο της πληροφορικής να μας ε, επιτάσσουν και να μας επιβάλλουν πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας. Θέλουμε να υπάρχει μια πρόταση για ένα πρότυπο για κοινό φορτιστή ασύρματο ή μη τους επόμενου έξι μήνε. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τον κοινό φορτιστή για πολλαπλές συσκευέ. και δεν θα πρέπει ο καταλωτής να αναγκάζεται να πληρώνει για, επιπρόσθετες, για επιπρόσθετους φορτιστές όταν αγοράζει μια οποιαδήποτε καινούργια συσκευή. Και τρίτον, να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότυπα ποιοτικά για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών απορριμμάτων και για την επίτευξη των στόχων σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Ο φορτιστής είναι μια μικρή συσκευή, αλλά το ζήτημα είναι τεράστιο. Και για το περιβάλλον και για τον Ευρωπαίο πολίτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Επόμενος ε, από την ομάδα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών, η κυρία Σουάλντε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ξέρετε, την τελευταία φορά που είχατε έρθει, είχατε δεχθεί τα συγχαρητήριά μου. Αλλά σήμερα δεν μπορώ να το πράξω αυτό. Είναι πολύ δυστυχέ και πολύ κρίμα ε, το γεγονός ότι συνεχίζει να ε, παραμένει αδύνατο να καταλήξουμε σε έναν κοινό και ενιαίο φορτιστή. Ε, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να βρείτε μια λύση το συντομότερο δυνατό. Είναι ίσονο σημασία στο πρόβλημα αυτό. Πώ είναι δυνατόν να έχουμε χρονοτριβήσει τόσο, να έχουν περάσει τόσα χρόνια πριν ε, καταλήξουμε σε μια λύση. Πώ είναι δυνατόν να μιλούμε για κυκλική οικονομία και να μην πράττουμε το αυτονόητο και το τόσο απλό αυτό για τον πολίτη και για το περιβάλλον. Ξέρω ότι προσωπικά εσεί έχετε προσπαθήσει. Όμω ε, δεν μπορούμε να έχουμε μια λύση βολονταριστική. Πρέπει ε, να πιάσετε τον, τον, τάβρο από τα κέρατα εσείς εκεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υιοθετήσετε λύσεις δεσμευτικές, υποχρεωτικής εφαρμογής για τις εταιρείε έτσι ώστε να έχουμε ένα κοινό και νέο φορτιστή για οποιαδήποτε φορητή ή κινητή συσκευή. Η κυρία Σουνανεμάχαρη Μάχαρη απο το Ρινιό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Επίτροπε, αγαπητοί συναδέλφοι, συχνά με ρωτούν τι κάνει για μας η Ευρώπη, τι σημαίνει η Ευρώπη. Και συχνά μιλάμε για μεγάλα και αφηρημένα ε, ζητήματα, η ασφάλεια, η δημιουργία της ενιαίας αγοράς για 550 εκατομμύρια ανθρώπους. Αλλά σε κάποιες περισσοπτώσεις τα πράγματα είναι απλά και πρακτικά, όπως το θέμα των φορτιστών, οι κοινοί φορτιστές για τις συσκευές. Ένας ε, φορτιστής για τα πάντα. Για την ταμπλέτα, για την ε, κάμερα, για το κινητό. Αυτό σημαίνει πιο μικρό κόστος και πιο μικρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Πιο μεγάλη άνεση για τον ε, καταναλωτή. Χρειαζόμαστε λοιπόν λιγότερου φορτιστέ τους, του οποίου θα του πετάξουμε στο επόμενο κινητό που θα πάρουμε. Και το θέμα αυτό είναι επίκαιρο εδώ και μία δεκαετία πλέον. Είναι λοιπόν ε, καιρός να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά και αν και σε πολλέ περιπτώσει οι παραγωγοί διαμαρτύρονται ότι χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται τόσο περιπλοκή. Έχουμε κάνει λοιπόν μεγάλα βήματα πρόοδου. τα τελευταία χρόνια από 30 ε, φορτιστέ έχουμε πάει σε τρει διαφορετικού τύπου φορτιστών. Αυτό είναι θετικό. Αλλά δεν έχουμε πετύχει το ευκταίο ακόμα. Χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω πέρα από την απλή ενθάρρυνση. Η τρέχουσα νομοθεσία λοιπόν εξακολουθεί να ακολουθεί την εθελούσια προσέγγιση, αν και διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει περαιτέρω μετακίνηση. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Θα πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει ένα σχέδιο για έναν καθολικό φορτιστή, ο οποίο θα είναι καλό για του φορτιστέ που θα μειώσει την επιβάρυνση του περιβάλλοντο και που θα αφήσει περιθώρια για καινοτομία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, για του πράσινου. Ο κ. Κόχμα. Για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, Κατά την ακρόαση της Επιτροπής μας τον Νοέμβριο καταγγείλαμε την απουσία σημαντικής προόδου για την επίτευξη του στόχου της ύπαρξης του κοινού φορτιστή για τις διάφορες κινητές συσκευέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά κρύφτηκε πίσω από μελέτες αντικτύπου οι οποίες δεν υπάρχουν και ποτέ θα τις περιμένουμε αλλά θα έπρεπε να έχουν ήδη δημοσιευθεί. Ε, ήδη παρουσιάστηκαν αυτές οι μελέτες τον Οκτώβριο και σε ομάδες εμπειρογνωμόνων. Όμως δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτές. Αναρωτιέμαι γιατί. Εδώ και 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να βασίζεται στην καλή βούληση του κλάδου. Τα λόμπι τρίβουν τα χέρια του, τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Φτάνει πια. Δεν είναι αποδεκτό για τον Ευρωπαίο πολίτη. Ένα μέτρο που μα επιτρέπει να καταπολεμήσουμε την προγραμματισμένη απαξίωση, που μα επιτρέπει να καταπολεμήσουμε την... Ε, και να ενισχύσουμε μάλλον την προστασία του περιβάλλοντο. Δεν γίνεται τέτοια μέτρα να καθυστερούν. Πρέπει να έχετε κατεξουσιοδότηση πράξη ε, επαρκή ή να ξεκινήσετε μια νομοθετική διαδικασία. Δεν μπορείτε να μιλάτε για νέα πράσινη συμφωνία, για New Green Deal και να μην τηρείτε τις υποσχέσεις που έχετε αναλάβει εδώ και 10 χρόνια. Την ύπαρξη δηλαδή ενός κοινού φορτιστή για τις πολλαπλές συσκευέ. Ο κύριος Ζωγόν παρακαλώ, η κυρία Ζωγόν, για ένα λεπτό. Ο κοινό φορτιστή για τα τάμπλετ και τις κινητέ συσκευέ 10 ε, χρόνια συζητείται στους διαδρόμου των Βρυξελών. Οι Ευρωπαίοι πολίτες αδυνατούν να καταλάβουν και να παρακολουθήσουν τη συζήτηση. Γιατί χρονοτριβούμε. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τις υπηρεσίες σας το 2009 και μου είπατε τότε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της διότι ζητά από τον κλάδο την ύπαρξη και σύντομα θα υπάρξει ύπαρξη κοινού φορτιστή. Αυτό μας είχατε πει το 2009. Εγώ πάλι, για να βάλω το κινητό στην πρίζα και βάλω φορτιστή άλλη μάρκα, δεν μπορώ να το φορτίσω. Η Επιτροπή έχει μπει στα πιάτα μας, στα όρια ταχύτητα, στα συνταξιδοτικά μα συστήματα. Αλλά εκεί που θα πραγματικά θα μας χρησιμεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι άχρηστη και ανύπαρκτη και απούσα. Η Apple, δύο εκατομμύρια τουλάχιστον ευρώ ε, ε δαπανά για το λόμπιν. η Nokia ήταν η πρώτη εταιρεία δεν δώσατε άδεια σε αυτήν, αλλά ενισχύσατε τη Microsoft. Έχουμε 16 εκατομμύρια ανέργους. Αν δώσουμε αυτό το φάκελο σε έναν από αυτούς τους ανέργους ή στην Κρέτα, ε, την ακτιβίστρια για το περιβάλλον, πιστεύω πιο καλά και πιο γρήγορα θα τα κάνουν από εσά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δέκα χρόνια για ένα τόσο σημαντικό θέμα για τους πολίτες μας είναι κρίμα. Ένας ενιαίος, ένας μοναδικός φορτιστής θα διευκόλυνε πολύ τη ζωή την καθημερινή των πολιτών μας. Θα ανταποκρινόμασταν και στις προσδοκίες των πολιτών μας. Τώρα ο πελάτης πρέπει να αγοράζει νέο ε, φορτιστή με κάθε νέα συσκευή. Λοιπόν, ένας κανονισμός που θεσπίζεται για να το αλλάξει αυτό θα ήταν κάτι πολύ ικανοποιητικό για τους καταναλωτές. Θα μας επέτρεπε επίσης να περιορίσουμε τα ηλεκτρονικά απόβλητα που σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας είναι δεκάδες χιλιάδες τόνοι το χρόνο. Θα πρέπει να προβούμε σε ενδελεχή ανάλυση του ζητήματος για να εξασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα των διαφόρων συσκευών λαμβάνοντας υπόψη και την φυσική τεχνολογική πρόοδο που είναι ωφέλιμη στους καταναλωτές. Χρειάζονται νέες λύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τις πρόσφατες τάσεις τεχνολογίας και τη σταδιακή εξάλληψη παραδοσιακών φορτιστών υπέρ των ασυρμάτων φορτιστών ούτω ώστε να περιορίσουμε έτσι τα ηλεκτρονικά απόβλητα και να διευκολύνουμε και τη ζωή και των οδηγών, Φερρυπίν. Σας ευχαριστώ. Ξέρω ότι το ένα λεπτό είναι πάρα πολύ σύντομο για να μπορέσετε να πείτε κάτι ουσιαστικό, αλλά παρόλα αυτά να μην τα πληρώνουν οι δερμηνείς που δεν παρακολουθούν. Από την ομάδα της ΓΚΟΕ είναι η επόμενη, η συνάδελφος η κυρία Κονέτσινα για μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλοι στο σπίτι μας έχουμε κάπου πολλούς παλιούς άχρηστους φορτιστές. Κάθε κατασκευαστής είχε ιδιαίτερο φορτιστή. Για τον καταναλωτή αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Ασκείται πίεση άχρηστη ε, πάνω του και είναι κατά το περιβάλλοντος. Με μεγάλη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε τα κινητά τηλέφωνα παράγονται για την ευρωπαϊκή αγορά ότι θα έπρεπε να διαθέτουν έναν γενικό καθολικό φορτιστή. Μέσω κατοξιδότηση πράξης έπρεπε να τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία, αλλά αδράνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν ανησύχησε μην εξοργιστούν οι Apple και είπα, αλλά τελικά δεν εφάρμοσε αυτό που συμφωνήσαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Juncker πολύ συχνά ε, είχε έλλειψη αρχών. Η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φοβηθεί ή θα εφαρμόσει μια οικολογική πολιτική ολιστική, κυρίαρχη, υπέρ των πολιτών. Προσωπικά ελπίζω ότι θα υλοποιήσει αυτό που διεκδικεί το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση από παλιά. Αλλιώς θα πρέπει να βάλουμε τη διακυβέρνηση της Ευρώπης στα χέρια των διαφόρων ομίλων επιχειρήσεων. Δεν χρειάζονται πλέον λόγια, χρειάζονται πράξεις, αποδείξεις. Να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί. Ευχαριστώ, συνάδελφε Μάντρος, για το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Είναι θετικό το γεγονός ότι μιλάμε εδώ για τους κοινούς φορτίστε. Το 2009 έκανα σχετικές ε, προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή και στον τριμερή διάλογο συμφώνησαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή. Δύο, δέκα χρόνια αργότερα ακόμα συζητάμε τους κοινούς φορτιστές. Είναι καλό το γεγονός ότι υπογραμμίζουμε τη μείωση των ε, ψηφιακών απορριμμάτων και αποβλήτων. Αλλά αυτό που δεν τονίζουμε και είναι κρίμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία για τα κινητά τηλέφωνα ε, στην Ευρώπη. Να είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι σε ό,τι αφορά ε, τις επαφέ του από το κινητό τηλέφωνο. Είναι κρίμα που δεν το αναφέρει κανεί. Σήμερα λοιπόν ήρθα από την Ολλανδία στο Στρασβούργο και δεν βλέπω πουθενά να υπάρχουν ε, δημόσια τηλέφωνα. Ε, άντε και δεν έχω μπαταρία και έχω ένα ατύχημα με το αυτοκίνητό μου. Δεν έχω να πάρω κανέναν τηλέφωνο να ειδοποιήσω ότι έχω ένα ατύχημα. Τα τηλέφωνα είναι λοιπόν απαραίτητα για την επιβίωση του ανθρώπου σήμερα πλέον. Το κόμμα μα, το 50 plus 50 Σύνα πιστεύει ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιμείνει στους κοινού φορτιστές για να μπορούν όλοι να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνα όπως γίνεται και τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος ο συνάδελφο Άγγιου Σάλιμπα για ένα λεπτό. Το να υπάρχουν διαφορετικοί φορτιστές ε, για διάφορες συσκευέ είναι βασικής αξίας. Μία, ε, είναι όμως καταρχάς μία, ε, ένας κλάδος ο οποίος επιφέρει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια σε έσοδα. Όχι μόνο οι εταιρείε βγάζουν καινούργια μοντέλα, αλλά κάποια μοντέλα από αυτά έρχονται πλέον στην αρχή με έναν αργό φορτιστή και στη συνέχεια επιβάλλεται πλέον τιμή και κόστος για ένα πιο γρήγορο φορτιστή. Προ... Προφανώς αυτό είναι εξαιρετικά επιζήμιο και για το περιβάλλον. Έχουμε πάνω από 50 δισεκατομμύρια τόνους κάθε χρόνο από τους φορτιστές. Κατά τρίτον, αυτό είναι εξαιρετικά δυσάρεστο για τον καταναλωτή, ο οποίος αναγκάζεται να πληρώσει ένα φορτιστή τον οποίο το χρειάζεται ή αν χρειάζεται κάποιον καινούριο φορτιστή, γιατί κανένα παλιό φορτιστή από αυτού που έχουν δεν ε, φτάνει, δεν κάνει. Φτάνει ω εδώ. Δέκα χρόνια είναι υπερβολικά μεγάλη διάρκεια και θα πρέπει να υπάρξει ένα καθολικό ε, φορτιστή. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα στι ευρωπαϊκέ εταιρείε, τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωή. Αυτή είναι η ευκαιρία μα λοιπόν. Α να δράξουμε. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατεπηγόντω να δράσει. Ευχαριστώ. Η συνάδελφο η κυρία Σαράνσοβα, για ένα λεπτό έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε. Η ομάδα Ρινιού υποστηρίζει την κατεξοδότηση πράξη που θα χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καθορίσει κοινά πρότυπα όσον αφορά ε, τα καλώδια και τους φορτιστές. Η εθελοντική προσέγγιση απέτυχε, δεν έδωσε αποτελέσματα και τα μνημόνια συνεννόησης αξίζουν μόνο εάν εφαρμόζονται πλήρως από όλους τους φορείς αγοράς. Τούτου λεχθέντος. Η καλύτερη λύση δεν είναι κοινό φορτιστής, αλλά το να απαιτούμε να απολούνται ξεχωριστά τα νέα τηλέφωνα και οι φορτιστές και όχι σαν ένα πακέτο. Οι παλιές συσκευές Εάν έχουν παλιό φορτιστή, δεν υποχρεωμένα να πάρουν νέα συσκευή να πάρουν και το φορτιστή το καινούριο. Έτσι μπορούν να πετύχουν καλύτερη τιμή και να περιορίσουμε και τα απόβλητα. Α περικόψουμε τα απόβλητα και α προστατεύσουμε την καινοτομία ταυτόχρονα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Ντεσούτερ, για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, ποιος άλλος γνωρίζει αυτό το πρόβλημα επί σειρά ετών όλοι έχουμε μαζέψει πολλούς φορτιστές για κινητά. Και όχι μόνο γιατί αλλάζουμε μάρκες. Τα καινούργια μοντέλα πολύ συχνά της ίδιας μάρκας έχουν διαφορετικό φορτιστή. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Πάνω από 51.000 τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων ανά έτος, σύμφωνα με της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιβάλλον δεν ωφελείται από αυτό. Όταν λησμονούμε κάπου το φορτιστή μας, μόνο εκείνοι που έχουν το ίδιο κινητό μπορούν να μας βοηθήσουν. Και έτσι και ο καταναλωτή δεν ωφελείται από αυτό. Μόνο βιομηχανία. Κάποιε εταιρείε περισσότερο από άλλε όπω ξέρουμε. Διότι το μεγαλύτερο τμήμα τη βιομηχανία κινείται προ το USB-C. Αλλά κάποιοι όμω αρνούνται να το χρησιμοποιήσουν. Δεν θα πρέπει τα συμφέροντα, τα ιδιωτικά των κερδών να είναι ει βάρο των λαών μα και του πλανήτη. Όταν αυτό που είναι καλό για τον αναλωτή συμπίπτει με αυτό που είναι καλό για το περιβάλλον, πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία. Κατακλείδη Επίτροπε, σας παρακαλώ, δώστε μια βιώσιμη λύση το ταχύτερο δυνατόν. Ήδη έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφε ΣΦΑΠ, για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, καταρχάς να πούμε τα θετικά. Έχουμε ένα φορτιστή ε, ο οποίος είναι αντάπτορας και χωράει όλες αυτές ε, τις ε, φορτιστές που έδειξε ο η κυρία Ντεσούτερ. Και αυτό θεωρώ ότι αποτελεί ένα πολύ μεγαλαφατικό μήνυμα και βήμα για την Ευρώπη. Και έτσι έχουμε πολύ πιο ευνοϊκέ τιμέ στην Ευρώπη. Η τυποποίηση πραγματικά μπορεί να έχει και μεγάλο αντίκτυπο στη μείωση του κόστου για του πολίτε. Αυτό το υπογραμμίζουμε. Θα ήθελα να πω όμω όλου του συναδέλφου οι οποίοι ζητούν αύριο να εισαχθεί ένας καθολικός φορτιστής ότι στην Ευρώπη έχουμε μια οικονομία της αγοράς και θα πρέπει να προσέχουμε όταν εισαγάγουμε τέτοιες λύσεις, να μην παρεμποδίζουν την οικονομία. Όλες αυτές οι εταιρείε που επιμένουν μετά από τόσα χρόνια να αναπτύσσουν δικούς τους ε, φορτιστές και το είπαν αυτό οι συνάδελφοι, να τους υπενθυμίσω ότι από τους 30 διαφορετικούς φορτιστές έχουμε τρεις. Άρα έχουν θετική επίδραση οι συστάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει όλοι να λογούν αν έχουν πραγματικά ξεχωριστό φορτιστή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε συναδελφό κυρία Μπόρζαν. για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πολλοί από εμά έχουμε πολλούς φορτιστές που πολλού, ποτέ δεν χρησιμοποίησαμε. Και έχουμε, ακόμα δεν έχουμε πετάξει παλιούς και σωρεύονται οι νέοι. 51.000 τόνοι ηλεκτρικά απόβλητα έχουμε κάθε χρόνο τα εθελοντικά μέτρα για τυποποίηση των φορτιστών δεν απέδωσαν καρπούς. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα αυξάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα ρυθμό περίπου 5% το χρόνο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα και μοναδικό φορτιστή για όλε τι μικρέ συσκευέ. Εκτιμάται ότι αυτό θα οδηγούσε σε μισό ε, δισεκατομμύριο ευρώ οικονομίε για τον καταναλωτή μέχρι το 2021. Θα πρέπει ένα μικρό βήμα για πιο βιώσιμη κατανάλωση αυτό του ενίου φορτιστή. Μέχρι 78% των καταναλωτών έπρεπε να αντικαταστήσουν το κινητό τους για λόγους που θα μπορούσαν να ήδη, ήδη να έχουν λυθεί στη φάση παραγωγής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε με το παραπάνω χρόνο να βρει ποιοτικέ λύσεις και μοντέλα φορτιστών. Θα πρέπει η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δείξει ότι τα συμφέροντα των πολιτών προηγούνται των συμφερόντων των εταιριών. Συνάδελφε Καρβάλιο, για ένα λεπτό έχετε το λόγο. Συνόρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το θέμα του κοινού φορτιστή έχει τεράστια σημασία, όχι μόνο για τον κατάλληλο διότι είναι υποχρεωμένο συνεχώς να αγοράζει πλειάδα φορτιστών αναλόγως με τη συσκευή που χρησιμοποιεί, αλλά είναι εξέχουσα σημασία σε θέμα και λόγω της οικολογίας. Δημιουργούμε ένα τεράστιο όγκο ηλεκτρονικών απορριμμάτων, ο οποίος είναι μάταιος, ο οποίος είναι άχρηστος. Μιλούμε για 50.000 τόνους φορτιστών που πετιούνται κάθε χρόνο. Επανελειμμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απευθύνει έκκληση να προσεγγίσουμε διαφορετικά το θέμα των φορτιστών, να εθωτήσουμε διαφορετική προσέγγιση. Η Επιτροπή οθέτησε την ε, εθελοντική προσέγγιση που δεν έχει φέρει αποτελέσματα. Πρέπει να επιδείξετε πολιτική βούληση για να επιλύσετε το πρόβλημα και να υιοθετήσετε, να υιοθετήσουμε δεσμευτική υποχρεωτική εφαρμογή νομοθεσία νομοθεσία για την επίτευξη στόχων συγκεκριμένων και ποσοτικοποιημένων αντικειμένων στην ευρωπαϊκή αγορά. Κύριε Γκέπχαρτ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ακούγοντα σα, κύριε Επίτροπε, έγνεφα το κεφάλι μου, γιατί αυτά τα οποία μα λέτε σήμερα, αυτά τα έχω ακούσει πολλές φορές και πριν από 11 χρόνια και πριν από 9 χρόνια και πριν από 10 χρόνια και τελικά τι άλλαξε, τίποτε. Γιατί αγαπητοί συνάδελφοι, λέτε ότι έχουμε μόνο τρει διαφορετικού φορτιστέ. Ε. Κοιτάξτε τα ζετάρια σα. Εγώ βλέπω πιο πολλού. Πολύ πιο πολλού γιατί το θέμα δεν είναι μόνο τα κινητά. Το θέμα είναι και τα τάμπλετ και τις μικρές ε, κάμερες. Και εδώ έχουμε συρτάρια ολόκληρα γεμάτα με φορτιστέ και δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτή την οδό. Θα πρέπει να υπάρχει ένα καθολικό φορτιστή. και είδαμε πραγματικά ότι υπήρξε μια τάση ότι μάλλον αυτή η εθελούσια προσέγγιση από πλευρά των επιχειρήσεων δεν αρκεί. Γιατί μετά από 10-10 χρόνια ακόμα περιμένουμε αυτέ τι υποτιθέμενε λύσει. Όχι λοιπόν, δεν φτάνουν αυτέ οι εθελούσιε λύσει. Χρειάζεται δράση, δράση κύριε Επίτροπε. Και ε, επ' αυτού θέλουμε να επιμείνουμε ω Κοινοβούλιο επιτέλου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Η συνάδελφο κυρία Τότ, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ και 10 χρόνια έχουμε συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξή μας το θέμα του κοινού και ενιαίου φορτιστή, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. Εκφράζω την ικανοποίησή μου διότι κατά την πρώτη σύνοδο Ολομέλεια το 2020, τον Ιανουάριο, έχει μπει το θέμα στην ε, ημερήσια διάταξη. Είναι μια συζήτηση που ωφελεί τον καταναλωτή και ωφελεί και το περιβάλλον. Θα μειωθεί το κόστος για τον καταναλωτή με την ύπαρξη κοινού φορτιστή. Ε, ο οποίος κοινός φορτιστής ε, να λειτουργεί όχι μόνο για τα κινητά τηλέφωνα αλλά και για τους φορητούς υπολογιστές, τις ταμπλέτες, τα διάφορα τάμπλετ ή διάφορες άλλες φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. Θα πρέπει να μπορεί ο καταναλωτής να αποφασίζει εάν θα αγοράσει καινούριο φορτιστή ή όχι. Να το αποφασίζει ελεύθερα και θα πρέπει να αποσυνδεθεί η πώληση της εκάστοτε κινητής φορητής ηλεκτρονικής συσκευής από την πώληση του αντίστοιχου φορτιστή που τη συναδεύει. Αυτό θα ήταν θετικό και για το περιβάλλον, γιατί έτσι θα μειώσουμε σημαντικά το νόγκο των ηλεκτρονικών απορριμμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής για το έλκο ο κύριος Αρίας Ετσεβαρία. 50.000 τόνοι, κυρία Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε, δημιουργούνται ετησίως από ηλεκτρονικούς φορτιστές που είναι πια απορρίμματα. Αυτό πλήττει το περιβάλλον. Πρέπει να έχουμε ενιαίο φορτιστή κοινό. Αυτό θα ωφελήσει τον Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίο όταν ε, ταξιδεύει πρέπει να ε, παίρνει μαζί του διαφορετικού φορτιστέ και αυτό περιορίζει την κοινοτικότητά του δυστυχώ. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για να δοθεί ένα τέλο στην τεράστια ποικιλομορφία φορτιστών. Εδώ και 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνηγορεί και ε, επιχειρηματολογεί υπέρ ενός και φορτιστή και ακόμα δεν τα έχει καταφέρει. Να απλουστεύσουμε παρακαλώ. Ναι, να απλουστεύσουμε και να διευκολύνουμε τη ζωή του Ευρωπαίου πολίτη και των επιχειρήσεων. Η υιοθέτηση ενό κοινού φορτιστή θα διευκολύνει και τη δουλειά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίε θα μπορέσουν να συμμορφωθούν πιο εύκολα με μια όλο και πιο περίπλοκη νομοθεσία. Θα διευκολύνει τη ζωή του Ευρωπαίου πολίτη και θα διευκολύνει και τη διαχείριση των αποβλήτων και απορριμμάτων. Θα μειωθεί ο αριθμό των φορτιστών. Μεγάλες προτεραιότητες τη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η ψηφιοποίηση και η νέα πράσινη συμφωνία. Επομένως, αδράξτε αυτή την ευκαιρία με τον ενίο, με τον κοινό φορτιστή, για να δείξετε στον Ευρωπαίο πολίτη πόσο χρήσιμη είναι η Ευρώπη για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, συνάδελφο Στέφανετ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κοινό φορτιστή θα μπορούσε να αποτελέσει υπόδειγμα. Υπόδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση βελτιώνει τη ζωή του Ευρωπαίου πολίτη. Όλοι έχουμε βρεθεί σε τέτοια κατάσταση όπου δεν βρίσκαμε φορτιστή και δεν μπορούσαμε να φορτίσουμε το κινητό μα τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη φορετή συσκευή χρησιμοποιούμε. Και στο παρελθόν τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα, γιατί ε, κάθε κατασκευαστή έβγαζε δικό του φορτιστή, ο οποίο ήταν διαφορετικό αναλόγω και με το μοντέλο το οποίο ε, ε, κυκλοφορούσε στην αγορά. Έχουν δημιουργηθεί τόνοι, χιλιάδε τόνοι άχρηστων ηλεκτρονικών απορριμμάτων. Οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν δείξει ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να προσαρμοστούν στο πρότυπο θύρα micro USB και να ε, το συμπεριλάβουν στις συσκευές τους. Παραμένουν λίγοι που επιμένουν να μην το κάνουν, παρόλο που δεν υπάρχει ε, εμπόδιο και βασικός και σοβαρός λόγος. Σε κάθε περίπτωση είναι νομοθεσία η οποία δεν περιορίζει την κινητικότητα, την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών, αλλά την ενισχύει, γιατί ενισχύει και την ασφάλεια. Είναι μια νομοθεσία την οποία χρειαζόμαστε απεγνωσμένα. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, η συνάδελφος Ντελκαστήγιο Βέρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας και το είπατε και εσείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ε, είναι όφελος για τον καταναλωτή ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Θα είναι όφελος τεράστιο για το περιβάλλον. Θα έχουμε μεγαλύτερα κέρδη στη νέα ενιαία αγορά. Θα ενισχυθεί ιδιαιτέρως και με ποσοτικοποιημένο και αξιολογήσιμο τρόπο η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μικρών, μεσαίων και μεγάλων. Γιατί λοιπόν δεν συμβαίνει. Καταργήσαμε την περιαγωγή. Υιοθετήσαμε σειρά αποφάσεων για το geo-blocking, για τη φορητότητα του αριθμού. Πολύ σημαντικά πράγματα. Το 2020 για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι η μαγική χρονιά. Πάρα πολλά πράγματα πρέπει να συμβούν το 2020. Υπότιτλοι τα έχετε προγραμματίσει για να δώσουμε μια οριστική απάντηση. Να ε, εκπληρώσουμε τις υποσχέσεις μας, να καταφέρουμε έτσι ώστε ο κοινό φορτιστής να γίνει πραγματικότητα το 2020. Let it happen, κύριε Επίτροπε. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηριζόμαστε πάνω σας. Ευχαριστώ. Και να περάσουμε τώρα στη διαδικασία Cards DI. 7 άτομα έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ήθελα να δώσω τους, το λόγο και στους επτά για να έχουμε μια ζωντανή συζήτηση. Αλλά αυτό θα μπορέσουμε να το κάνουμε μόνο αν δεν ξεπεράσετε αυστηρά το ένα λεπτό. Θα σας ε, κόβω λοιπόν μετά το ένα λεπτό να είσαστε προετοιμασμένοι. Η συνάδελφος η κυρία Τόμς. Σας ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση για τον κοινό αυτό φορτιστή δείχνει ότι μπορούμε να ακούσουμε τους πολίτες μας για συγκεκριμένα θέματα. Όμως έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν σε μια δεκαετία αυτή η συζήτηση, δίκαια λένε οι πολίτες ότι ήμασταν αποτελεσματικοί και ότι είμαστε υπό την επιρροή των πολυεθνικών εταιριών που έχουν άλλα συμφέροντα. Μέσω ενός ε, κοινού φορτιστή, καταρχάς, διευκολύνουμε την καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων. 51.000 τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων έχουμε κάθε χρόνο. Και θα μπορούσαμε να μειώσουμε αυτή την ποσότητα, θα ήταν καλό για το περιβάλλον και θα μπορούσαμε να βρούμε και πιο φθηνές λύσεις για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες. Ελπίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα ολοκληρωθεί στο εγγύς μέλλον Σα είχα προειδοποιήσει ότι θα σα κόψω στο ένα λεπτό. Ο συναδελφό Μαλδονάδο Λόπε. Η κυρία Μαλτονάδο Λόπεθ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πολύ συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, απαγγέλλεται η εξή κατηγορία, ότι δεν δίνουμε λύσεις και, όχι, και αν δώσουμε δίνουμε λύσεις πολύ αργά. Και αληθεύει, ξέρετε αυτό. Από το 2014 χρονοτριβούμε. Ε, υπάρχει οδηγία. Δεν είναι φυσικό και δεν είναι και φυσιολογικό το 2020, ε, όντας η ψηφιακή εθνική και ευρωπαϊκή κυριαρχία μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να υπάρχει αυτό και να μην το έχουμε λύσει ακόμα. Και πολλοί συνάδελφοι το είπαν έχουμε τεράστιο ρυθμό φορτιστών που δεν χρησιμοποιούμε πια. Είναι πολύ σημαντικό και οι νέοι σας το ε, έδειξαν με τα παραδείγματά τους για τους λόγους της κλιματικής αλλαγής. Δεν γίνεται κάθε φορά να αγοράζουμε ηλεκτρονική συσκευή, ηλεκτρονικό ρολόι, ηλεκτρονική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ και κάθε φορά να αγοράζουμε νέο φορτιστή. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Διακόπτη πρόεδρος. Ο συνάδελφος κ. Μπότος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, εδώ και πολλά χρόνια κάναμε ένα βήμα προόδου για την τυποποίηση των φορτιστών. Θα ήταν κάτι επωφελές για τους ε, καταναλωτές. Έναν κοινό τώρα φορτιστή αν είχαμε για όλες τις κινητές ηλεκτρονικές συσκευές θα ήταν καλό για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Πρέπει να εξασφαλίσουμε όμως ότι τα επόμενα βήματα θα γίνουν ταχύτερο δυνατόν ούτως ώστε οι Ευρωπαίοι να μπορούν να απολαύσουν ταχύτερο δυνατόν τα ωφέλη των κανονισμών. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε τους στόχους που είχαν τεθεί μέσω της Πράσινης Συμφωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επίσης να επιβάλλουμε τεχνολογίες παραγωγής που θα εστιάζονται στην προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει να υπάρχουν προγράμματα ανακύκλωση, ώστε το ίχνος άνθρακα του τελικού προϊόντος να είναι το ελάχιστο δυνατόν. Αυτά τα πρότυπα θα πρέπει να τα πληρούν οι φορτιστές που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προϊόντα που εισάγονται. Ευχαριστώ. επόμενο. συνάδελφε Φερέρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι φορτιστές των κινητών τηλεφώνων. Υπάρχουν ε, πολλά προϊόντα που είναι ασύμβατα με φορτιστή ε, άλλης εταιρείας. Οπότε έχουμε τώρα αυτά τα απειρχιωμένα προϊόντα που ε, παραμένουν άχρηστα. Υπάρχει ασυμβατότητα που κοστίζει ε, και η προγραμματισμένη ε, χρήστευση αυτών των φορτιστών είναι κάτι που είναι σβάρος των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Η στρατηγική για την προστασία του περιβάλλοντος και του, της ανθρώπινης επιρροής στο περιβάλλον είναι η λύση που θα βρούμε για αυτό το πρόβλημα πώς μπορούν να αποσυναρμολογούνται οι συσκευές, παραδείγματο χάρη, ε, ούτως ώστε να μπορούν να αντικαθίστανται διάφορα ανταλλακτικά πιο εύκολα και να επικαιροποιείται και το λογισμικό και τα ανταλλακτικά και συσκευές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εξετάσει τα κατάλληλα μέτρα γι' αυτό. Λεϊτάου Μάρκε. η κυρία Λεϊτάου Μάρκε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Νομίζω ότι ακούσατε ότι υπάρχει συνένεση εδώ στο Κοινοβούλιο για τα μέτρα τα οποία θέλουμε να ληφθούν. Ανησυχούμε, ανησυχούμε για τις καθυστερήσεις που διαπιστώνουμε, γιατί είναι σημαντικά τα μέτρα αυτά για τους ε, καταναλωτές, όπως ήταν και στο παρελθόν η περιαγωγή. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε λοιπόν τέτοια μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή κόσμου και μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η ψηφιακή μετάβαση, αλλά και το θέμα της μετάβασης σε θέματα περιβαλλοντικά. Είπαμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε περαιτέρω για την πρωτοβουλία αυτή της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Θα χρειαστεί να υπάρξουν νομοθετικά μέτρα και πρότυπα προδιαγραφέ ή και τα δύο για να υπάρξει η απαραίτητη ευελιξία για την κοινοτομία. Δεν μπορούν να συνεχιστούν όλα αυτά. Δεν μπορούν να τα πετύχουμε όλα αυτά, κύριε Επίτροπε, αν σήμερα κάτσουμε να περιμένουμε άλλα 10 χρόνια ε, ενώ οι ενιαίοι αυτοί οι φροντιστέ ε, μπλοκάρονται από τι επιχειρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σόιντροβα. Σας ευχαριστώ πολύ και συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι και θα στραφώ προς τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί όλοι τονίζουμε ότι δεν θέλουμε να περιμένουμε 10 χρόνια και στα 10 χρόνια να ξαναρχίσουμε να μιλάμε για το θέμα των καθολικών φορτιστών, των ενιαίων φορτιστών. Θεωρώ ότι αυτό που αποτέλεσε πρόβλημα το 2014 δεν εξακολουθεί να αποτελεί σήμερα μόνο πρόβλημα των καταναλωτών. Το θέμα είναι και ο όγκος πλέον των απορριμμάτων που είναι περιττός. Αν θέλουμε λοιπόν να πάρουμε στα σοβαρά αυτό το πράσινο σύμφωνο, την πράσινη συμφωνία, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι και η κάθε καινούργια καινοτομία θα πρέπει να είναι καινοτομία πράσινη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ε, ενιαίος φορτιστής. Ε, αν θεωρούμε ε, ότι έτσι μπλοκάρουμε την καινοτομία, ουσιαστικά αυτή είναι λάθος σκέψη. Δεν βλέπω εδώ την επόμενη συνάδελφο, λέει η Πρόεδρος. Α, εδώ είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Επίτροπα. Θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να υπάρξει πραγματικά ένας ενιαίος φορτιστής στην Ευρώπη και όχι μόνο για λόγους αλλά γιατί ένας καθολικός φορτιστής θα επέτρεπε να γίνει σημαντική εξοικονόμηση κόστους και του καταναλωτή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να υποκύπτει στα επιχειρήματα των επιχειρήσεων για την ε, καταπίεση της καινοτομίας δήθεν. Όχι, οι τιμές που πληρώνουμε για τις νέες ε, συσκευές για τον νέο εξοπλισμό αποτελούν από μόνο τους λόγο να πούμε στις εταιρείε αυτές ότι φτάνει πια και θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ και τώρα να ακούσουμε τον Επίτροπο τον κ. Ζεύτσοβίτση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ για τις τοποθετήσεις σας. Θα ήθελα να πω ότι τις παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή και το μήνυμα πραγματικά ελήφθη. Πολύ σπάνιο είναι όλοι οι βουλευτές να εκφράζονται ομόφωνα για ένα θέμα που αποσχολεί την ολομέλειά σας και αυτό συνέβη σήμερα το απόγευμα. Το δείξατε αυτό. Συμφωνώ μαζί σας ότι παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταβάλει προσπάθειες, πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη εναρμόνιση και να ασκήσουμε πίεση για πιο αηφόρα προϊόντα. Και σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα της προσπάθειάς μας δεν ήταν τα αναμενόμενα και αυτό το δέχομαι. Θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η έλλειψη πρόοδου ε, έλαβε χώρα όχι γιατί φοβόμασταν ε, μια κάποια εταιρεία μια οποιαδήποτε εταιρεία. Αντιθέτω, ε, δεν σημειώσαμε πρόοδο γιατί προσπαθούσαμε να βρούμε ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο να προχωρήσουμε προς τα, μπροστά και να σημειώσουμε πραγματικά πρόοδο. Η μείωση των ηλεκτρονικών απορριμμάτων ενισχύει ε, η ενίσχυση της ασφάλειας, η βελτίωση της διαλειτουργικότητας. Αυτές θα είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που θα διέπουν το έργο μας. Και συντάσσομαι μαζί, μας, μαζί σας και απευθύνω και εγώ έκκληση στον κλάδο να καταβάλει κάθε να την προσπάθεια να επιτεχύνει την τεχνολογία, να έχει νέα προϊόντα πιο αποτελεσματικά με καλύτερες επιδόσεις προς όφελος του καταναλωτή, προς όφελος της οικονομίας αλλά και του περιβάλλοντος. Πιστεύω ότι πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι η εθελοντική προσέγγιση σε αυτή την περίπτωση δεν στάθηκε στο ύψος των προσδοκιών των βουλευτών, στο ύψος των προσδοκιών των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά ούτε και στο ύψος των δικών μας προσδοκιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ με όσους το έθεσαν ξεκάθαρα η κυρία Τουνχώσερ, η κυρία Σάλτεμόζε, αλλά και όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πήραν το λόγο το διαπίστωσαν και συμφωνώ μαζί σας. Θέλω λοιπόν να επαναλάβω αυτό το μήνυμα προς το κλάδο. Δεν είναι αργά να ε, καταλήξουν σε συγκεκριμένες προτάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, μετά από τόσα πολλά χρόνια, πρέπει να εξετάσουμε το εδεχόμενο να υιοθετήσουμε την νομοπαρασκευαστική και νομοθετική διαδικασία. Έχουμε ως πρόθεση να αναλύσουμε και άλλες επιλογές, π.χ. τακτή νομοθετική διαδικασία, συνηθισμένη με, στόχος να, με στόχο να υπάρχει ε, σημαντική σχέση κόστους-οφέλους προς το συμφέρον του Ευρωπαίου καταναλωτή. Όσοι τόνισαν την τεράστια σημασία της ψηφιακής ευρωπαϊκής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της Ευρώπης με βρίσκουν σύμφωνο. Σήμερα βλέπουμε πόσο μεγάλη σημασία αποκτά όλο και μεγαλύτερη θα έλεγα το ζήτημα αυτό. Και έρχομαι εδώ να προσθέσω ένα σημαντικό στοιχείο και ένα δίδαγμα που έχουμε αντλήσει από όλη αυτή την προσέγγιση. Ένα δίδαγμα το οποίο θα διέπει και το έργο ε, που θα πράξουμε για το European Battery Alliance. Ας ε, καταλήξουμε στο εξής συμπέρασμα όσο γρηγορότερα έχουμε υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα, όχι μόνο για τους φορτιστές αλλά και για τις μπαταρίες, τόσο το καλύτερο για εμάς και για το μέλλον μας. Έτσι θα εξυγχρονίσουμε το κλάδο, έτσι θα ε, υπογραμμίσουμε τη δέσμευσή μας για την αηφορία των ευρωπαϊκών προϊόντων και αυτό ακριβώς θα πράξουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για το πολύ σαφές μήνυμα που στείλατε, το οποίο ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα αναλάβει ταχεία και ενεργητική δράση και ελπίζω ότι θα μπορώ να βασιστώ στη στήριξή σας όταν επιστρέψουμε με συγκεκριμένες προτάσεις για να τι καταθέσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Η πρόεδρο, και εγώ σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ του συναδέλφου Συγγνώμη που αγενός στέρισα το λόγο από κάποιους, αλλά δεν έχουμε αρκετό χρόνο δυστυχώς. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτηση αυτή και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σε μελλοντική συνεδρίαση. Και έχουμε την επόμενη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη στέχαση Housing First. Ε, στέκει αυτό, λέει η Πρόεδρος. Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την διαφορά, το μισθολογικό κενό που υπάρχει μεταξύ άνδρων και γυναικών. να περιμένουμε την Επίτροπο, στην οποία θα δώσουμε παραφαδό λόγο. Welcome. Herzlich Καλώς ορίσατε λοιπόν, κυρία Επίτροπε Ντάλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχετε το λόγο. Αξιότιμοι βουλευτέ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για που με συμπεριλάβατε που συμπεριλάβατε το θέμα της, ε, του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των ε, φίλων στη σημερινή ατζέντα. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό προφανώς για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό αποτυπώνεται και στα ψηφίσματά σας που κατζητούν ε, νομική δράση για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού και της διακριτικής μεταχείρισης. Βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο, έχουμε την ίδια αντίληψη για τα θέματα αυτά. Αυτές οι διακριτικές ε, μεταχειρήσεις υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτή η ισότητα υπάρχει θεωρητικά από το 57, αλλά οι γυναίκες εξακολουθούν να λαμβάνουν μισθούς χαμηλότερους κατά 16% κατά μέσο όρο σε σχέση με τους άντρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε δράση. Η πρόεδρος Φοντερ Λάιεν μου ανέθεσε το καθήκον να αναπτύξω μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα την μισθολογική για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Θα δώσουμε λοιπόν στην ποιότητα της εργασίας ε, ύψιστη σημασία για να υπάρχει διαφάνεια σε ό,τι αφορά τι αποδοχέ των ατόμων. Αυτό θα χρειαστεί λοιπόν μια νέα στρατηγική από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία θα παρουσιάσουμε την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Στόχο μα είναι να έχουμε μια ισχυρή και φιλόδοξη και ευρεία προσέγγιση με συγκεκριμένα μέτρα για να κλείσει επιτέλου αυτό το χάσμα. Η ίση αμοιβή θα είναι βασική αρχή τη νέα στρατηγική και θα επιμείνει σε θέματα διαφάνειας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπήρξαν ε, μη δεσμευτικέ συστάσεις εδώ και πέντε χρόνια πλέον, οι οποίε έδωσαν στα κρατημέλη μια εργαλειοθήκη με μέτρα για να εφαρμοστεί η αρχή της ίση αμοιβή. Κάποια κράτη εισήγαγαν τα μέτρα αυτά, πολλά εξ αυτών όμω δεν το έπραξαν. Και υπάρχει έλλειψη διαφάνεια. και έτσι πολλές γυναίκες δεν γνωρίζουν ακόμα καν ότι πληρώνονται λιγότερο, ότι αμείβονται χαμηλότερα. Η εργασία λοιπόν των γυναικών συστηματικά και διαστατικά ανταμείβεται πιο χαμηλά σε σχέση με την εργασία που κάνουν οι άνδρες, ακόμα και αν πρόκειται για εργασία ίσης ε, αξίας. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό το σκέλος της διαφάνειας. Θα εξετάσουμε λοιπόν μια ευρία γκάμα εναλλακτικών λύσεων σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για την διαφάνεια σε ό,τι αφορά την αμοιβή. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την υποχρέωση οι εταιρείε να αναφέρουν τα επίπεδα αμοιβή των επαλληλών τους στους σχετικούς ελέγχους. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο να εισαχθούν τέτοια δεσμευτικά μέτρα. Θέλουμε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των υπαλλήλων ε, να έχουν πιο, πολλά, πιο πληροφορίες για τα επίπεδα τα μισθολογικά. Αλλά κάποια από τα μέτρα αυτά ενδεχομένω να σημαίνουν και μισθολογικό και γραφειοκρατικό άχθο για τι εταιρείε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρξει διαβούλευση και με τι εταιρείε και με του ε, υπαλλήλου και του εργαζόμενου και με τι εθνικέ αρχέ για να βρεθεί μια σωστή ισορροπία για το μέτρο αυτό. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια για, τα μισθολογικά, για τις μισθολογικές αποδοχές είναι ένα βήμα και μόνο για να αντιμετωπίσουμε το μισθολογικό χάσμα η κάλυψη του χάσματος αυτός σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει και μία συνεκτική προσέγγιση και να καταπολεμήσουμε όλες τις βαθύτερες αιτίε σε ό,τι αφορά τη ε, χρήση απασχόλησης, ε, μερικής απασχόλησης των γυναικών, ε, της διακοπής, της καριέρας σε σχέση με τους άντρες, τα στερεότυπα που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τα φύλλα, η διακριτική μεταχείριση και ούτω καθεξής. Επίσης, οι γυναίκες είναι υπερβολικά δραστήριες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και συχνά έχουν προσωρινέ συμβάσεις και μεταβαλλόμενα ωράρια. Αυτά προφανώς και αυξάνουν το μισθολογικό χάσμα. Από την άποψη αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τα κρατημέλη για να εξασφαλίσει ότι δεσμευτικέ νομοθετικέ δράσει θα ληφθούν και για να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη προκειμένου να επωφεληθούν από τις νομικές διατάξεις. Αυτό συμπεριλαμβάνει και πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, την οδηγία για την μερική απασχόληση, την οδηγία για διαφανείς όρους εργασίας και προβλέψιμους όρους εργασίας και φυσικά σε ό,τι αφορά την οδηγία για την εξισορρόπηση επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. Σκοπεύω να συνεργαστώ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία αυτή και προσβλέπω να ακούσω και τις δικές σας απόψεις από αυτού σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επιτροπέ. Από την ομάδα του ΕΛΚ η συνάδελφο κυρία τα έχει καταρχά ε, το λόγο. Να σα υπενθυμίσω και πάλι ότι ο χρόνο μετράει αντίστροφα στο ρολόι μα σήμερα. Και αυτό που είναι ίδιο, ωστόσο, είναι ότι μόλι περάσετε στα κόκκινα ψηφία θα πρέπει να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Καλωσορίζω αυτά που είπατε απόψε. Χαίρομαι που είμαστε όλοι συντονισμένοι. Έτσι πρέπει για να δραστηριοποιηθούμε όσον αφορά το θέμα. Αν είμαστε σοβαροί για την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν είμαστε σοβαροί για τους στόχους χιλιετίας βιώσιμης ανάπτυξης, και για τον κοινωνικό πυλώνα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, τότε είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων. Η ισότητα έχει σημασία και είναι σοβαρότατη αυτή η ανισότητα που έχει διαρκέσει επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η οικονομική ισότητα είναι κρισίμου σημασία, διότι χωρί την ισότητα στην αμοιβή για να ζήσουν οι άνθρωποι, η κοινωνική ισότητα δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. 16% είναι η διαφορά, αυτό το μισθολογικό χάσμα σε κάποια μέρη και έχουμε και το θέμα του χάσματος μεταξύ των συντάξεων, που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Η παρούσα διαφορά μεταξύ των φύλων συντάξη είναι διπλάσια διαφορά, είναι 37,5% η διαφορά. Σκεφτείτε τι συνέπειες έχει αυτό για τις γυναίκες, για τα παιδιά, για τις οικογένειές τους όσο μεγαλών και γερνάνε. Δεν έχουν πρόσβαση στα ίδια χρήματα για να μπορέσουν να ζήσουν τη ζωή τους και οι συνέπειες και του μισθολογικού χάσματος και του συνταξιοδοτικού χάσματος είναι πολύ σοβαρές, κοστίζουν στην κοινωνία μας, ε, κοστίζουν διότι διονύζουν τη φτώχεια των παιδιών, διονύζουν την έλλειψη δεξιοτήτων και βεβαίως υπάρχει τεράστιο κόστος που δημιουργείται για τις οικονομίες όλων των χωρών μας, διότι υποχρησιμοποιούν τις δεξιότητες των γυναικών και υπάρχει σοβαρό φραγμό όσον αφορά εδώ την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Όλοι τα γνωρίζουμε αυτά. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε. Αυτό που βλέπουμε ήδη σε αρκετέ χώρε, βλέπουμε να δραστηριοποιούνται ευπρόσδεκτα αυτά που είπατε για τα διάφορα ζητήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν εάν πάρουμε σοβαρά το θέμα. Η διαφάνεια των αμοιβών είναι κρισίμου σημασία. Είδαμε ήδη τι αντικτυπώ έχει. Η μεγαλύτερη διαφάνεια, παραδείγματο χάρη, όταν εξετάζεται ε, στις διάφορες ε, ασχολίες. Χρειάζονται εφαρμοστικά μέτρα ε, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ. Για σοσιαλιστές, συνάδελφε Ρέγκνερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αξιότιμη κυρία Επιτροπέ. Είναι λυπηρή αυτή η ημέρα, γιατί αυτή η μεγάλη διαφορά του μισθολογικού χάσματος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταδεικνύει ότι αυτή την ημέρα τη ε, μισθολογική ισότητα δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Και αυτό αφορά τι ε, γυναίκε και του άντρε. Και το γεγονό ότι υπάρχει αυτή η αρχή για την ίση αμοιβή, για ίση εργασία. Αυτό κατοχυρώνεται στι ευρωπαϊκέ συνθήκε. Παρά το γεγονό ότι έχουμε την οδηγία για την ίσια μεταχείριση και στο κεφάλαιο 4, στο άρθρο 4, απαγορεύεται η διακριτική μεταχείριση. Εξακολουθούμε να έχουμε 16% χαμηλότερη μισθολογική αποδοχές για τις γυναίκες σήμερα. Και οι γυναίκες κατά 40% έχουν χαμηλότερες συντάξεις σε σχέση με τους ε, άνδρες. Και οι μητέρες με νεαρά παιδιά κατά από 6 χρονών είναι Αυτέ που έχουν την μεγαλύτερη διακριτική μεταχείριση. Οι γυναίκε λοιπόν ουσιαστικά έχουν χαμηλότερε αποδοχέ, ακριβώ επειδή είναι γυναίκε. και αυτό βασίζεται σε ε, στερεότυπα για το ρόλο των γυναικών οι οποίε εξακολουθούν να αναλαμβάνουν το πιο πολλά καθήκοντα στι οικιακέ εργασίε και για τη φροντίδα των παιδιών. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουν οι σημερινέ νοοτροπίε και ισορροπίες δυνάμεων αν θέλουμε να υπάρξει πραγματική πρόοδο. και γι' αυτό λοιπόν στρέφουμε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειαζόμαστε πιο πολλά α, σκληρά μέτρα για την ε, μισθολογική ισότητα, για την διαφάνεια, κυρώσεις όταν υπάρχει διακριτική μεταχείριση και ολική αποζημίωση των ε, πληγέντων. Αυτό αναμένουμε για να υπάρχει πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την Renew, η κυρία Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ αγωνίζομαι για ισότητα, για την εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος. Έτσι καταπολεμούμε τη γυναικεία φτώχεια και το γυναικείο κοινωνικό αποκλεισμό. Η απόκληση στις αμοιβέ είναι απαράδεκτη και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο κοινωνικό, διότι καταστρατηγείται η αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης που κατοχυρώνεται στις ευρωπαϊκές, ε, στα ευρωπαϊκά συνταγματικά κείμενα. Επίσης, θεωρούμε ότι αν μειωθεί κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, θα υπάρξει δημιουργία πλούτου 40 δις ετησίως στην Ευρωπαϊκή ε, Ήπειρο. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Κατόφλι για τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα και πρέπει να το εφαρμόσουμε. Πρέπει να ενημερώσουμε και να επικαιροποιήσουμε την ευρωπαϊκή δράση γύρω από τρει άξονε. Πρώτον, διαφάνεια στοιχείων και πληροφοριών για τι αμοιβέ να βελτιωθεί. Δεύτερον, υποχρέωση διορθωτικών μέτρων και ε, εκτίμησης αποτελεσμάτων. Τρίτον, συνοδευτικά μέτρα πλαισίωσης για καλύτερη οργάνωση. Έχουμε μέτρα ελέγχου ε, για τη μισθολογική κλίμακα, για τις απολαβές, για το μισθολογικό χάσμα, για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το περίγραμμα των διακρίσεων που σημειώνονται και να μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε και να μετρήσουμε την πρόοδο που σημειώνεται. Χαίρομαι, διότι βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται προς την κατεύθυνση της διαφάνειας, διότι πρόκειται για την οδηγία του 2014 για τα στοιχεία τα έξω χρηματοπιστωτικά. Ε, ο κοινωνικός και εργασιακός διάλογος είναι εξαιρετικά σημαντικός μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για να έχουμε διορθωτικά μέτρα υποχρεωτικά χαρακτήρα και δεσμευτικού χαρακτήρα, αλλά και γενικότερη βελτίωση της διοργάνωσης της αγοράς εργασίας για να κατοπολεμήσουμε τα στερεότυπα τον επαγγελ... στον επαγγελματικό προσανατολισμό μεταξύ άλλων. Περιμένουμε με ανυπομονησία τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των ανθρώπων. Για ίδια δουλειά, ίδιος μισθός παραμένει το σλόγγαν που μας δονεί. Ευχαριστώ. Και να καλωσορίσουμε και τους έξι άντρες που θα πάρουν το λόγο στην συζήτηση αυτή. Καταρχάς, ο κύριος Ούρτασον έχει το λόγο για μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι φυσιολογικό να είμαστε τόσο λίγοι σε αυτή την αίθουσα εδώ όταν συζητείτε ένα τέτοιο θέμα και πρέπει να το πω. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για αυτά που μας παρουσιάζετε. Μας έχετε γεμίσει ελπίδες ότι θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το μισθολογικό χάσμα, τις μισθολογικές αποκλήσεις που πλήττουν πάρα πολλές γυναίκες. Μιλήσατε εσείς για τα νούμερα, αλλά έχουμε απόκληση μετά ε, και στην ίσπραξη ε, των συντάξεων, το οποίο είναι απότοκος του φαινομένου του μισθολογικού χάσματος ε, εξ αρχής. Δύο είναι τα σημαντικά κατεμέ να έχουμε μια στρατηγική συγκεκριμένη, ένα σχεδίο δράσης για την καταπολέμηση των μισθολογικών αποκλήσεων. Αυτή η στρατηγική δεν δούλεψε. Πρέπει να έχουμε σαφείς δείκτες, ποσοτικοποιημένα μετρήσιμα στοιχεία για να εκτιμήσουμε το φαινόμενο. Και έχουμε και τη νέα οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια που έχετε παρουσιάσει στο περιεχόμενο αυτής θετικό βρήκα την ύπαρξη υποχρέωσης ελέγχου, δηλαδή οι εργαζόμενες να μπορούν να γνωρίζουν τις διάφορες κλίμακες, αναφύλλο και ούτω καθεξής, πρέπει να υπάρξει καθεστώς κυρώσεων και προστατευτικών μέτρων για τα θύματα που έχουν πέσει, ε, για όσους έχουν πέσει θύματα αυτές, αυτών των μισθολογικών αποκλήσεων. Τελικά στην Ιρλανδία έχει, εξαλειφθεί αυτό το χάσμα και πρέπει να δούμε τι έχουν κάνει εκεί και θα πρέπει να συνεργαστούμε ε, και να ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο. Δεν θέλω... Δεν θέλω αυτό το κείμενο να αποδυναμωθεί στο Συμβούλιο. Έχουμε εξαιρετική Υπουργό Αρμόδια στην Ισπανία και είμαι σίγουρος ότι θα σταθεί στο πλάι σας. Ευχαριστώ πολύ. Κρά, για ένα λεπτό έχει το Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίε και κύριοι, το μυστολογικό χάσμα είναι ένας από τους ε, ε, μοντέρνους μύθους και όσο πιο πολύ το κοιτάμε τόσο πιο ε, λίγο ουσία φαίνεται, λίγη ουσία φαίνεται να υπάρχει. Υπάρχει λοιπόν ένα 7% μισθολογικό χάσμα και στους νέους είναι ακόμα και αντίστροφο. Και βλέπουμε λοιπόν στη Βρετανική αριστερά ότι υπάρχει το εξής. Θα πρέπει όλα αυτά να αποτυπώνονται η μητρότητα και όλα αυτά να αποτυπώνονται στις ε, συντάξεις. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Πολωνίας που λαμβάνουν υπόψη τις μητέρες προκειμένου να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα. Αν ναι, θέλουμε λοιπόν να δώσουμε στις γυναίκες την αξία τους, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια νέα ιδεολογική τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρξει προστασία των γυναικών και της μητρότητας και όχι να γίνονται τέτοιες επίπλαστες συζητήσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Βυσνίσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αληθεύει ότι μιλάμε συνέχεια για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών και φτάνει το 16%. Εγώ είμαι αρκετά τυχερή που είμαι από την Πολωνία και από εκεί το χάσμα είναι 7% και μειώνεται σχετικά με την ανεργία των γυναικών μειώθηκε αυτή από 18% σε 5%. Αλλά πολλά απομένουν να γίνουν. Υπάρχουν πολλά αίτια για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φίλων, αλλά πιστεύω το πιο σημαντικό αίτιο είναι ότι οι γυναίκες είναι υπεύθυνε για τη φροντίδα των οικογενειών. Ασχολούνται γιατί έχουν να προσέξουν τα παιδιά τους και τους ηλικιωμένους γονείς. Πολύ συχνά οι γυναίκες εργάζονται σε μερική απασχόληση σε τομείς που αμείβονται χειρότερα. Θα πρέπει να εξετάσουμε ενδελεχέστερα τι μπορούμε να κάνουμε με τις γυναίκες που είναι μητέρες, που φροντίζουν και τους ηλικιωμένους ασθενείς γονείς τους. Πώς μπορούμε να τις αποζημιώσουμε για το πολύτιμο έργο τους. Να προσθέσω επίσης ότι είμαστε μάρτυρες τη φτώχεια που πλήττει περισσότερο τι γυναίκε. Παίρνουν συντάξει πολύ πιο χαμηλέ από του άντρε οι γυναίκε. Συνάδελφε, περίεργα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι μια πραγματικότητα και όταν εργάζεται κανείς και επιδεινώνεται με τις συντάξεις. Μπορεί να τεθεί τέρμα αυτό με στοχευμένα μέτρα για να καταπολεμήσουμε τα αίτια αυτού του χάσματος η εγγύηση της ισότητας μισθολογικής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η αύξηση της αξίας των συλλογικών συμφωνιών και η ρύθμιση των ορών εργασίας. Πέραν από αυτά πρέπει να προστατεύεται η μητρότητα και να έχουμε δίκτυα προστασίας των ηλικιωμένων και των παιδιών και μέτρα που δίνουν στις δημόσιες υπηρεσίες επαρκείς πόρους ε, από πλευράς οικονομικής ε, προσωπικού και μέσων για να καταπολεμήσουν αυτή τη διάκριση και να συμμορφωθούμε την νομοθεσία. Θα πρέπει να πασπιστούμε και την δημόσια ε, κοινωνική ασφάλιση που είναι ένα κοινό αγαθό και που αποτελεί μια εγγύηση ε, για τις συντάξεις. Ευχαριστώ Ραντισόφσκι. δεν είναι εδώ. Μήπως έχει κάτσει κάπου αλλού. Αν δεν είναι στην αίθουσα να πάμε παρακάτω και ήμουν κάπως πιο γενναιόδορη σε ό,τι αφορά τους ομιλητέ ομιλητές από πλευρά των πολιτικών ομάδων, αλλά θα είμαι πιο αυστηρή τώρα. Και τώρα έχουμε την συνάδελφο, την κυρία Εστέρα Σφραγκούτ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, η αρχή των μισθολογικών απολαβών, των ίσων μισθολογικών απολαβών, κατοχυρώνεται στα ευρωπαϊκά κείμενα και αποτελεί μέρος των στόχων της ε, κοινωνικής μας ανάπτυξης, αποτελεί μέρος του κοινωνικού και εργασιακού πυλώνα που έχουμε εγκρίνει. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το θεώρησε βασική προτεραιότητα στη νέα στρατηγική για την ισότητα και αντίστοιχη η Επίτροπος μίλησε για η αρμόδια δεσμευτικά μέτρα έτσι ώστε να εξαλείψουμε με αυτή την καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, η οποία έγκυται στο να ε, παίρνει κανείς χαμηλότερη αμοιβή για ε, εργασία ίδιας και ίσης αξίας. Αυτό πλήττει το συνταξιδοτικό σύστημα, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων, ενισχύει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. άλλωστε η γυναίκα δυσκολεύεται να μπει και να βγει από την αρκορά εργασία και λόγω της εγκυμοσύνης και της τεκνοποίησης. Υπάρχει αυτή η γυάλινη οροφή, όπως γνωρίζουμε που καθιστά πολύ δύσκολο για τη γυναίκα να ανέβει στα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα επιδιορθώσουμε, να τα καταπολεμήσουμε, να έχουμε μια αγορά εργασίας ευέλικτη, ευκίνητη, ε, για να έχουμε περισσότερες ευρωπαϊκές αξίες και περισσότερη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ένα λεπτό, κύριε Γιουγκέρη, έχει τώρα Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Όταν ε, το 87 ξεκίνησα στην πρώτη μου θέση απασχόλησης ήμουν πάρα πολύ ευτυχής. Με μία ομάδα ανδρών και γυναικών ξεκινήσαμε, όλοι μαζί στο ίδιο επίπεδο, κάναμε την ίδια δουλειά και τα ίδια χρήματα παίρναμε. Τουλάχιστον αυτό θεωρούσα τότε, μέχρι όταν ακάλυψα ότι οι άντρες βγάζαν πιο πολλά από ότι εγώ και οι υπόλοιπε γυναίκε υπάλληλοι. Πήγαμε λοιπόν σε μία δικηγόρο, σε έναν δικηγόρο ο οποίο έγραψε μία επιστολή προ την ε, διοίκηση και ευτυχώ δεν χρειάστηκε να παρέμβει ο δικαστή, αλλά αναλάβαμε δράση κατά των ε, διαφορών αυτών των μισθολογικών. Δεν είναι μύθια αυτή, δεν είναι παραμύθια. Η άντρε εξακολουθούν να βγάζουν πιο πολλά από ότι οι γυναίκε. 5.000 παραπάνω το χρόνο κατά μέσο όρο στην Ολλανδία. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Και συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει σύντομα να εισαχθεί νομοθεσία για να υπάρχει διαφάνεια μισθολογική, για να μην μέχρι το 2000, για να μην φτάσουμε το 2021 μέχρι ότου εξαλείψουμε αυτές τις διαφορές τις μισθολογικές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος η κυρία Μάξοβα έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστούμε στην Τσεχική Δημοκρατία. Έχουμε τη διαφορά τη μεγαλύτερη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 21,1% είναι η διαφορά. Παρά που οι Τσέχες γυναίκες έχουν καλύτερη εκπαίδευση, πληρώνονται λιγότερο. Αρκετά συχνά κατέχουν σημαντικές θέσεις, αλλά πληρώνονται λιγότερο. Στον τομέα της ε, παιδείας, των κοινωνικών, κοινωνικής προστασίας, δεν εκπροσωπούνται επαρκώς σε διευθυντικές θέσεις. 15% μόνο των γυναικών στα ε, συμβούλια διοικητικά ε, στην Τσεχική Δημοκρατία. Υπάρχει και το πρόβλημα ε, τις που είναι περισσότερο τις γυναίκες. Οι συνταξιούχες και οι γυναίκες σε μονογονική οικογένεια ζουν στη φτώχεια. Θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση, να εφαρμοστεί ε, η αρχή ίση αμοιβή για ίση εργασία, δυνάμει της οδηγίας για ίση ευκαιρίες του 2006 ή δυνάμει της οδηγίας για τη διαφάνεια τη μισθολογική. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται τη μισθολογική διαφάνεια στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, διότι δεν έχουμε εγγύηση για την ισότητα. Πίτερ Χένσεν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Επίτροπε, πολύ για την εισαγωγή που κάνατε στο θέμα. 4 Νοεμβρίου πέρσι υποτίθεται τελευταία ημέρα εργασία στι 4 Νοεμβρίου έπρεπε να σταματήσουμε στις 4 Νοεμβρίου να μην εργαστούμε το υπόλοιπο έτος, εάν θέλαμε να τηρήσουμε την αναλογία αμοιβή με εργασία. Εργαζόμαστε δωρεάν για το μεγαλύτερο κομμάτι του χρόνου οι γυναίκε. Φέτο θα πρέπει να εστιαστούμε ε, για την ισότητα των φύλων. Χαίρομαι που έχουμε επίτροπο τώρα που έχει αυτό το θέμα ε, που θέλει να προωθήσει, αλλά ο τίτλο δεν αρκεί. Ελπίζω να κάνει αυτό που πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση τη διαφάνεια όσον αφορά τι αμοιβέ στου χώρου εργασία των Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δικαίωμα των γυναικών να ξέρουν αν πληρώνται λιγότερα από του άρενε συναδέλφου που κάνουν την ίδια δουλειά. Ελπίζω επίση ότι η Επίτροπο θα εστιαστεί επί τη οδηγία για την ισορροπία ε, ε, οικογενειακή επαγγελματική ζωή και η άδεια μητρότητα αποτελεί ένα τμήμα του προβλήματο όσον αφορά το ε, μισολογικό χάσμα. Θα πρέπει να μείβονται εξίσου άντρε και γυναίκε. Ε, το Βαλιέρη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, η μεγάλη κλοπή τη ιστορία έτσι καθορίστηκε από τον ΙΕ και εξακολουθεί να μην τιμωρείται αυτή η ληστεία στα μάτια μα. Ακόμα σήμερα στον κόσμο οι γυναίκε κερδίζουν κατά μέσο όρο το 23% λιγότερο από του άντρε. Η Ευρώπη δεν κάνει αρκετά πράγματα, δεν αρκεί το ότι αφιερώνουμε ποσοστώσεις εκπροσώπησης των γυναικών εντάξει, των μεγάλων διοικητικών συμβουλίων, των μεγάλων εταιριών, ε, είναι αντιπροσωπευτικές ποσοστώσεις που δεν αρκούν για να επιλύσουν το πρόβλημα. Είναι μια λύση που δεν είναι φιλελεύθερη. Ε, δεν θα πρέπει να καταστέλει την ελευθερία της επιχειρήσης, θα πρέπει να εκοδηγεί στα κάτι μέλη να καταρρύψουν τα εμπόδια, τα πολιτισμικά και τα οικονομικά που εμποδίζουν την πρόσβαση των γυναικών στα ύψιστα επαγγελματικά και μισθολογικά επίπεδα. Ε, δεν πρέπει να περάσει θασμένο επικίνδυνο μήνυμα ότι οι γυναίκε είναι προστατευμένη κατηγορία από ροζ ποσοστώσει, διότι έτσι τι αποδυναμώνει αντί να τι ενισχύει. Η σωστή αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων των γυναικών είναι η μόνη δυνατή λίστη για να συνδυάσουμε ίση, ε, ίσες ευκαιρίες με ίσες αμοιβέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα η συνάδελφος Ραφάλσκα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Η κατάσταση στην Πολωνία σε ό,τι αφορά το μισθολογικό χάσμα είναι καλύτερη σε σχέση με άλλες αναπτυγμένες χώρες και η κατάσταση αυτή βελτιώνεται διαρκώς. Το 2007 με το 2017 η Πολωνία έκανε μεγάλη πρόοδο σε ό,τι αφορά την κατάσταση των γενικών στην αγορά εργασία. Η Πολωνία λοιπόν πέρασε από την 17η θέση στην 8η σχετική θέση το 2017. Το μισθολογικό χάσμα ήταν 7,2% ενώ στην ίδια περίοδο το κατά μέσο όρο ε, ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 16%. Μόνο η Ρουμανία ήταν σε χαμηλότερο επίπεδο. Αλλά να έχετε υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα είναι πολύ περίπλοκο φαινόμενο, το οποίο έχει να κάνει και με πολλούς διαφορετικού παράγοντες που επηρεάζουν την ε, κατάσταση των ανθρώπων και των γυναικών στην αγορά εργασίας. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν την εμπειρία, το επάγγελμα και το καθεξής. Επίσης να έχουμε υπόψη είναι ότι οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τη ζωή τους και το επαγγελματικό τους, την πολιτική τους εξέλιξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συνάδελφος Ροντρίγκες Παλόπ για ένα λεπτό, λέει πρόεδρος. Ε, Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι γυναίκες δουλεύουν δύο μήνες δωρεάν το χρόνο συγκριτικά με τους άνδρες γιατί τόσο πολλοί δουλεύουν σε συνθήκες δουλείας χωρίς να αμείβονται. Γιατί γιατί οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες φροντίζουν τον οικοκυριό και τα παιδιά ε, και τους υλοκιωμένους στο σπίτι με άτυπο και μη αμοιβόμενο τρόπο μεταξύ άλλων. Γνωρίζουμε τα μέτρα που πρέπει να θετήσουμε, αλλά δεν το κάνουμε. Πρέπει να υποχρέσουμε να υποχρεώσουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις να ε, υποστούν ελέγχους από την επιθεώρηση εργασίας και να επιβάλλουμε κυρώσεις. Όταν γίνεται διάκραση σε βάρος των γυναικών, όταν αυτές θέλουν να τεκνοποιήσουν. Η εκπαίδευση των ε, παιδιών ε, σε νηπιακή και βρεφονηπιακή ηλικία είναι κάτι το εξαιρετικά ακριβό και δεν προσφέρεται σε όλους. Δεν υπάρχει πρόσβαση ε, επίσης σε ένα σύστημα πρόνοιας και φροντίδας της τρίτης ηλικίας, έτσι ώστε να μην πέφτει το βάρος της φροντίδας των ηλικιωμένων μελών της οικογένειας στη γυναίκα, η οποία τελικά βγάζει τρία μεροκάματα, τρία οχτάρα δουλεύει. Ε, δεν έχουμε αρκετή κοινωνική κάλυψη και έχουμε ε, πολύ μικρή μισθολογική ε, ανταμοιβή των γενικών. Νομίζω ότι κάνουμε τα ελάχιστα και είναι πολύ δυστυχέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διάκριση μισθολογική είναι μια μορφέ ανισότητα κοινωνική που είναι πιο διάχυτη και εμποδίζει τι γυναίκε να συμμετέχουν πλήρω στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τη χώρα του. Αυτή η διάκριση σχετίζεται πολύ με την οτροπία και τα στερεότυπα που χαρακτηρίζουν σήμερα τα κοινωνικά μοντέλα και την αγορά εργασία σε εθνικό επίπεδο. Επίτροπε Ντάλη, η πρόταση για διαφάνεια όσον αφορά τι αμοιβέ είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε. Αλλά σαν κίνημα πέντε αστέρε, σα ζητούμε η νέα πρόταση τη οδηγία να μην αντιπροσωπεύει μήπω άλλο ένα κατάλογο τη αρχή των καλών προτάσεων. Αλλά θα πρέπει να αναφέρει λύσει στα κράτη-μέλη για να επιλύσει άπαξ διαπαντό το πρόβλημα τη ε, διαφοροποίηση των φύλων στα διάφορα επαγγέλματα, στου διάφορου τομεί δραστηριοτήτων. Απομόνωση και διαφοροποίηση που είναι βασικό αίτιο της, ε, του μισθολογικού χάσματος των κυναικών. Θα πρέπει να συζητήσουμε ένα σύστημα αναρμονισμένων κυρώσεων που θα επιβάλλει κυρώσει εκείνων που προφανώς παραβιάζει την μισθολογική ισότητα και εκμεταλλεύεται σκόπιμο την εργασία των γυναικών ε, και αυτό στέφεται κατά της δικαιοσύνης της κοινωνικής. Σα ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει συνάδελφο κυρία Φράντσνα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε αξιότιμη επιτροπέ, το μυστολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων εξακολουθεί να αποτελεί μια βασική πρόκληση. Και το 2020 οι γυναίκε εξακολουθούν να βγάζουν πιο λίγα από ότι οι άντρε. Και εδώ πέρα οι ανισότητε εντείνονται και στι συντάξει. Θα πρέπει λοιπόν να κατεπηγόντω κάτι να γίνει. Πολλά έχουμε ακούσει. Δύο πράγματα θέλω να τονίσω. Οι γυναίκε έχουν πιο συχνά μερική απασχόληση και αυτό οδηγεί σε χαμηλότερο μισθό και έτσι είναι σε πιο ευάλωτη κατάσταση. Έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για φτώχεια. Και η μείωση του μυστολογικού χάσματος σημαίνει ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και την ε, κατανομή των ήπιων καθηκόντων και αυτό θα πρέπει να σημαίνει και η εφαρμογή, η εφαρμογή της ίσης αμοιβή για ίση εργασία σε ό,τι αφορά και τις αρχές που τόνισε η Μάριαν Τέισεν. Όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν. Δεύτερο στοιχείο θα πρέπει να ε, κοιτάξουμε εγκάρσιες και σε διακρίσεις στην αγορά εργασίας, να σταματήσουν τα στερεότυπα και ο, ο ψηφιακός κλάδος είναι το μεγάλο μήνυμα. Θα πρέπει να δοθεί λοιπόν μεγαλύτερη όθηση προς τις γυναίκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συνάδελφος αδελφός κυρία Φρίτσον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Επίτροπο για την πολύ καλή εισαγωγή που έκανε. Η αρχή της ίσης αμοιβής για συνεργασία μεταξύ γυναικών και ανδρών έχει κατοχυρεωθεί από... έχει μάλλον αναφερθεί στι ευρωπαϊκές συνθήκες το 57 και τώρα 63 χρόνια αργότερα βρισκόμαστε και οι γυναίκες εξακολουθούν να βγάζουν πιο λίγα από ότι οι άντρε για την ίδια δουλειά. Είναι το ότι δεν έχουμε σημειώσει πιο πολύ πρόοδο, ότι δεν έχουμε αναλάβει μεγαλύτερη δράση προκειμένου οι γυναίκες να βγάζουν τα ίδια όσο οι άνδρες. Και φυσικά είναι ντροπή ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακηρύττουμε τις αξίες μας αυτές και δεν ε, μπορούμε να υλοποιήσουμε την ίδια τη συνθήκη. Χρειάζεται πολιτική βούληση λοιπόν για να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Αν ρωτιέμαι λοιπόν, τι να πω στις κόρες μου. Έχει νόημα να τους πω ότι κοιτάξτε καλά πτυχία έχετε, αλλά σε σχέση με του άντρε, θα πρέπει να δουλέψετε δύο μήνε χωρί αμοιβή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρο. Η συνάδελφο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σήμερα συζητάμε ένα θέμα που θα έπρεπε να είχε λήξει, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκε ε, αμοιβόμαστε κατά 16% λιγότερο από ότι οι άνδρε και γι' αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία σε θέματα ισότητα, να αναθεωρήσει το συντομότερο δυνατό τη σχετική οδηγία, να μα προβάλλει και να μα παρουσιάσει μέτρα που θα υιοθετηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συμφιλίωση εργασιακή και οικογενειακή ζωή. Ξέρετε, εγώ είμαι μηχανικό και με ενδιαφέρει ε, ο αντίκτυπο τη ψηφία στο μισθολογικό χάσμα. Πολλά θέματα εργασίας θα ε, υπάρξουν πολλά, πολλές θέσεις εργασίας, θα υπάρξουν πολύ καλά αμοιβόμενε ε, και σε αυτούς τους κλάδους η παρουσία η γυναικεία είναι πολύ ε, χαμηλή. Κατά 17% λιγότερο εκπροσωπούνται οι γυναίκες σε αυτούς τους κλάδους της ψηφιοποίησης, της τεχνολογίας. Πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε να είναι περισσότερες οι νεαρές οι οποίες θα ακολουθήσουν αυτή την εκπαίδευση, αυτές τις σπουδέ και θα μπορέσουν να στελεχώσουν αυτούς τους κλάδους. Ιδαλλιώς το μισθολογικό χάσμα θα οξύνεται αφού θα θα έχουμε μικρότερη παρουσία γυναικών στις υψηλά αμοιβόμενες θέσεις και τους υψηλά αμοιβόμενους κλάδους. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Φίλιπς, ε, η οικονομία ουσιαστικά οδηγείται από κλέφτες, γιατί οι γυναίκες ε, ουσιαστικά είναι θύματα κλοπής και καθημερινά έχουν μία σύνταξη η οποία είναι κατά μέσο όρο 35% χαμηλότερη από ό,τι οι άνδρες. Για τις ε, γυναίκες λοιπόν που έχουν θέματα σε ό,τι αφορά την... είναι μετανάστριες, ε, έχουν θέματα σεξου... είναι διαφορετικές σεξουαλικής προσανατολισμού, το θέμα αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο και στο, στον Εμένο Βασίλειο η ίση αμοιβή κατοχυρώθηκε νομικά το 1970. Ακόμα όμω σήμερα επαναλαμβάνουμε τις ίδιες αρχές εκ νέου. Αν κάποιο έβλεπε σε λεωφορείο έναν κλέφτη να κλέβει ε, ένα χαρτονόμισμα από την τσέπη μία γυναίκα, θα έβγαινε και θα το κατέκυλε και θα φώναζε αστυνομία. Κλέφτη. Αλλά έτσι θα πρέπει να αντιδράσουμε και τώρα, να φωνάξουμε και να πούμε ότι οι γυναίκε δεν μπορούν να περιμένουν άλλα 50 χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφο κυρία Μπρούνα για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μια γυναίκα που κάνει την ίδια δουλειά και έχει τα ίδια καθήκοντα θα πρέπει να έχει τον ίδιο μισθό για την ίδια δουλειά, ίδια αμοιβή. Ε, αυτό πρέπει να κάνουν τα εθνικά κράτη και αυτή η αρχή πρέπει να γίνει σε σεβαστή. Τώρα συζητάμε για το μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών, δηλαδή διαφορά στην αμοιβή ε, μεταξύ των δύο φύλων που μπορεί να εργάζονται ε, με την ίδια εμπειρία και στι ίδιε θέσει. Η διαφορά αυτή έχει να κάνει και με τις επιλογές ε, των γυναικών. Θα πρέπει η αμοιβή να είναι ίδια για την ίδια δουλειά και θα πρέπει οι γυναίκες να έχουν πρόσβαση στι ίδιε θέσει και την ίδια αμοιβή με του άντρε. Ωστόσο, εδώ βλέπουμε να υπάρχουν απόψει που ε, δίνουν άλλε αποχρώσεις στι διαφορέ ανδρών και γυναικών. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι οι γυναίκες θα πρέπει να αναβάλουν την ε, ε κυοφορία ε, και να παγώνουν τα ωάριά τους προκειμένου να ανταποκρίνονται στις επαγγελματικέ τους υποχρεώσεις. Ευχαριστούμε συνάδελφος Στέκρουτ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Η διαφορά στο εισόδημα αντρών και γυναικών ύψους σε 16% σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν οφείλεται στην διάκριση. Η Σουηδία είναι μια από τις χώρες του κόσμου με ε, τη μεγαλύτερη ισότητα ενώ έχει ε, διαπιστωθεί ότι στη Σουηδία δεν, υπάρχει, ε, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η διαφορά αυτή οφείλεται σε διακρίσεις αλλά έχει να κάνει με τη διαφορά τις ε, ώρες που εργάζονται, ε, ε, το είδος τη δουλειάς κτλ. Θα απαιτούνταν απολυταρχικές μέθοδοι για να έχουμε ίση αμοιβή κάτι που περιορίζει τις επιλογές του κάθε ατόμου. Πρέπει η δουλειά πάνω στην ισότητα να βασίζεται σε δεδομένα και όχι σε υπερβολικούς μύθους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα ο συνάδελφος Νικαλό Αλαβάνος για να λυθώ. Η λεγόμενη πολιτική της συμφιλίωσης οικογενειακής επαγγελματικής ζωής των ίσων ευκαιριών μέσα στις εισαγωγικά έχει οδηγήσει στην πλήρη ευελιξία του εργάσιμου χρόνου και του χώρου εργασίας για τη γυναίκα εργαζόμενη με αποτέλεσμα στην ευρωπαϊκή ένωση το 1 τρίτο των γυναικών να δουλεύουν με μερική απασχόληση. οι ευέλικτε εργασιακέ σχέσει είναι ένα από του παράγοντε που στην ελλάδα ευθύνονται για παράδειγμα για το γεγονό ότι ο μισθό τη γυναίκα είναι τη γυναίκα εργαζόμενης κατά 17,5% χαμηλότερο σε σχέση με του άντρε ενώ στην ευρωπαϊκή ένωση η μέση διαφορά των αποδοχών φτάνει έω και το, κοντά στο 40%. τα σύγχρονα δικαιώματα των γυναικών στην εργασία δεν εξασφαλίζονται με την εξίσωση των απολαβών για άντρε και γυναίκε προ τα κάτω όπω κάνει η ευρωπαϊκή ένωση ιδιαίτερα σε μια περίοδο που το κεφάλαιο για τη βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων συστηματικά ξυλώνει την προστασία τη μητρότητα άδειε και επιδόματα τα οποία τα θεωρεί κόστο εξαναγκάζοντα χιλιάδε εργαζόμενε στην ανεργία στη μισή δουλειά μισή ζωή. η αποφασιστική πάλι των εργαζομένων ενάντια στην επιθετικότητα τη ευρωπαϊκή ένωση των αστικών κυβερνήσεων μπορεί να προσδώσει νέα πνοή και δύναμη στην εργατική λαϊκή πάλι για τι σύγχρονε ανάγκε στην εργασία στην κοινωνική προστασία της μητρότητας στον ελεύθερο χρόνο. Ευχαριστώ η συνάδελφος Hübner. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, η Ευρώπη πρέπει να ανανεώσει την ενότητά της, να κοιτάξει πέρα από τον ορίζοντα και το να διατηρεί ε, την ψαλίδα στις αμοιβέ ανδρών και γυναικών ε, είναι αναχρονιστικό. Όταν οι πιο έξυπνες γυναίκες έχουν χαμηλότερες αμοιβέ από τους άνδρες συναδέρφους τους, αυτό περιορίζει και τον, την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να προετοιμαστούμε για τον 21ο αιώνα πρέπει να απαλλαγούμε από αυτήν την διαφορά του 16%. Στο μέλλον ε, η αγορά, δεν θα είναι, η αγορά εργασίας δεν θα είναι απαραίτητα πιο φιλική ε, προς τις γυναίκες. Ενθαρρύνονται οι γυναίκες να αποκτήσουν δεξιότητες και να μάθουν νέες τεχνολογίες, αλλά ε, το χάσμα στις αμοιβέ μπορεί να αυξηθεί στο μέλλον. Και γι' αυτό είμαι πεπισμένη ότι το Κοινοβούλιο θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να στηρίξει την ε, προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να κλείσει τελείως το χάσμα. Ευχαριστώ. Γκουαλμίνη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Επίτροπε, για να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό το μισθολογικό χάσμα, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ξαναβρούμε κοινωνική δικαιοσύνη. Άλλωστε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το μισθολογικό χάσμα, είναι και αυτέ οι γυάλινε οροφές, τι οποίε υφίστανται στη διάρκεια όλη τη σταδιοδρομία τους ε, οι γυναίκε. Επίση, το γεγονό ότι πολύ συχνά είναι οι μόνες παρέχουσε φροντίδα στο σπίτι. Ε, οι γυναίκε επίση συχνά δεν θεωρούν θεωρούνται αρκετά κατάλληλες για κάποιες θέσεις και επίσης πάνω από 30% των γυναικών μία φορά τουλάχιστον στη ζωή τους έχουν, υπο, ε, ε, έχουν ε, αποτελέσει κειμενοβία. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δράξουμε την ευκαιρία έτσι ώστε οι γυναίκες πια να γίνουν πραγματικά ίσες με τους άντρες και οι γυναίκες να αποκτήσουν συγγνώμη συνείδηση του γεγονότος ότι είναι το ίδιο ικανό με με του άνδρε έχουν την ίδια αξία με του άνδρε. Α ξεκινήσουμε λοιπόν την προσπάθεια να μειώσουμε, να κλείσουμε αυτό το μισθολογικό χάσμα. Θα είμαστε πάντα κοντά σα και εμεί πάντω δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ αυτόν τον αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. σα ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Και τώρα ο λόγο στη συνάδελφο Ραφαέλα για ένα λεπτό. Madam Commissioner, achieving... Κύριε Επίτροπε, η επίτευξη ε, ίσων αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι προϋπόθεση εκ των να αισθανθούν και οι γυναίκες ελεύθερες. Οι γυναίκες δεν έχουν την ίδια ελευθερία λόγω ακριβώς του μισθολογικού χάσματος ε, που παραμένει στο 16% σχεδόν απαράλλαχτο και μη μετακινούμενο τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Ε, οπισθοδρομούμε λοιπόν και θα συνεχίσουν οι γυναίκες να ε, δρομούν ενώ ε, οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν τα μάλλα στην οικονομική ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, θέσει ως προτεραιότητα το θέμα των γυναικών, της ενεργού συμμετοχής τους ε, στην κοινωνία και του κλεισίματος του μισθολογικού χάσματος. Θα πρέπει να κατανοήσουμε το χάσμα ωραία, αλλά κυρίως θα πρέπει να κλείσουμε το χάσμα αυτό. Οι συγμένες λοιπόν εταιρείε και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι απολύτως διαφανείς στον τρόπο με τον οποίο φέρονται στις υπαλλήλου τους και στον τρόπο με τον οποίο ε, ε, ε, δρούν έτσι ώστε να κλείσει το χάσμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο λόγος του συνάδελφου Μπεάτα Σιζίλντο. Κυρίες και κύριοι, επίτροπε. Αυτό είναι ένα από τα μείζωνα ζητήματα που συζητούμε σήμερα. Το μισθολογικό χάσμα θα έπρεπε να είναι ένα από τα πλέον ουσιώδη με τα οποία ασχολείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχει να κάνει με την ισότητα των δικαιωμάτων. Ισότητα για όλους, ασχέτως του που κατοικούν και το, της προέλευσής τους, ή το που εργάζονται. Στην Πολωνία έχουμε προβλέψει μια λύση για το θέμα αυτό. Και μάλιστα εξαλείψαμε τη φτώχεια. Όπως είπαν προηγουμένως οι Πολωνοί συνάδελφοι, μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες θέλουν να εργάζονται, θέλουν ε, να ναι, ε, δραστήριες επαγγελματικά, αλλά θέλουν να μπορούν να επιτελέσουν και τα καθήκοντά τους ως μητέρες. Θέλουν να αναθρέψουν τα παιδιά τους. Γι' αυτό έχουμε προβλέψει ειδικό επίδομα για τις γυναίκες που έχουν τουλάχιστον τέσσερα παιδιά. Και είναι χαρακτηριστικό της σημερινής συζήτησης ε, το γεγονός ότι κυρίως οι γυναίκες ε, ζητούν το λόγο. Όλοι στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασχολούνται με την επίλυση του ζητήματος αυτού. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και τώρα ο λόγος στη συνάδελφο Μαρία Ντεγκράσα Καρβάλιου για ένα λεπτό. Πρόεδρε, Επίτροπε, με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μέσα στις 100 πρώτες μέρες της θητείας της προτείνει μέτρα για την μισθολογική διαφάνεια μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ωστόσο, η αρχή τη ίση αμοιβή για ίση δουλειά είναι κάτι που ούτω ή άλλω προβλέπεται από τι συνθήκε. Κι όμω, η πραγματικότητα στην πράξη είναι εντελώ διαφορετική με μεγάλε ανισότητε μεταξύ των κρατών μελών. Παραμένει ένα παράγοντα δικαιωτική μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Γιατί ε, οι γυναίκε σε μεγάλη, σε τομεί αυξανόμενη σημασία στην κοινωνία, όπω τι επιστήμε των υπολογιστών ή στι ψηφιακέ τεχνολογίε, η επαναχώρηση. Εδώ λοιπόν δεν πρέπει να περιορίσουμε κι άλλο την πρόσβαση των γυναικών στις ε, καλά αμοιβόμενε θέσει εργασία. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, μέτρα που θα επιτρέπουν τη συμμετοχή των γυναικών και θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό. Και θα πρέπει να έχει και την τολμή για να ξεμπλοκαριστούν οδηγίε που ε, καλύπτουν ακριβώ την ε, σωστή μισθολογική αμοιβή των γυναικών. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Και τώρα ο λόγος Jackie, στην συνάδελφο Τζάκι Τζόντς. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. Όταν ήμουν παιδί τη δεκαετία του 1971, ε, πέρασε, εγκρίθηκε μια σειρά νομοθετικών μέτρων για την ισότητα πάνω, πριν από 40 χρόνια είχαμε την ε, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για ε, την εξάλληψη των διακρίσεων και στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Μετά από διάφορες υποθέσεις εγκρίθηκαν πολλές οδηγίες εδώ και 50 χρόνια. Ωστόσο δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που να αμύδει ίσα την ίδια εργασία. Γιατί λόγω διακρίσεων δεν υπάρχει ούτε μία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει ίση αμοιβή. Πρέπει να κλείσουμε το χάσμα. Εγώ γερνάω, θα αποχωρήσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήλπιζα κατά τη διάρκεια τη ζωή μου ε, να δούμε ισότητα και προώθηση των γυναικών ε, και ε, μια αναθεωρημένη οδηγία για την ίση αμοιβή που θα πρέπει να αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής για την ισότητα των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Δώστε μου να αναφερθώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, τώρα που εγκαταλείπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είπε κατά λάθο η ομιλήτρια. θα ήθελα στην κυβέρνηση Τζόνσον να πω ναι, να ε, αναλάβετε τον έλεγχο λέτε, αλλά τώρα ε, να κλείσουμε το μισθολογικό χάσμα, ε, το χάσμα στις συντάξεις και να δώσουμε στις γυναίκες την σύνταξη που τους αξίζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα η συνάδελφος Μπιλμπάο Μπαραντίκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η συνθήκη της Ρώμης ε, ε, ε κατήγγειλε και έκανε τα πρώτα βήματα για το κλείσιμο του μισθολογικού ε, χάσματος. ξεκίνησε δε από, την, από τις χείρες των πεσόντων στο μέτωπο που έπαιρναν λιγότερο από τους, τους υπόλοιπους από τους άνδρες. αλλά βεβαίως το θέμα είναι εδώ να μπορέσουμε να ε, ε, βρούμε μια νέα τάξη πραγμάτων έτσι ώστε ε, νέα ταλέντα να μπορέσουν να αναδειχθούν. Είναι γεγονός ότι το μισθολογικό χάσμα φτωχαίνει όλο τον κόσμο. Η πρόεδρος Φόντερ Λάγεν αναφέρθηκε και στην γυάλινη ορυφή. Ελπίζω πάντως ότι μετά το τέλος της θητείας αυτής της Επιτροπής θα υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μισθολογική ισότητα. Θα έχει κλείσει αυτό το χάσμα. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Μοντζανόφσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα, διότι ασχέτως φίλου, όλοι μιλάμε για το κλείσιμο του μισθολογικού χάσματος που ε, αφορά ε, τις περισσότερες χώρες και τις γυναίκες στις χώρες αυτές. Σήμερα είναι η μέρα που μιλάμε με μία φωνή και όπου επιστρατεύουμε όλα μας τα επιχειρήματα για να βρούμε συστημικές λύσεις. Ε, χρειάζεται όμως να συνεργαστούμε και με τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες. Ε, μια προσωπική ιστορία να σας πω. Όταν ήμουν υφυπουργό ε, ανάπτυξης στην πολωνική κυβέρνηση είχα ανταλλαγή απόψεων με επιχειρήσεις και βρήκαμε διάφορες συνεργατικές λύσεις. Η πολωνική κυβέρνηση, για παράδειγμα, ε, βρήκε ένα μέσο που ε, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να υπολογίσουν ε, τις ανισότητες. Μπορείτε, μπορεί κανείς να υπολογίσει και την μέση αμοιβή στον τομέα του και να τη συγκρίνει με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι μπορούσαν οι επιχειρήσεις ίδιες να ελέγχουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Αυτό σε συνδυασμό με τρόπους υποστήριξης της οικογένειας προσπαθούν να βελτιώσουμε την ισορροπία ανάμεσα στην ιδιωτική και επαγγελματική ζωή. Ε, αλλά ε, η πρόοδος είναι αργή, γι' αυτό πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Ευχαριστούμε και τώρα ο λόγος στην συνάδελφο Σόιντροβα για ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι, η οι διακρίσεις, δηλαδή διαφορετική αμοιβή για την ίδια εργασία είναι παράνομη. Ο νόμος λέει ε, ίση αμοιβή για την ίδια δουλειά. Παρ' όλα αυτά έχουμε μισολογικό χάσμα ύψους 16%, 16% και σε κάποιες χώρες είναι μεγαλύτερο το χάσμα αυτό, ε, συμπεριλαμβανομένες της Τσεχίας όπου είναι 22%. Ε, πρέπει να εξετάσουμε φυσικά το ρόλο της μητρότητας, αλλά εάν δεν θέλουμε η μητρότητα και η οικογενειακή ζωή να είναι ο δρόμος προς την καταστροφή. Θα πρέπει ε, να εκτιμήσουμε το ρόλο των γυναικών ε, ως μητέρες και τον ρόλο των γονέων γενικά. Θα πρέπει το κράτος και οι εργοδότες να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι οι νέοι γονείς χρειάζονται ένα νέο ξεκίνημα στη δουλειά τους ε, όταν επιστρέφουν από τη γονική άδεια. Κυρία ε, Επίτροπε, ε, παρακαλώ να διασφαλίσετε την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία ανάμεσα στον οικογενειακό και επαγγελματικό βίο. Οι γυναίκες θα πρέπει να είναι πιο καλά ενημερωμένες ώστε να μπορούν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Θα πρέπει να εκτιμούμε τη μητρότητα χωρίς να γίνονται διακρίσει εξαιτία αυτή. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο συνάδελφος Μάρκ Αντζέλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, τα στερεότυπα, τα με έμφυλα κλισέ ε, είναι αυτά τα οποία δείχνουν στην ουσία τα όσα υφίστανται οι νέες γυναίκες ε, είτε στην αγορά εργασίας είτε και όταν έχουν πλέον συνταξιοδοτηθεί. 16,3% η διαφορά η μισθολογική αλλά πολύ μεγαλύτερη η διαφορά εισοδήματος τεράστια αντίθεση με την ε, κοινωνική Ευρώπη του Γκέτεμπουργκ του 1997. Αυτές ε, οι ανισορροπίες ε, είναι ακριβώς αυτές οι οποίες απορρέουν από την πατριαρχικά δομημένη κοινωνία. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν δεσμευτικά μέτρα, να ξεμπλοκάρει η οδηγία, να γίνει ξεκάθαρος ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων, να υπάρξει συγκεκριμένη δράση κατά των κοινωνικών ε, στερεοτύπων ε, και οποιονδήποτε άλλων κοινωνικών προβλημάτων. Um Ευχαριστώ πολύ και τώρα ένα λεπτό για τη συνάδελφο Μελμπάρντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι, επιτροπέ, είναι θλιβερό που όχι μόνο οι γυναίκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν περίπου το 1 πέμπτο λιγότερο από ό,τι οι άντρε, αλλά και το μισθολογικό χάσμα έχει αυξηθεί κατά 1% τα τελευταία 7 χρόνια. Και μάλιστα ακόμα χειρότερο, οι γυναίκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν λιγότερη εκπαίδευση από ότι άντρε. Ε, είναι πολύ θλιβερό και για τι ε, ανώτατε θέσει, τα ανώτατα κλιμάκια στι εταιρείε και τι επιχειρήσει. Η ισορρόπηση στι θέσει των, ε, των και το πόσο προσλαμβάνονται ε, οι γυναίκες σε ε, μεγάλες επιχειρήσεις, σε υψηλές θέσεις, είναι πολύ θλιβερό σε σύγκριση με χώρες όπως την Ισία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ε, γυναίκες δάσκαλοι ε, και καθηγητές πληρώνονται λιγότερο από ότι άντρες. Όμως, δεν είναι μόνο εξισορρόπηση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου που θα πείσει τι γυναίκε να, να αναζητήσουν μια κατάλληλη επαγγελματική σταδιοδρομία, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και το στοιχείο όπου ε, τα επαγγέλματα όπου κυριαρχούν οι γυναίκες όπως οι γραμματείς είναι πιο ευάλωτα σε σχέση με αυτά όπου τα μονοπολούν οι άντρες. Θα πρέπει λοιπόν το ζήτημα αυτό να το αντιμετωπίσουμε σφαιρικά και να κοιτάξουμε να χτυπήσουμε την αδικία ε, στη ρίζα της. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, η συνάδελφός σου Τσάνα Γκλάβακ για ένα λεπτό. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Επίτροπε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι τις 4 Νοεμβρίου του, ε, ε θα ε, ε, ε, άρχισαν να δουλεύουν με μισθό. Πραγματικά αυτή η δωρεάν εργασία θα πρέπει να σταματήσει. Είπαμε ότι υπάρχει 16% διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες και σε βεβαίως αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με τους άνδρες οι γυναίκες δύο μήνες κάθε χρόνο δουλεύουν δωρεάν. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Ε, πέρα όμως και πάνω από όλα αυτά υφίστανται ε, και στο τέλος της σταδιοδρομίας τους ε, μεγάλο χάσμα όσον αφορά την σύνταξή τους και επομένως αυτό προκαλεί κοινωνικό αποκλεισμό αλλά και μεγάλο βαθμό εξάρτησης των γυναικών αυτών από τους ε, συζύγους τους. Θα ήθελα τελειώνοντας να δώσω ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει αυτούς που παίρνουν αποφάσεις. Το αποτέλεσμα μιας έρευνας του ε, Διεθνούς ε, Ινστιτούτου Μακένση, όπου δείχνει ότι το διεθνές ε, ΑΕΠ θα μπορούσε ε, να αυξηθεί ε, κατά 1-3-200 δις δολάρια εάν οι γυναίκες είχαν την ίδια αμοιβή και πραγματική ισότητα με τους άντρες. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό για τον συνάδελφο Ρόμπερτ Πιεντρών. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι. Η αρχή της ίσης αμοιβή για άντρες και γυναίκες ε, ισχύει από το 1957. Επί 63 χρόνια περιμένουν οι γυναίκες να αρχίσει να εφαρμόζεται στην πράξη η αρχή αυτή και περιμένουν ακόμα. Εάν δεν εισάγουμε κατάλληλη νομοθεσία, όλες οι έρευνες συμφωνούν ότι η ίση αμοιβή θα εφαρμοστεί σε 257 χρόνια. Το 2272. Κανείς μας δεν θα ζει τότε να δει τη μέρα εκείνη. Κυρία Επίτροπε, λοιπόν, θα ήθελα να δηλώσω εδώ και τώρα. ότι όλοι χρειάζεται να έχουμε την ίδια αποφασιστικότητα με σας. Πολλοί άντρες εδώ στο Κοινοβούλιο ε, συμμερίζονται την αποφασιστικότητα αυτή, όπως και ε, πολλές γυναίκες που πήραν το λόγο. Θέλουμε λοιπόν να σπάσουμε ε, την τελευταία γυάλινη οροφή που εμποδίζει τις γυναίκες να πετύχουν την πολιτική ισότητα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια αυτή, κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ. συνάδελφοι, ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις βάσει του καταλόγου αγορητών. Ακολουθεί η διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΕ, προσέλκυση της προσοχής του Προέδρου. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε δίκη κατανομή του χρόνου μεταξύ των πολιτικών ομάδων και έχοντας υπόψη ότι κάποιοι ήδη έχουν λάβει το λόγο κατά την προηγούμενη φάση της συζήτηση. Πρώτα λοιπόν ο λόγος στη συναδέλφο Βιρκούνεν για ένα λεπτό. Πρόεδρε, στην Ευρώπη οι γυναίκες έχουν καλύτερη εκπαίδευση από τους άντρες και όμως κερδίζουν 16% λιγότερο από ό,τι εκείνοι. Γιατί? Ερωτώ γιατί οι γυναίκε δουλεύουν περισσότερο σε θέσει μερική απασχόληση. Χρειάζονται περισσότερες άδειε. γονικέ, με μητρότητα. Περισσότερο από ότι οι άντρε. Τα συμβόλαιά του είναι περιορισμένου χρόνου και έχουν και λιγότερο μισθό, αμοιβή, από ότι οι άντρε για την ίδια δουλειά. Είναι λοιπόν άκρο σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί σοβαρά με το ζήτημα αυτό και να προτείνει κάποια νομοθεσία για να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την ε, αμοιβή. Ακόμα και η γονική άδεια μητρότητα ή πατρότητα πρέπει να διανέμεται και να κατανέμεται σωστότερα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η σχετική οδηγία είναι ήδη αρκετά καλή, όμω το τίμημα το πληρώνουν οι γυναίκε. Οι γυναίκε παίρνουν και 36% λιγότερη σύνταξη από του άνδρες επειδή ακριβώ έχουν ε, εξαντλήσει την άδειά του. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ευχαριστούμε πολύ. Η ε, συνάδελφος Μαργαρίδα Μάρκης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας την Επίτροπο για την παρουσίαση που μας έκανε εδώ και πάνω απ' όλα γιατί μας λέτε ποιες θα είναι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε εμπιστοσύνη στην θητεία σας, διότι δεν μπορούμε να έχουμε μια επιτρόπο που να είναι υπεύθυνη για την ισότητα των ευκαιριών και να μην έχει την εξουσία εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κάνει κάτι γι' αυτό ε, και τη δυνατότητα επίσης να επηρεάσει τους υπόλοιπους επιτρόπους του Κολεγίου, του Κολεγίου των Επιτρόπων. Παρόλα αυτά χρειαζόμαστε και μια σφαιρικότερη στρατηγική και ελπίζουμε ότι αυτή η σφαιρική στρατηγική θα συμπεριλαμβάνει διαφορετικές παραμέτρους, όλες τις παραμέτρους δυνατόν. Θα ήθελα εδώ να επενθυμίσω ότι είναι γεγονός ότι υπάρχει χάσμα 16% στην μισθολογική απόκληση ανδρών γυναικών. Η διαφορά αυτή έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ε, μελλοντική ζωή των γυναικών και επίσης και στη σύνταξή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο λόγος τώρα στον ε, συνάδελφο Σποτόφ για ένα λεπτό. Ε, ίσως μισθός για ίση δουλειά. Αυτό επιδιώκουμε και αυτό ακούμε. Μισθολογικό χάσμα. Αλλά τώρα το πρόβλημα είναι χειρότερο, διότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι σε πολλού τομεί η κατάσταση έχει επιδενωθεί. Ε, και οι γυναίκε παίρνουν λιγότερα από το γενικό μέσο όρο. Οι γυναίκε θέλουν επαγγελματική σταδιοδρομία. Όμω τι κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι έχουν πραγματικά την επιλογή. Υπάρχουν εκπαιδευτέ στα σχολεία που λένε στα παιδιά ότι τα αγόρια είναι πιο ε, καλά στα θετικά ε, μαθήματα και τα κορίτσια πρέπει να ασχολούνται με τα του σπιτιού. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να σταματήσουμε να μεγαλώνουμε τα κορίτσια καλά και είναι μικρά λουλουδάκια ενώ τα αγόρια ήρωε. Θα πρέπει οι ρόλοι αυτοί που σχετίζονται τα στερεότυπα των φίλων να αλλάξουν. Θα πρέπει να αλλάξει αυτή η εκπαίδευση που βασίζεται στα έμφυλα πρότυπα και να κοιτάξουμε πώς επηρεάζεται και η επιλογή τη επαγγελματική σταθερομίας. Θα πρέπει να ε, σκεφτούμε πραγματικά προγράμματα με πραγματική ε, επίδραση στην πραγματικότητα. Ευχαριστούμε και τώρα ο λόγο στη συνάδελφο ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το μισθολογικό χάσμα δεν είναι μύθος παλαιός ή νέος όπως ακούστηκε προηγουμένως. Είναι αντιθέτως ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και πρόβλημα οικονομικό, γιατί εμείς ε, οι γυναίκες ε, είμαστε ε, ε, ε διπλωματούχες πανεπιστημίου. Είναι γεγονός ότι το μισθολογικό χάσμα μειώνεται, αλλά ειδικά την τελευταία δεκαετία με πολύ αργό ρυθμό και πιστεύω ότι αυτή η οδηγία για την διαφάνεια ναι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη αλλά πιστεύω ότι δεν θα είναι επαρκής γιατί ε, οι πιο απαιτητικές και καλύτερα αμοιβόμενες εργασίες ε, αφορούν την τεχνολογία ε, και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας η παρουσία των γυναικών στον τεχνολογικό τομέα μειώνεται διαρκώς κατά 17% έχει μειωθεί. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα κατά την έννοια αυτή και να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό με ευρύ τρόπο. Επομένως η ερώτησή μου είναι η αξίση και συγκεκριμένη ποια είναι τα μέτρα τα οποία τα συγκεκριμένα θα πάρετε για να μειώσετε το μισθολογικό χάσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό για την ε, Κατρίνα Κονέκτα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κυρία Επίτροπε, οι διαφορές οι μισθολογικές ε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, υπάρχει διαφορά και ανάμεσα στα φύλλα και ανάμεσα στις χώρες και ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Ε, το μισθολογικό χάσμα ε, είναι πολύ μεγάλο και από τα στοιχεία τα οποία είναι πιο δια παρουσιάζουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα χάσματα επηρεάζουν την καθημερινή ζωή, την εργασιακή ζωή, αλλά και μετά το πέρας αυτής την ζωή κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης. Δεν ε, υπάρχει καμία λογική βάση για οποιαδήποτε μισθολογική διαφοροποίηση. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει πραγματικά ε, να μιλά για ε, δικαιώματα των πολιτών, θα πρέπει οπωσδήποτε να καταπολεμήσει το μισθολογικό χάσμα. Η, η Ζαμπέλ Καρβάης, τελευταίο ομιλητρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, Είμαστε ήδη ε, στον 21ο αιώνα και έχει προχωρήσει και συζητάμε ακόμα τις ανισότητες ανδρών και γυναικών. Ε, εδώ ε, οι κοινωνίες μας όταν χρειάζονται υποχωρήσεις στην διέρεση των οικογενειακών, των ιδιωτικών υποχρεώσεων, ουσιαστικά αναγκάζουν τις γυναίκες να εξασφαλίσουν την, την διαφορά να καλύψουν μάλλον τη διαφορά και να αναλάβουν και τις περισσότερες ώρες ε, απλήρωτης κακώς πληρωμένης εργασίας. Άρα δεν υπάρχει ακόμα αρκετή συνείδηση στην κοινωνία για τις διαστάσεις του προβλήματος αυτού. Πρέπει να δούμε τη συλλογική ευθύνη για το ζήτημα αυτό, όπως ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που αγγίζουν την ηθική ε, διάσταση του πώς προσεγγίζει τέτοια θέματα η κοινωνία μας. Θα πρέπει οι γυναίκες να δούμε ότι έτσι εργάζονται και στην Ήπεθρο με 30% των γυναικών να καλύπτουν την αγροτική δραστηριότητα χωρίς όμως να πληρώνονται ε, με τον ίδιο τρόπο που πληρώνονται οι άντρες και σε άλλους τομείς. Γι' αυτό λοιπόν κυρία Επίτροπε χρειάζεται μια σφαιρική στρατηγική για να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα, τα έμφυλα στερεότυπα και ε, να αντιμετωπίσουμε αυτή τη πραγματικότητα ακόμη και στο σχολείο διότι με ε, στόχοι θα πρέπει να να αντιμετωπίσουν αυτήν την ανισότητα που οδηγεί και σε δομική βία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ολοκληρώνονται τι παρεμβάσει βάσει της διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΙ και τώρα ο λόγος στην Ελένα Ντάιλε, την Επιτρόπο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων για την προσήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό και την υποστήριξή του. Σας ευχαριστώ όλους ε, για τις ε, πολύ σωστές παρεμβάσεις σας απόψε. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί με βάση τα γεγονότα, τα δεδομένα και είναι γεγονός ότι οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο από τους άντρες. Είναι επίσης γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει δράση πάνω στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να κλείσω θυμίζοντάς σας ότι πέρα από δεσμευτικά μέτρα διαφάνειας ε, για ε, τις αμοιβέ υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν ε, στο οι γυναίκες ε, να μην μπορούν να αναπτύξουν πλήρως ε, τις ικανότητές τους και να μην αμείβονται παρκώς για αυτό που κάνουν. Η νέα μας στρατηγική λοιπόν για την ισότητα των δύο φύλων που που θα εφαρμοστεί θα ασχοληθεί και με άλλους τέτοιους παράγοντες όπως επισημάνθηκε στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ε, καταβάλουμε προσπάθειες λοιπόν ε, για να καταπολεμήσουμε την βία ει βάρο των γυναικών και την ε, επιγραμμική, διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και την παραμονή τους σε σχέσεις όπου υφίστανται βία. Υπάρχουν συνέπειες εάν δεν ε, λυθεί ικανοποιητικά το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Θα ήθελα να δω ισορροπία ανάμεσα στα δύο φύλλα και σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων, βελτιωμένη ισορροπία ανάμεσα στον επαγγελματικό και οικογενειακό βίο άνδρων και γυναικών, διότι αυτό είναι κάτι που επηρεάζει γενικά τη ζωή όλων μας και των οικογενειών μας. Θα ήθελα λοιπόν ε, ισότητα των δύο φύλων, και να λαμβάνεται υπόψη και αυτή η πτυχή ε, σε θέματα όπως είναι η αλλαγή του κλίματος ε, και η ψηφιοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή της οδηγίας ε, για την ισορροπία οικογενειακού και επαγγελματικού βίου στα κράτη-μέλη θα ε, προωθήσουμε τις ευέλικτες μορφές εργασίας ε, και την ε, χρήση του ιδιαίτερα από άντρες, πιο σωστό επιμερισμό των καθηκόντων φροντίδα σε κάτι που είναι απαραίτητο για να κλείσει το μισθολογικό χάσμα. Βλέπετε ότι όλα αυτά τα θέματα συνδέονται μεταξύ τους. Θέλουμε οι γυναίκες να αναπτύξουν πλήρως τις ικανότητές τους συμπεριλαμβανομένες ε, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών τους δυνατοτήτων. Το να ε, έχουν θέσεις χαμηλότερης αμοιβή ε, δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Οι κατευθυντήρες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Επιτροπή στόχο έχουν βελτίωση τη θέση των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Θα εργαστώ σκληρά, θα συνεργαστώ με τα κράτη-μέλη για να πετύχουμε πλειοψηφία για να λύσουμε το θέμα των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων. Βασίζομαι στην υποστήριξη του ε, Κοινοβουλίου. Ε, μπορούμε να ε, φροντίσουμε να νίκει στο παρελθόν το μισθολογικό χάσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε, και για την προσελευσή σας και για την ομιλία σας. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση για το σημείο αυτό. Η ψηφοφορία θα γίνει στην δεύτερη ολομέλεια του Ιανουαρίου, ε, το τέλος του μήνα. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης, που είναι η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με τίτλο «Προτεραιότητα στη στέγαση» ως μέτρο επίγουσας δράσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης των αστέγων στην Ευρώπη. Ε, χωρίς ε, περαιτέρω καθυστερήσεις, να ξεκινήσουμε. Θέλω να δώσω το λόγο στον ε, κύριο Σμιτ. Περιμένουμε να λάβει θέση για να μπορέσει να εκφωνήσει την ομιλία του. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οργάνωσε τούτη τη συζήτηση, διότι πρόκειται για μια συζήτηση η οποία αγγίζει ένα από τα μείζωνα προβλήματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο ε, ε, του κοινωνικού αποκλεισμού και της μιζέριας. Ο αριθμός των αστέγων διαρκώς αυξάνεται. Άλλωστε, αρκεί να περπατήσει κανείς ε, στις πόλεις μας για να το συνειδητοποιήσει αυτό. Ε, η, η αξιοπρεπή στέγαση ε, σε προσβάσιμη τιμή και κόστος είναι πραγματικά μία προϋπόθεση που σχεδόν αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Ε, αυτή τη στιγμή όμως αυτό το δικαίωμα δεν υπάρχει στις περισσότερες ε, ε, χώρες. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία αξιόπιστα όσον αφορά αυτό το πρόβλημα. Ωστόσο, έχουμε κάποια αριθμιστικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι ο αριθμός των αστέγων στις περισσότερες χώρες μέλη έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία υπολογίζουμε περίπου στα 3 εκατομμύρια τους ανθρώπους, τον, τον αριθμό των αστέγων στην ε, ε, Ευρώπη. Κάθε νύχτα περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι κοιμούνται στους δρόμους. Ε, πρόκειται για ένα καθημερινό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στις πόλεις μας και που βεβαίως μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Τα αίτια του προβλήματος είναι πολλαπλά και περίπλοκα. Ωστόσο είναι σαφές ότι οι παράμετροι της ε, αγοράς ε, ακινήτων έχουν συγκεκριμένη, ε, συγκεκριμένο αντίκτυπο σε αυτήν την μορφή κοινωνικού αποκλεισμού των αστέγων και που αφορά ακόμα περισσότερο ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσχερή θέση και μετανάστες. Η αύξηση των τιμών της στέγασης και η μείωση των διαθέσιμων, της διαθέσιμης κοινωνικής στέγης ε, α, αποτελεί ε, πηγή του προβλήματος. Κατά την έννοια αυτή, τα κοινωνικά διαμερίσματα, ε, καθώς επίσης και μια διαφοροποίηση της αγοράς θα μπορούσε να βοηθήσει τις οικογένειες. Είναι γεγονός ότι και πολλές οικογένειες χωρίς ε, να γίνουν άστεγοι υφίστανται ε, σε πολλές περιπτώσεις αυτήν την κακή πολιτική ε, όσον αφορά την στέγη και τις αστρονομικές τιμές των ακινήτων. χρειάζονται συγκεκριμένες επενδύσεις. Η Task Force σχετική με το θέμα αυτό το 2018 στην έκθεσή της ανέφερε ότι 55 δις ε, ευρώ θα χρειαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα όσον αφορά τη στέγαση ε, που αποτελεί συνήθως ε, ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών η, κοινωνική, το θέμα αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Χάρτα Δημολιωδών Δικαιωμάτων ρητά αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ως δικαίωμα το δικαίωμα στην αξιοπρεπή στέγη ως ε, ε, στοιχείο και παράμετρο αξιοπρεπούς ε, διαβίωσης ο, ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων αναφέρεται επίσης στο ίδιο γεγονός αναφέροντας ότι η ε, καταπολέμηση της ε, έλλειψης στέγης ε, καθώς αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα και επομένως και κοινωνικό δικαίωμα των πολιτών. Θα πρέπει να υπάρξει κοινωνική αντιμετώπιση μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή δημιουργεί ένα συνολικό πρόγραμμα σε τοπικό, εθνικό και ε, ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό ε, προς όφελος των πολιτών ε, και οπωσδήποτε στη διαδικασία αυτή η στέγη θα πρέπει να αναφέρεται με σαφή τρόπο. Η αρχή παριθμών 19 του κοινωνικού πυλώνα αναφέρεται ακριβώς στο ΠΔΠ μετά το 2020 η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της στέγης θα πρέπει δεν να συνδυαστεί με θεματικά πεδία τα οποία μπορούν να ε, υποστηριχθούν από το Κοινωνικό Ταμείο πλάσμα. Ε, και στο Invest ε, EU, καθώς επίσης και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία ε, προτείνεται να χρησιμοποιηθούν ακριβώς για το θέμα αυτό. Μέσω της χρηματοδότησης μεγάλου αριθμού κοινωνικών προγραμμάτων κοινωνικής υποδομής ε, καθώς επίσης και κοινωνικής στέγασης ε, μπορεί να δοθεί κάποια λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ε, θα, και προτίθεται να υποστηρίξει τις εθνικές κυβερνήσεις ή σε την διαμόρφωση εθνικών πολιτικών για την στέγαση έτσι ώστε να υπάρχει προσιτή και προσβάσιμη κοινωνική στέγαση και λειτουργική στέγαση για όλους τους πολίτες. Ε, πράγμα που αυτή τη στιγμή ε, δεν υπάρχει και άλλωστε ε, και η κοινωνική, ο ρυθμός των, της κοινωνικής είναι ανεπαρκής. Αυτός ο αγώνας εντάσσεται στο γενικότερο αγώνα καταπολέμησης της ένδυας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δουλέψει πάνω σε αυτό. Υπάρχει ένα καλό παράδειγμα με το οποίο αφορά την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της στέγασης μέσω του προγράμματος Housing First, όπου η επίγουσα ε, δράση αντιμετώπισης της ε, κατάστασης συνδυάζεται ε, με μεγαλύτερης διάρκειας δράσης. με τα εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, διάθεσή της ε, μπορεί να προχωρήσει και σε μια διαδικασία ανταλλαγής καλών πρακτικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης η υποστηρίζει ε, άμεσα την ΦΕΑΤΣΑ, αυτήν την ε, οργάνωση ε, που δρά για την καταπολέμηση το, της κατάστασης των αστέγων σε τοπικό επίπεδο και που έχει λάβει υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Επίτροπε και τώρα να ξεκινήσουμε με τις ε, ομιλίες των συναδέλφων. Πρώτα απ' όλα ο συνάδελφος Ράτκε για 1,5 λεπτό. Ja, Herr ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Ε, κάποιοι θα έλεγαν ότι γιατί ασχολείστε με το θέμα αυτό, δεν είναι καν αρμοδιότητά σας. Και εγώ θα απαντούσα ότι ναι, πιθανότατα, αλλά ένα θέμα που έχει να κάνει με την ραγδαία αυξάνουσα ε, κατάσταση όσον αφορά τους αστέγους στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συζητηθεί. Ε, το Κοινοβούλιο. Εάν κλείσουμε τα μάτια μας εμείς οι Ευρωβουλευτές σε ένα τέτοιο πρόβλημα, τότε ε, δεν ε, μας αξίζει να είμαστε μέλη του Κοινοβουλίου. Αν εξετάσουμε ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις ε, την κατάσταση, όπου από τη μία μεριά έχουμε ε, ραγδαία αύξηση των τιμών των ε, ενοικίων ε, και αύξηση της τιμής της ενέργειας. 400.000 νοικοκυριά έχουμε στη Γερμανία χωρίς ρεύμα. Πολύ περισσότερα τα νοικοκυριά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι μια εξέλιξη με την οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε θα πρέπει να εξετάσουμε και τις ε, ε, επιχειρηματικές πρακτικές όπως είναι το Airbnb που ε, προωθεί τον αθέμητο ανταγωνισμό και οδηγεί και σε όξυνση της κατάστασης όσον αφορά την στέγαση. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το θέμα των αστέγων και πέρα από αυτό θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ε, προωθήσουμε τη στέγαση, ε, τις ιδιόκτητες κατοικίες μάλιστα, για τις νέες οικογένειες. Θα πρέπει να εξετάσουμε ε, το πρόβλημα αυτό στην αρχή της αλυσίδας του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Άγνες Γιονγκέριους. Ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις κάτω χώρες 300.000 κατοικίες λείπουν. Ε, μία πόλη δηλαδή ε, στο μέγεθος ε, της πόλης μου της Ουτρέχτης που είναι η τέταρτη μεγαλύτερη στη χώρα. Υπάρχει λοιπόν έλλειψη οικονομικής κατοικίας και ενοικιαζόμενης και προσπόληση. Είναι πολύ λίγες ε, οι κατοικίες που είναι αρκετά οικονομικές και που βρίσκονται κοντά ε, στους χώρους εργασίας. Επίσης, όσον αφορά τις ενοικιαζόμενες ε, κατοικίες, είναι πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις. Τρεις φορές το ενίκιο θα πρέπει να βγάζει κανείς το μήνα και υπάρχει μακρύς κατάλογος αναμονής σε 10 χρόνια στη δική μου πόλη. Βλέπουμε λοιπόν διπλασιασμό των αστέγων τα τελευταία δέκα χρόνια στις κάτω χώρες. Καλώ όλους σας να υπογράψετε το ψήφισμα «Στέγαση για όλους». Έτσι, τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσουν εργασίε για να φροντίσουν να υπάρχει οικονομική στέγαση για όλου. Καλείται επίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει ευρωπαϊκό σχέδιο ε, για οικονομική στέγαση για όλου του Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ. Και τώρα για δύο λεπτά ο συνάδελφος Πισλάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω ρουμάνικα. Χίλιοι άνθρωποι είναι χωρίς ε, ε, στέγη ε, κάθε βράδυ στην πόλη μου. Η Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Οργανισμών των Αστέγων το δείχνουν αυτό. Επίσης, το 2017, σύμφωνα με την Eurostat, ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους που ζει σε συνθήκες φτώχειας ε, ζούσε σε στέγη αμφιβόλου ποιότητος ε, ή κοινωνική στέγη. Στην ε, Ρουμανία 9% των ευάλωτων ανθρώπων ε, ε, είναι οικογένειες με ε, παιδιά. Επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Μιλάμε για κατοικίες οι οποίες είναι ακατάλληλες για οικογένειες με παιδιά. Το πρόγραμμα Housing First, προτεραιότητα στη στέγαση, έχει και μπορεί να έχει πολύ καλά αποτελέσματα τα στοιχεία για τη Ρουμανία αλλά και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες ε, ε, δείχνουν ότι οι πολιτικές ε, έχουν μειωμένο αντίκτυπο. Στην Ρουμανία μάλιστα οι λύσεις που έχουν βρεθεί μέχρι τώρα δεν γίνονται αποδεκτές από όλους και επίσης τα διάφορα υπουργεία δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει το πρόγραμμα στην Ευρώπη, να βρεθούν ε, οι κατάλληλες κατοικίες και να δοθούν σταθερές λύσεις. Ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή και προτίθεμαι και έχω κάθε διάθεση να συμμετέχω, να προωθηθεί η πολιτική αυτή. Επίσης, αυτό το πρόγραμμα Housing First αποτελεί και, και πρέπει να αποτελέσει μέρος των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών στρατηγικών. Ε, θα πρέπει όλες οι χώρες ε, ε, να σέβονται, τις, να σέβονται κοινέ αρχές, θα πρέπει να έχουν κοινή προσέγγιση όσον αφορά την κοινωνική στέγη. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο λόγος του συναδέλφου Λάγκεντζιπεν για ένα λεπτό. Θα μιλήσω γερμανικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο καθένας χρειάζεται ένα σπίτι. Το που κατοικεί κανείς είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Ε, το να αρνούμαστε σε κάποιον τη στέγη σημαίνει ότι το αρνούμαστε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ένα βασικό δικαίωμα, το δικαίωμα να οργανώσει την αιστεία του και να ε, μπορεί να καθορίσει το μέλλον του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα βασικά δικαιώματα ε, να ε, είναι υποτίθεται αυτά που προστατεύει, θα πρέπει να αναλάβει δράση για την εξάλληψη του φαινομένου των αστέγων, τη έλλειψη στέγη δηλαδή, στο 2030. Θα πρέπει να σκεφτούμε αυτό που έκανε και η Φινλανδία με το Housing First, προτεραιότητα στη στέγαση και τη σχετική στρατηγική. Θα πρέπει να να κοιτάξουμε ότι η έλλειψη στέγης δεν είναι ποτέ σφάλμα του ίδιου του αστέγου. Στη Γερμανία υπάρχει δυνατότητα, ε, όπως και στην ε, Φινλανδία, να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη όμως να αναλάβουν δράση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να να απαιτήσει από τα εθνικά κράτη να καθορίσουν μια θετική στρατηγική. Χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο για να υπάρχουν όχι μόνο μέτρα πρόληψη, αλλά και συγκεκριμένοι στόχοι μέσω του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ώστε να γίνει κάτι και στην πράξη. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Ζαμέ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, Συνάδελφοι, πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και την επισφάλεια που ε, πλήττει όσους ε, δεν έχουν στέγη ή δεν έχουν κατάλληλη στέγη, τουλάχιστον στη Γαλλία είναι 12.000. Ε, θα πρέπει να κοιτάξουμε την επιδείνωση του φαινομένου αυτού σε πολλά κράτη-μέλη και να μας απασχολήσει. Οι πολιτικές λιτότητες εδώ και 10 χρόνια είναι από εσά αποφασισμένες. Οπότε δεν έχετε καμία νομιμοποίηση για να αντιμετωπίσετε τις παρεκτροπές του άκρα του φιλελευθερισμού και των ελεύθερων συναλλαγών. Ακόμα και ο κύριος Μακρό, ο οποίος ε, είναι πλήρως συμμορφωμένος με τις επιταγές σας, θα πρέπει να ε, βρει άλλο τρόπο για να ξεφύγουμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο και σίγουρα ε, ο μόνη διέξοδος φαίνεται να είναι εθνική. Είστε συνυπεύθυνοι για όλα αυτά και βλέπει ο Θεός τα ε, αίτια των δεινών αυτών ε, που πλήττουν τους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος Ραφάλσκα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, το πρόβλημα της έλλειψης στέγης είναι πολύ περίπλοκο και χρειάζεται μια κοινωνική πολιτική η οποία δεν, ε, δεν συγκεφαλείται μόνο στο, στα της κοινωνικής ασφάλειας. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα ε, πρόληψη για να αποφύγουμε το να προκύπτουν τέτοια φαινόμενα, τέτοιε καταστάσει. Και μετά πρέπει να υποστηρίζουμε όσου είναι άστεγοι, ώστε να μπορούν να ξεφύγουν από την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν. Μιλήσαμε για υπηρεσίε προ του ανθρώπου αυτού, για την ε, έκφραση ανθρωπιά. Σίγουρα αυτό το δέχομαι, αλλά πρέπει να χτυπήσουμε και τα γενεσιουργά αίτια τη ε, ε, έλλειψη στέγης, ε, οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακές συγκρούσεις ή ένα διαζύγιο μπορεί να είναι η πηγή του προβλήματος και πολλά παρόμοια. Μιλήσατε για την αύξηση του αριθμού αστέγων στην Ευρώπη, στην ε, Πολωνία. Πριν από λίγα χρόνια κάναμε σχετικές μελέτες και είδαμε ότι τα ποσοστά έχουν μειωθεί κατά 9%. Ε, πρέπει ε, να στηρίξουμε τον κόσμο για να επιστρέψει στην ε, εργασία. Ακόμα και η παροχή στέγης είναι σημαντική ε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως χωρίς κυβερνητική στήριξη, χωρίς τις κατάλληλες υποστηρικτικές πολιτικές, δεν θα ήταν εφικτό να υπάρξει ευθυνή στέγη και να προσφέρεται σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα για ένα λεπτό η συνάδελφος Λέιλα Σαϊμπή. Συνάδελφοι, 100.000 ε, άνθρωποι κοιμούνται στους δρόμους στην Ευρώπη κάθε βράδυ. Ε, επίσης, ε, είναι πολλοί αυτοί που έχουν ένα κεραμίδι από το κεφάλι τους, αλλά μπορεί να βρεθούν από τη μια στιγμή στην άλλη στο δρόμο. Ε, αυξάνονται η αξία των ε, κατοικιών, γι' αυτό η κοινωνική στέγαση θα ήταν μια λύση. Αλλά έχω και μια ερώτηση. Από τη μια, πώς η στέγη αναφέρεται ε, ε, στο σύνολο των βασικών δικαιωμάτων, ε, στη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και από την άλλη υπάρχουν κράτη-μέλη που επενδύουν στις κοινωνικές κατοικίες αλλά δέχονται κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί πλήττουν την ιερή αυτή αρχή της ελεύθερης αγοράς. Επίτροπε, αν τα λέτε σοβαρά αυτά που είπατε, αποδείξτε το και κάντε με τον κανόνα του 3% αυτό που λέτε για τις ε, κοινωνικές κατοικίες. Διότι για να μπορέσει κανείς να ξεφύγει από μια τέτοια κατάσταση, εφόσον έχει περιέλθει σε αυτή, πρέπει να ξέρει και πού θα κοιμηθεί πρώτα-πρώτα. Σας ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό, ο κύριος Παπαδάκης. Τα αμερικανόπνευστα προγράμματα Housing First που σχεδιάζεται ούτε καινούρια είναι, ούτε έλυσαν ποτέ κανένα πρόβλημα απευθύνονται σε ελάχιστους άστεγους και εξαθλιωμένους από τα εκατομμύρια σε όλη την ευρώπη που η ανεργία και οι τσακισμένοι μισθοί όσων δουλεύουν κάνουν πολυτέλεια την αξιοπρεπή στέγαση στις συμπληγάδες του airbnb και των πανάκριβων σπιτιών που ξεπερνούν και τους κόπους μιας ζωής η ευρωπαϊκή ένωση χύνει προκλητικά κροκοδίλια δάκρυα για τους αστέγους την ίδια ώρα που στην τέταρτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση για την ελλάδα εκθιάζει το διακηρυγμένο στόχο της νυν και πρώην κυβέρνησης για 120.000 πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών ως το 2021. Με αλλεπάλληλες κεφαλαιοποιήσεις, απαλλαγές κόκκινων δανείων, πρημοδοτούνται τράπεζες και φαντς με το λογαριασμό να πληρώνει ο λαός με απολύσεις τραπεζοϋπαλλήλων και απαγορεύσεις κινητοποιήσεων ενάντια σε πληστηριασμούς. απαιτούμε νομοθετική απαγόρευση πληστηριασμών λαϊκών κατοικιών και κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών μισθοδοσίας σύνταξης από το κράτος τράπεζες και funds. όπως έχει αποδειχθεί μόνο με κεντρικά σχεδιασμένη σοσιαλιστική οικονομία πάβει η στέγη να είναι εμπόρευμα και μπορεί η λαϊκή κατοικία να εξασφαλιστεί. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Παπαδάκη. Υπάρχει όμως γαλάζια κάρτα. Τη δέχεστε? Από τον συνάδελφο Χάτκε. Δέχεστε την γαλάζια κάρτα. Ε, Ωραία, 30 δευτερόλεπτα. Συνάδελφε, θα με ενδιέφερε να ρωτήσω το εξής. Εάν η κατάσταση ε, μπορούσε να εξηγηθεί τόσο εύκολα όσο κάνατε εσείς τώρα μόλις, τότε ρωτώ, μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς στις χώρες όπου δεν έχει λάβει αποφάσεις η Τρόικα, ε, τι εξοικονομήσεις έγιναν για να φτάσουμε στην κατάσταση αυτή, εάν ισχύουν όσα είπατε. Κύριε Παπαδάκη ένας λόγος παραπάνω σε αυτές τις χώρες όπως η ελλάδα που είναι ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση όλα αυτά τα ευχολόγια που ακούμε εδώ δήθεν και τα κλαψουρίσματα για τους αστέγους ένας λόγος παραπάνω η στάση της ευρωπαϊκής ένωσης που ακριβώς προωθώντας όλα αυτά τα αντεργατικά μέτρα τσάκισε ένα λαό και ταυτόχρονα τον οδήγησε σε πληστηριασμούς τους οποίους και ε, θέτει αριθμητικούς στόχους για 120.000 μέχρι το 2021 και προκαλεί και προωθεί μέχρι και διώξεις και απαγορεύσεις. άρα λοιπόν αυτή είναι η πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης και σε αυτές τις χώρες και συνολικά στις υπόλοιπες. Και τώρα η κυρία Φράνσεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Το θέμα των αστέγων είναι ένα θέμα που μας πονάει όλους ε, πολύ πάνω από 800.000 είναι τελικά οι άστεγοι αυτή τη στιγμή στην ε, Ευρώπη. Επίσης ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε αστέγους που έχουν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες στις διάφορες χώρες μέλη. Υπάρχουν όμως και κάποιες πρακτικές οι οποίες φαίνεται να λειτουργούν και αρκετοί αστεγοί μέσω των προγραμμάτων αυτών των διαφόρων έχουν βρει σταθερή στέγη. από την άλλη παιδιά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να καλυφθούν οι άνθρωποι αυτοί και να ξεπεράσουν και τα ψυχολογικά και άλλα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουν έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση και στην αγορά εργασίας. Επίσης ε, η εγγύηση για τα παιδιά ε, και τους ε, νέους θα φτάσει και θα ισχύσει και για τα παιδιά και νέους των αστέγων θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε πολυσχηδή προσέγγιση ε, και το πρόγραμμά μας να είναι φιλόδοξο. Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο έχει ε, πλέον ε, ο κύριος Πισάρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σε αυτές τις κρύες νύχτες και αυτή την κρύα νύχτα της δικής μας συζήτησης σήμερα, πραγματικά η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στους αστέγους. Με εξαίρεση τη Φιλανδία, σε όλα τα κράτη-μέλη επιδεινώνεται η κατάσταση. Γνωρίζω ότι η, η λύση μπορεί να είναι μόνο περίπλοκη. Ε, θα πρέπει όμω να βρούμε λύσει στον τομέα τη υγεία, τη κοινωνία, ακόμα και στο ψυχολογικό επίπεδο. Χρειάζεται μια ε, στατική σφαιρική και η λύση, η απόκριση που θα δώσουμε, πρέπει να ε, δοθεί κατεπηγόντω. Είναι πολλά τα προβλήματα που υπάρχουν και που πρέπει να απασχολήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εγγύηση για τα παιδιά, για του νέου, η καταπολέμηση τη φτώχεια, Όμω ε, πρέπει επιτέλου να περάσουμε στη φάση τη δράση. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα δράση για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο αυτό. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένε δράσει φιλόδοξε ε, ανά κράτο μέλο, ανά γεωγραφική περιοχή και ανά ε, συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε στην επίκαιρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν δικαίωμα σε στέγη είναι ένα από τα βαθύτερα κοινωνικά προβλήματα. Κύριε Επίτροπε, έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη. Θα αναλάβετε δράση για να επιληθεί το ζήτημα αυτό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η συνάδελφος Βερονίκα Τριγέλιο Νουάρα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω στα γαλλικά. Ε, η στέγη ε, είναι επίγουσα, ε, επίγον θέμα που αφορά την δημόσια υγεία. Ε, οι άνθρωποι που ζουν στο δρόμο ζουν κατά μέσο όρο 30 χρόνια λιγότερο από τους υπολείπους. Το να είναι κανείς άστεγος είναι, ε, είναι απόλυτα ευάλωτος όσον αφορά συμπεριφορές επικίνδυνες αλλά και προβλήματα υγείας που από αυτή την κατάσταση προκύπτουν. Όπως δείχνει και η πρόσφατη τη μελέτη του παρατηρητηρίου των γιατρών του κόσμου η κατάσταση των ανθρώπων αυτών είναι ιδιαίτερα τροτή. κυρίως όσον αφορά την υγεία και τα υγειονομικά ζητήματα. Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, ε, ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων θα πρέπει να συμπεριλάβει και τους αστέγους. Κανείς δεν πρέπει να μείνει απ' έξω, πολλό δε μάλλον που πρόκειται για θέμα υγείας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Τριγέλο Νουάρ και έχει τώρα το λόγο ο συνάδελφος Κιμ Βαν Σπάρεντακ για ένα λεπτό. Thank you. Η συνάδελφος Κιμ. Αυτή τη στιγμή ή το πρόβλημα της ε, στέγης σε όλη την Ευρώπη ε, προκύπτει με ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Ε, χρειάζεται να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα και συγκεκριμένες δράσεις. Το τελευταία δεκαετία δεν δείξαμε τη δέουσα προσοχή στο θέμα αυτό ε, της ε, κατοικίας ε, και μάλιστα οι πολλές πολιτικές λιτότητες που εφαρμόστηκαν σε διάφορες χώρες οπισθοδρόμησαν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Επίσης το θέμα της υψηλής τιμής της ενέργειας και της ακρίβειας της ζωής γενικότερα έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στο να χάσουν το σπίτι τους θα πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτον όλοι ότι δεν είναι δυνατόν να ποινικοποιείται το γεγονός ε, του ότι κάποιος είναι άστεγος. Επίσης ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και η εγγύηση για τα παιδιά και τους νέους έτσι ώστε να σπάσει ο κύκλος ε, της έλλειψης ε, κατοικίας. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε οι άνθρωποι αυτοί να μην βοηθηθούν έτσι ώστε να επιβιώνουν, αλλά να σπάσει αυτός ο κύκλος και να αρχίζουν να ζουν πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ. Τον ε, ρόλο έχει ο Σνέφος Γκίντο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είμαι ευγνώμων που από τη στιγμή που δηλώθηκε ότι θα συζητηθεί το θέμα ε, των ε, αστέγων, επιτέλους ε, συζητιέται εδώ πέρα. Εδώ και έξι μήνες που είμαι στο Κοινοβούλιο, βλέπω αστέγους και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, ενώ στο παρελθόν έβλεπα και στην πατρίδα μου ξέρετε τι γίνεται κάτω από τις γέφυρες του ε, Στρασβούργου. Επικρατεί ε, ανάγκη και στέρηση. Τρία εκατομμύρια Ευρωπαίων ε, είναι άστεγοι. Είναι ο λοιμός του 21 ου αιώνα και αγνοούμε το πρόβλημα αυτό ε, τους ανθρώπους αυτούς δεν τους βλέπουμε καν πια. Δεν έχουμε καμία λύση, ε, ούτε καν ε, έχουμε ε, ξεκινήσει να ασχολούμαστε με το πρόβλημα. Πρέπει επιτέλους να το λύσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η συνάδελφος Μπεάτα Σίτλο για ένα λεπτό. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Τώρα που συζητάμε ένα τόσο σημαντικό θέμα, ε, τους αστέγους δηλαδή, Πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει ε, να το θεωρήσουμε σύμβολο προβλήματος ε, που δεν έχει λυθεί και που θα πρέπει όλοι μας ε, να ασχολούμαστε με αυτό. Όπως είπε και ο συνάδελφος, βλέπουμε αστέγους ακόμα και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Η μεταναστευτική κρίση έχει οξύνει το πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε να παραμένουμε άπραγοι, πρέπει να αναλάβουμε δράση. Και θα ήθελα να αναφέρω άλλη μια διάσταση του προβλήματος των αστέγων ε, που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Η Ευρώπη γυράσκει, διαλύονται οι οικογενειακοί δεσμοί, ε, δεν ε, υπάρχει επαρκής φροντίδα για τους ηλικιωμένους, κάτι που συχνά αφήνει τους γέρους σε προβληματική κατάσταση τους κάνουν έξωση από τα σπίτια τους, δεν έχουν που να μείνουν. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε το θέμα και των, αστε... των ηλικιωμένων αστέγων που χρειάζονται ιδιαίτερα τη φροντίδα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Ζωζέ Μάου, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ε, πρόγραμμα για την πρώτη κατοικία έδωσε αποτελέσματα, διότι πολλοί πολίτες ε, έλυσαν το πρόβλημα της στέγασης και άλλα προβλήματα φτώχεια και κοινωνικού αποκλεισμού λύθηκαν με αυτά. Στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα, εφαρμόζεται μια πρώτη φάση του προγράμματο για την πρώτη κατοικία. Ε, είναι ε, χωρί καμία μάλλον στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει αυτή την πρώτη κατοικία, τι θα γίνει για το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τόσο πολύ αγωνίστηκε για την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματο, για την ε, κτηματομεσητική αγορά, με τι αρχέ τη λιτότητα που οδήγησαν σε πλήρη κατάρρευση των αγοραστική δύναμη των ε, Ευρωπαίων πολιτών, με όσα συνέβησαν σε όλη την Ευρώπη, τι θα κάνετε επιτέλου, έχετε κάτι ουσιαστικό να μα ε, υποβάλλετε για να υποστηρίξετε αυτά τα προγράμματα που τόσο πολύ έπληξαν του Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστούμε. Η ε, συνάδελφος Κλέρ Φόξ για ένα λεπτό. Πριν πολλά χρόνια εργαζόμουν σε καταφύγιο για στέγους ε, στην ε, Αγγλία και είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Έχω όμως και κάποιες ανησυχίες. Φοβάμαι ότι υπάρχει ε, πρόβλημα εάν έχουμε μία υπερεθνική λύση που θα αγνοεί τις τοπικές συνθήκες και τις λύσεις που μπορούν να βρεθούν. Οι αιτίες που οδηγούν τους ανθρώπους στην απόλυτη σχόλια ε, δεν είναι ήδη παντού. Σε κάποιες χώρες το πρόβλημα ε, ε, ήταν αποτέλεσμα πολιτικών λιτότητας που επιβλήθηκαν σε χώρες της Ευρωζώνης από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει οδηγήσει στην ανεργία και σε αστέγους. Αλλά γλυμνάζουσες οικονομίες σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης έχει οδηγήσει ανθρώπους να αναζητήσουν καλύτερη ζωή αλλού ε, και τελικά καταλήγουν να είναι άστεγοι. Φαίνεται ότι οι άστεγοι ε, από την υπηρετική Ευρώπη ε, αντιπροσωπεύουν το 1 τρίτο των αστέγων στους δρόμους του Λονδίνου ένας άστεγος Πολωνός ε, ε, επί πέντε χρόνια ε, στην Αγγλία που προχώταν από την Πολωνία είπε ότι τίποτα δεν μου κάνει εμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Και τώρα η Αντιπρόεδρος Μακίνες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Τον Σεπτέμβριο του 2018 προβλέψαμε μια ε, αρχή για την Ιρλανδία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των αστέγων, αυτών που βλέπουμε στην πρωτεύουσά μας του Δουβλίνου συγκεκριμένα. Υπήρξε μια μικρή, ε, ένα μικρό αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να προβλεφθούν μέτρα για όλες τις χώρες. Έχω εργαστεί στα Midlands της Αγγλίας, όπου προβλέφθηκε στέγη σε κοινωνικά κτίρια για ανθρώπους που χρειάζονταν υποστήριξη. Και έγινε αυτό και πραγματικά τους προσφέρθηκε κάτι. Όμως, Επίτροπε, πρέπει να γίνει μια ευρύτερη, ευρύτερη συζήτηση από το Housing First προτεραιότητα τη στέγαση, διότι δηλαδή στη χώρα μου, με τι τιμέ που έχουν τα ακίνητα, ε, για κάποιε οικογένειε γίνεται αρκετά δύσκολο ε, να αντιμετωπίσουν τα προστοζήν και να καλύψουν το βιωτικό του επίπεδο ε, με τον περιορισμό των εξόδων του, με τι εμπειρίε των εσόδων του. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τα προβλήματα φτώχεια σε όλη την Ευρώπη και θα πρέπει να δούμε τι υποσχέσει που είχαμε δώσει για να βρούμε κοινέ λύσει. Πρέπει να υπάρχουν χαμηλότερε τιμέ. Χρειάζονται επίση δεξιότητε και τεχνικοί ε, χτίστε με δεξιότητε που να χτίσουν τα κατάλληλα σπίτια. Τα γνωρίζουμε εδώ. Ε, οι τιμέ των κτηρίων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υπάρχουν πολλά ελπιδοφόρα μηνύματα όμω εκτό κοινοβουλίου, στι Βρυξέλλε. Βλέπουμε πω οι άστεγοι κυκλοφορούν έξω από τα κτίρια μα. Και το βλέπουμε εδώ και στο Στρασβούργο. Είναι ένα πρόβλημα που ε, κρατάει χρόνια. Ε, πρέπει λοιπόν κάτι να σκεφτούμε. Ευχαριστούμε και τώρα ο λόγος για την ε, συνάδελφο Στρέλα Ντουρά Φεράντης. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Το να είναι κανείς άστεγος δεν σημαίνει απλώς ότι δεν έχει σωστή ε, αλλά σημαίνει και προβλήματα υγείας, προβλήματα κοινωνικά, προβλήματα ακόμα και για την ε, ίδια την ασφάλειά του. Το Housing First είναι μια στρατηγική ε, η οποία συνδυάζει την ε, κατοικία μαζί με ταυτόχρονη παρακολούθηση κοινωνική και υγείας. Θα πρέπει σε όλα τα κράτη-μέλη η Κομισιόν να βοηθήσει για να εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο με κατάλληλη χρηματοδότηση και βεβαίως στο, στα πλαίσια του βιώσιμου βιώσιμου εξαμήνου να προσθεθεί και αυτό το θέμα των αστέγων. Κύριε Επίτροπε, η Κομισιόν θα πρέπει ε, πρώτα απ' όλα να ε, ε, προτείνει σειρά συστημάτων έτσι ώστε να εκριζωθεί αυτό το φαινόμενο, να μην υπάρχουν πλέον άστεγοι. Θα πρέπει Επίσης να βοηθηθούν οι κινητικοί εργαζόμενοι εντός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε οι ε, μετακινούμενοι εργαζόμενοι και οι αποσπασμένοι να έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και να μην τα χάνουν λόγω της μετακίνησης. Ευχαριστώ. Και τώρα ο συνάδελφος Φρανσίσκου Γκεγαϊρου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε Επίτροπε. Υπολογίζουμε ότι υπάρχουν 700.000 άστεγοι περίπου, ακόμη και οικογένειες όμως που ζουν σε κατάσταση ε, ε, ε, σε ευπαθείς κατοικίες σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν ε, βαθιέ ανισότητε μεταξύ των χωρών. Γι' αυτό για του αστέγου ε, θα πρέπει να ε, καταλάβουμε ότι υπάρχουν λύσει που θα μπορούσαν να είναι και χειροπιαστέ. Ξέρουμε το πρόγραμμα τη Φιλανδία στο Housing First. Θα πρέπει λοιπόν την αξιοπρεπή στέγη που προβλέπει το πρόγραμμα αυτό να την πάρουμε ω προτεραιότητα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και κοινωνικοί στόχοι, κοινωνικέ πολιτικέ που απαιτούν συντονισμό των πολιτικών υγεία με τι πολιτικέ απασχόληση και τα κοινωνικά. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε την εκρίζωση τη ακραία φτώχεια. Μια από τι προτεραιότητε που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρξει και μια βιώσιμη ανάπτυξη και επιτεύξη των στόχων αυτών. Ε, ευχόμαστε λοιπόν να κάνετε την πόρτα για την επιτεύξη των στόχων αυτών και θα πρέπει να ασχοληθούμε και με ε, housing first προγράμματα σε επίπεδο κάθε χώρα. Να υπάρξουν εθνικά προγράμματα με την προτεραιότητα στην στέγαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ε, προχωρήσει κατεπηγόντω με ένα μηχανισμό που να προλαμβάνει την ε, δημιουργία τέτοιων καταστάσεων που οδηγούν του πολίτε στου δρόμου. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο λόγο στη Σίλβια Σαρντόνε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Και βεβαίω όλοι είμαστε υπέρ προγραμμάτων που βοηθούν ε, είτε τους ε, αστέγους να του βοηθήσουν να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω το κεφάλι τους, ε, να τους εντάξουν στην κοινωνία κλπ. Αλλά μια και είμαστε εδώ θα πρέπει λίγο να δούμε λογικά και να αντιμετωπίσουμε τα αίτια. Γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποιες ευθύνες γιατί ε, ναι, τελικά έχει αυξηθεί ο αριθμός των αστέγων που ε, ξεχύνονται στους ε, δρόμους μας. νομίζω ότι αυτό είναι και αποτέλεσμα αυτής της υποδοχής χωρίς όρια του ότι ανοίγουμε τις πύλες μας και τις πόρτες μας προς όλους και θέλουμε να δεχτούμε όλους τους μετανάστες στις χώρες μας. Ή χωρίς όριο και φρένο μετανάστευση μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα προβλήματα στις πόλεις μας, στους δρόμους μας. Ε, γι' αυτό λοιπόν ας ε, κάνουμε λιγότερη ρητορική και περισσότερη αυτοκριτική. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον συνάδελφό μας Κωνσταντίνο Αρβανίτη. Ένα λεπτό. Καλησπέρα σας. Θα μιλήσω ελληνικά. Είμαι από, την, από τον ΣΥΡΙΖΑ και την QNGL η απώλεια της κατοικίας είναι η πρώτη συνέπεια της πολιτικής της φτωχοποίησης κύριε επίτροπε κύριε πρόεδρε. είναι πολιτική συνέπεια δεν είναι φυσική δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Και ειδικά στι χώρε του Νότου η στέγη ήταν το τελευταίο καταφύγιο στη διολίσθηση προ την απόλυτη φτώχεια. Επί Πρωθυπουργία Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάδα η πρώτη κατοικία προστατεύθηκε με νύχια και με δόντια. Και σήμερα ο Υπουργό Ανάπτυξη τη νέα κυβέρνηση δεξιά δήλωσε ότι από 30 Απριλίου μπαίνει πλαίσιο απόλυτη ε, μη προστασίας της πρώτης κατοικίας δηλαδή σχέδιο τέτοιο δεν θα υπάρξει. με βάση τους στόχους που έχει θέσει ο οηε για βιώσιμη ανάπτυξη και το πρόγραμμα της κυρίας φον για άμεση εφαρμογή της 19ης αρχής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ρωτώ πώς θα διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των αδύναμων στα προγράμματα στέγης. δεύτερον ζητώ την απαγόρευση των πληστηριασμών πρώτη κατοικία. και ρωτώ πάλι και πιστεύω ότι πρέπει η ενίσχυση της υπάρχουσας στέγασης να είναι δικαίωμα καθολικό δικαίωμα διασφαλιζόμενο πρωτίστως από την ευρώπη δικαίωμα επανένταξης στην κοινωνία. και τονίζουμε όχι χρηματοδότηση κατοικιών σε ειδικέ περιοχές όχι σε γκέτο αλλά μέσα στο βασικό κοινωνικό ιστό. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η Ντανιέλα Ροντινέλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, η καταπολέμηση της ε, ένδυας σε οποιαδήποτε μορφή ε, αποτελεί πλέον προτεραιότητα και πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Ωστόσο εμείς από την πλευρά των πέντε αστέρων πιστεύουμε ότι και αυτή η προτεραιότητα μπορεί να θρηματιστεί μέσα σε αυτή τη σκόνη και τη διασπάθηση των ε, προσπαθειών. Αναφέρεται βεβαίως ότι θα, και αναφέρεται σαφώς και τις προθέσεις της Νέας Επιτροπής, ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί αυτό και να υπάρχει κοινωνική ε, μέρημνα για τους ανθρώπους. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι ε, μονάχα εάν καταφέρουμε να μαζέψουμε δυνάμεις και χρηματοδοτήσεις θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της φτώχειας. Μας το ζητούν, ε, κύριε Επίτροπε, οι πολίτες μας τεπιτάσεως μάλιστα. Ε, ε, θέλουμε και ζητούν και εκείνη αξιοπρέπεια και αξιοπρεπή στέγη για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Σέντρο Τόμσκα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Πρέπει να πω ότι η Ευρώπη από κοινωνικής πλευράς αποτελεί πρότυπο για το υπόλοιπο του κόσμου. Ε, λαμβάνουμε υπόψη μας ε, ε, μειονοτικές ομάδες. Είμαστε από τους μεγαλύτερους χορηγούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τους ανθρώπους σε μειονεκτική θέση να έχουν αξιοπρεπή ζωή, δηλαδή να έχουν στέγη πάνω από το κεφάλι τους. αυτό αποτελεί τη βάση. Κάποιοι δεν έχουν τα μέσα για να έχουν κατάλληλη στέγη και θα πρέπει να τους φροντίσουμε. είναι οι άνθρωποι τους οποίους πέταξαν στο περιθώριο η ζωή. Και θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να βοηθήσει τους αστέγους του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να ανταλλάξουμε τις καλές πρακτικές μας. Εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να ε, ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν τον καλύτερο δρόμο για να λύσουν ε, το πρόβλημα αυτό. Ταυτόχρονα όσοι λαμβάνουν τέτοια κοινωνική βοήθεια θα πρέπει ε, να την ε, λάβουν με υπεύθυνο τρόπο. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον Επίτροπο Μίλαν Μπριγκλέτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε κάθε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να ε, διασφαλίσουμε ε, το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Η στέγη συχνά αποτελεί πρόκληση για του ανθρώπου. Τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει να εφαρμόσει μέτρα για την εξάλληψη του προβλήματος των αστέγων και άλλα μέσα δεσμεύουν ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη τη, ε, όπως είναι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, και ο κοινωνικό Πυλώνα. Οι άστεγοι αυξάνονται. Μόνο η Φιλανδία έχει καταφέρει να περιορίσει τον αριθμό τους και αυτό μας αναγκάζει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα προτεραιότητα στη στέγη θα πρέπει να παρέχουμε αξιοπρεπή στέγαση σε όλους. Ευχαριστούμε και τώρα ο λόγος στην συνάδελφο Ντελή για ένα λεπτό. Συνάδελφοί μου, κύριε Επίτροπε, πριν από εννέα χρόνια κοίταξα να περάσει η πρώτη στρατηγική για την προστασία των αστέγων. Ήμουν εισηγήτρια για την κοινωνική πολιτική και κάθε χρόνο κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Και ξέρετε κάτι, οι κυβερνήσεις κοιμούνται τον ύπνο των δικαίων. Ε, πού είναι η υπεύθυνοι, πού είναι η ανάληψη δράσης ε, τη στιγμή που έπρεπε να αναλυφθεί. Ε, αύξηση κατά 70% σε 10 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε μέρα ε, πεθαίνουν ένας ε, στους τρεις στην Γαλλία, 59% στην Αγγλία. Και λέτε ότι δεν έχουμε αριθμητικά στοιχεία. 11 εκατομμύρια άνθρωποι δεν ζουν σε εξωπρεπή κατοικία. Είναι σκανδαλώδες. 11 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άντρε, γυναίκε, παιδιά που υποφέρουν. Υποφέρουν στο... και μάλιστα σωματικά. Και μου λέτε ότι θα πρέπει να υπάρξει πολιτική υποδοχή. Η πολιτική τη υποδοχή πρέπει να οργανωθεί από τα κράτη-μέλη. Και όντω κοστίζει πολύ, μέχρι τώρα είναι αποτελεσματική και δεν κάνει τίποτα. Δεν έχουμε πλέον χρόνο για, ε, για προσωρινές λύσεις. Χρειάζεται να ξυπνήσουμε συνάδελφοι, να δείξουμε κάποια στιγμή ανθρωπιά, να ξυπνήσουμε για να βοηθήσουμε τους πιο αδύναμους. Ήρθε η στιγμή κύριε Επιτροπέ να πείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει τις ευθύνες της, θα καλέσει τα κράτη-μέλη αντί να ευνοούν ε, μόνο τις εταιρείε με φορολογικές εκτόσεις να κάνουν κάτι για την κοινωνική στέγαση και κατοικία και ολοκληρώνω. Θα πρέπει να κινητοποιούμαστε όχι μόνο για τις τράπεζες. Επιτέλους, καλό θα ήταν να κουνηθείτε και λιγάκι ε, μπροστά στην φτώχεια και την δυστυχία. Δεν μπορεί να διακυβερνάτε η Ευρώπη μέσω της αδιαφορίας. Και τώρα η συνάδελφος Αντρουέ για ένα λεπτό. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που κλαίνε για τις συνέπειες των αιτίων που προκάλεσαν. Ε, αν θέλετε να, να βελτιωθεί η κατάσταση των 700.000 αστέγων στην ε, Ευρωπαϊκή μας Ένωση, πρέπει να αλλάξει τα μέσο λογισμικό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δείτε ε, ε πώ θα πάψουν να συγκεντρώνονται οι υπηρεσίε και οι θέσει εργασία σε μεγαλοπόλει που ε, έχουν μόνο μπετόν και τεράστιε τιμέ και αναγκάζουν τον κόσμο να παίρνει τα μέσα μεταφορά για να φτάσει ω εκεί. Μετά να βρούμε ένα τόπο κατοικία, ενδιαιτήματα για τι οικογένειε που είναι φυσικό τόπο κατοικία με κατάλληλου δημόσιου χώρου και αξιοπρεπεί συνθήκε. Και να σταματήσετε να ε, επιβαρύνετε τη θέση των αστέγων ε, ει βάρο και μάλλον η προς όφελος των ε, ε, μεταναστευόντων και των, των μεταναστών και των προσφύγων. Βλέπουμε ότι τα δύο φαινόμενα είναι αλληλένδετα. Μέσα σε 10 χρόνια αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμό των αστέγων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσει ένα τεράστιο επικοινωνιακό πρόγραμμα για το θέμα αυτό, χωρί να πάψει τη δράση τη, για να πάψει να πλήττεται ο καθένα από το θέμα αυτό, κυρίω οι πιο φτωχοί. Ευχαριστούμε πολύ ο συνάδελφός μας Κυμπουρόπουλος. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, υπάρχουν διάφορες αιτίε που κάποιος θα βρεθεί στον δρόμο. Η αποτυχημένη παιδεία, η ελλειπής ενδοοικογενειακή κατανόηση διακρίσεις, η ενδοοικογενειακή βία, οι εξαρτήσεις, η ξαφνική ανεργία και ένα θέμα υγείας. Οι μακροπρόθεσμες λύσεις βρίσκονται πάλι στην παιδεία και την οικονομία. Επειδή όμω η ανάγκη είναι άμεση, θέλω να αναφερθώ και εγώ στις καλές πρακτικές της Φιλανδίας και του προγράμματος Housing First. Χρειαζόμαστε φιλόδοξους στόχους δεκαετίας. Μια προσφερόμενη κατοικία για λίγο, με κοινωνικούς λειτουργούς και ευκαιρίες εργασίας αποτελούν ένα καλό πλαίσιο επανένταξης. Ευκαιρία για εργασία. Αυτό θέλουν οι άνθρωποι, για να μπορέσουν να σταθούν και να δουν τον ήλιο αυτοί οι συνάνθρωποι μας δεν είχαν την τύχη να έχουν ανθρώπους γύρω τους να τους στηρίξουν στη δυσκολία. Ας γίνουμε εμείς οι άνθρωποι τους. Ας φτιάξουμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης και υποστήριξης, καθώς πρώτα απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Ας το δείχνουμε στις δυσκολίες και όχι μόνο τα Χριστούγεννα. Σας ευχαριστώ. Muito obrigado. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Τσίμνιοκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από το 2006 έως το 2015 ανοίξαμε τα σύνορα και στην Γερμανία είχαμε ένα τέταρτο το 250.000 ανθρώπους που έφτασαν ε, στη χώρα και βρέθηκαν άστεγοι. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε να λέμε το τι συνέβη και να αντιμετωπίσουμε το 1 εκατομμύριο ε, αστέγων που υπάρχουν στη Γερμανία. Έχουμε ε, ανεπίσημες μόνο στρατηγικές ως τώρα. Είναι πολλά τα παιδιά, οι γυναίκες, οι νέοι και ολόκληρο ολόκληρε οικογένειε που αναγκάζονται να ζήσουν στι οικογένειε. Την γενέτειρά μου, την, το Μόναχο, βλέπω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το 2015 περίπου 5.000 άνθρωποι βρέθηκαν στο γετό. Σήμερα έχουμε 10.000 διπλασιασμό. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει μια προσιτή τιμή στην στέγη, δεν υπάρχουν προσιτέ τιμέ στι και κατάλληλε θέσει εργασία. Βλέπουμε ε, να είναι ανεξέλεγκτη η μετανάστευση και να πλήττεται και η αγορά κινήτων. Ε, δεν υπάρχει πλέον κανένα σύστημα στην προσφορά στέγης ε, στο Μόναχο. Οι τιμές φτάνουν τις 10.000 ε, στο επιδόματα που προσφέρονται σε μετανάστες και τις οικογένειές τους. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τους ανθρώπους που ζουν στους δρόμους. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει επιτέλους τη δουλειά της, να κλείσει τα εξωτερικά σύνορα, προτού έχουμε κοινωνική δυσφορία και διαδηλώσεις στους δρόμους. Ευχαριστούμε πολύ. Είπα δεν θα δεχτώ γαλάζιες κάρτες, επειδή έχει προχωρήσει πολύ η ώρα. Και θα επιτρέψω μόνο την κανονική διεξαγωγή της συζήτησης ε, με τον κύριο από επόμενα αγορητέ, αλλά δεν βρίσκεται εδώ, οπότε περνάμε απευθεία στη διαδικασία Κατσδιάη. Στην, ε, στα πλαίσια τη διαδικασία Κατσδιάη θα δώσω το λόγο μόνο σε έναν ευρωβουλευτή από κάθε πολιτική ομάδα, επειδή ακριβώ έχει περάσει η ώρα, και θα ξεκινήσω από τον συνάδελφο Πόλκακ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο πρέπει να πω ότι το πρόβλημα της διαθεσιμότητας ε, των κατοικιών είναι πραγματικά πάρα πολύ ε, μεγάλο και μάλιστα δυσχεραίνει η κατάσταση μέρα με την ημέρα. Η προσφορά σπιτιών ε, είναι πάρα πολύ μικρή και καθόλου προσιτή. Φαίνεται λες και η αλληλεγγύη η ευρωπαϊκή σταμάτησε ε, σε αυτόν τον ε, τομέα. Είτε πρόκειται για την Βερολίνο, για, τον για το Μόναχο, για την Πράγα παντού. Ε, η πρόσβαση ε, σε καλή στέγαση είτε ε, στους νέους είτε σε ανθρώπους με χαμηλότερο εισόδημα γίνεται όλο και πιο δύσχερης. Επομένως θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στην αγορά εργασίας και την αγορά των ακινήτων. Και βεβαίως δεν μπορεί να ασχοληθούν μονάχα η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι κεντρικές κυβερνήσεις με το θέμα αυτό, αλλά περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις επίσης επίσης θα πρέπει να ασχοληθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό. John Howard. Uh, Mr. President, you'll have to bear with Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ ε, για την κατανόησή σας. Ε, έχω το λαιμό μου, θα πρέπει λοιπόν να μιλήσω ε, σιγανά και αργά. Υπάρχουν διαφορές αλλά και ομοιότητες ανάμεσα στις Βρυξέλλες και το Λονδίνο ενώ είναι και οι δύο πλούσιες ε, πόλεις, ε, βλέπουμε ε, βουλευτές και ευρωβουλευτές να περνούν πάνω από τους αστέγους. Αυτό αποτελεί σημαντική αποτυχία της δημόσιας πολιτικής. Δεν είναι πρόβλημα μετανάστευσης, είναι αποτυχία ε, στην ε, επένδυση στη στέγη. Αντιπροσωπεύω μια από τις πλουσιότερες περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα νοτιοανατολικά της Αγγλίας ε, και δεν θα έλεγα ποτέ σε κάποιον ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί σε εσά. Αν συμβεί σε εσά ή στο γιο σα, την κόρη σα, το γονιό σα, θέλετε να του αντιμετωπίσουν ως εγκληματίες, ως ναρκωμανείς. Το δικαίωμα στη στέγη θα έπρεπε να είναι δικαίωμα κάθε πολίτη αλλά βλέπουμε αστέγους παντού. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη σωστή προσέγγιση. Θα ήθελα λοιπόν η οθέτηση ενός πυλώνα δικαιωμάτων για τους αστέγους. Εάν δεν χτίσουμε σπίτια θα ε, έχουμε άστεγους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο συνάδελφος Σιέραν Κούφε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην Ιρλανδία έχουμε 4.000 παιδιά που δεν έχουν σπίτι. Η έλλειψη στέγης πλήττει γυναίκες, παιδιά και νέους, ε, καθώς και μετανάστες. Δυστυχώς δεν πιστεύω ότι ο Ιρλανδός υπουργό ε, στέγασης ε, για τους μετανάστες καταλαβαίνει το κατεπήγον του προβλήματος και μπορεί να αντιμετωπίσει την έκταση του φαινομένου στο Δουβλίνο, την Ιρλανδία και σε μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη. Μιλήσαμε προηγουμένως ε, για τα ποσοστά που υποτίθεται ότι είναι υπήρξε μείωση στα ποσοστά των αστέγων. Και όμω στην Ιρλανδία είχαμε διπλασιασμό ε, κυρίω μεταξύ των γυναικών και διπλασιασμό μεταξύ των παιδιών. Ε, ε, στην Ιρλανδία και μόνο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να πάνε απλώ σε ένα κέντρο υποδοχή, σε μια προσωρινή στέγη. Πρέπει να ασχοληθούμε με την οικοδόμηση κτηρίων, όπω έκαναν η Φινλανδία ή μπορεί να κάνουν η Αυστρία. Θα πρέπει να δούμε ότι το πρόγραμμα αυτό, το Housing First, δηλαδή η προσφορά ενό κεραμιδιού πάνω από το κεφάλι του κόσμου, είναι το μόνο που φέρνει αποτέλεσμα. Θέλω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει τη δουλειά τη με μια διάσκεψη για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αστέγων, για να χτίσουν σπίτια και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώ και η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα να ασχοληθούν με την ε, καταπολέμηση του προβλήματος αυτού. Δεν πρέπει να το ζούμε αυτό τον 21ο αιώνα. Ευχαριστούμε. Τελευταία παρέμβαση στη διαδικασία Κατσιάη Σάντρα Περέιρα. Για ένα λεπτό. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των αστέγων αυξήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με την, κοινωνική, με την υποβάθμιση των κοινωνικών συνθήκων. Έχει να κάνει με την αγορά εργασία, την ενέργεια, ε, την ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών, τον τομέα της υγείας. Η προσφορά στέγη σε διάφορα κράτη-μέλη δεν έχει να κάνει με την μείωση των εισόδημάτων και ε, πολλές φορές οι κάτοικοι ε, πρέπει να, σπατα... ξοδέψουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους ε, για την κάλυψη των ε, δαπανών στέγασης. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε, ε, να δούμε αυτά που έχουν ήδη συμβεί σε χώρε όπω η Πορτογαλία, η Δημοκρατία τη Πορτογαλία. Δεν μπορούμε να έχουμε το φαινόμενο των αστέγων χωρί μια κρατική πολιτική που θα αντιμετωπίσει την αγορά, τα όσα συμβαίνουν στην αγορά κινήτων. Μια, αγορά, μια πολιτική απασχόληση. Κατεπίγουσα καταπολέμηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει το δικαίωμα στην εργασία, οι συνθήκε αξιοπρεπού κατοικία και στέγαση να ε, συνάδουν με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Ευχαριστούμε και τώρα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας ο Επίτροπος Νίκολα Σμιτ. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, η συζήτηση αυτή δείχνει σαφώς ότι το πρόβλημα των αστέγων υπάρχει στο νότο όπως και στο βορρά, στην Ανατολή όπως και στη Δύση. Υπάρχει σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Δείχνει λοιπόν ότι είναι ένα πρόβλημα τοπικό, αλλά ταυτόχρονα και ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό. Και δεν είναι δυνατόν να ξεφύγουμε, να αποστρέψουμε το βλέμμα από το πρόβλημα αυτό λέγοντας ότι αυτό δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι είναι θέμα των τοπικών και εθνικών αρχών. Μας προβληματίζει το θέμα αυτό πολύ και μετά από την συζήτηση που είχαμε εδώ, για ένα λόγο παραπάνω θέλουμε να δεσμευτούμε. Τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρατε είναι πολύ εντυπωσιακά. Ε, και πρέπει και οι πόροι που θα έχουμε να είναι ε, ε, αρκετά υψηλοί και να μπορούν να κινητοποιηθούν γρήγορα. Βεβαίως το ζήτημα αφορά κυρίως την προσφορά στέγης, γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη όσον αφορά την προσφορά. Ναι, και θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα ότι ε, η αγορά κινήτων έχει γίνει μια αγορά κερδοσκοπική και ε, ε, βεβαίως στις πόλεις μας, ε, στις χώρες μας ε, η προσφορά έχει και την αντίστοιχη ζήτηση και ακολουθεί την ζήτηση. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα παράπλευρα ζητήματα, όπως ας πούμε η εργασία. Εάν δεν έχει κανείς στέγη, δεν μπορεί να έχει εργασία. Εάν δεν έχει κανείς σταθερή στέγη, τότε θα έχει ε, ε, ε, προβλήματα υγείας. Και όσο περισσότερο μένει κανείς στο δρόμο, τόσο τα προβλήματά του διευρύνονται, πληθαίνουν. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια πολιτική η οποία ναι θα χτυπήσει κατά πρώτο λόγο την ε, στέγη και να πάψει δηλαδή ο άνθρωπος να είναι άστεγος αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να τον ακολουθήσει όσον αφορά όλα αυτά τα στοιχεία που αποτελούν την αξιοπρέπειά του γιατί πραγματικά εδώ το θέμα της αξιοπρέπειας είναι θεμελιώδους σημασίας. Έχουμε θαυμάσια κείμενα, έχουμε ε, την διακήρυξη, έχουμε τον κοινωνικό πυλώνα, ε, έχουμε ένα σωρό πράγματα ε, από την άλλη μεριά όμως ακούμε και την έκκληση ε, που γίνεται από όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου να μην ε, μείνουμε χωρίς αντίδραση απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Όταν εμείς μιλάμε για εγγύηση για τα παιδιά, είναι σαφές ότι η στέγη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εγγύησης. Ε, εγώ δεν θέλω να αναλάβω αυτή τη στιγμή εξαιρετικά συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Είναι όμως πολύ σημαντικό να δουλέψουμε από κοινού για να συμφωνήσουμε επί κάποιων αρχών τα κράτη-μέλη ή ε, τοπικές οντότητες σε συνεργασία οπωσδήποτε μεταξύ άλλων και με την Επιτροπή των Περιφερειών θα πρέπει να οργανώσουμε μια κοινή προσέγγιση δεν, είναι, ε, δεν μπορούμε να έχουμε μία λύση που να δώσει λύση στα πάντα και σε όλους, γιατί η κάθε κατάσταση είναι διαφορετική. Ωστόσο, Ελπίζω και μάλλον να πω είμαι πεπισμένος ότι το Κοινοβούλιο θα ε, δουλέψει μαζί μας για μια πολιτική στέγαση ε, η οποία ε, θα δώσει στην Ευρώπη τον ηγετικό ρόλο και θα, η Ευρώπη πλέον θα αποτελέσει πηγή έμπνευση όσον αφορά τη λύση αυτών των προβλημάτων. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Και... Με αυτή την παρέμβαση ολοκληρώνει τη συζήτησή μας. Και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο, τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης για σήμερα, συγκεκριμένα τις αγορεύσεις διαρκείας ενός λεπτού, βάσει του άρθρου 172 του κανονισμού. Θα ζητήσω από τους συναδέλφους να λάβουν το λόγο, ε, σεβόμενοι το χρόνο που τους ε, αναλογεί. Να ξεκινήσουμε με τον συνάδελφο Στέφανετς ε, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Έχουμε νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαφώς έχει αναφέρει ότι δεν θα δεχτεί καμία σύγκρουση συμφερόντων. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς τους πολίτες μας. συζητάμε το πρόγραμμα και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να τονίσω μία από αυτές που την θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την κατάσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, αγροτικών επιχειρήσεων, ε, ψηφιακών επιχειρήσεων, ε, επιχειρήσεων γενετικής τεχνολογίας. Νομίζω ότι θα τις βοηθήσουμε καλύτερα εάν περιορίσουμε τη γραφειοκρατία, εάν καταστήσουμε πιο εύκολη την ανταλλαγή υπηρεσιών, εάν έχουμε μια ενιαία αγορά υπηρεσιών και μια ψηφιακή αγορά υπηρεσιών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της οικονομίας μας και γι' αυτό θα πρέπει να τις βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος στον συνάδελφο Ιβο Χρήστοφ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν ε, περίπου έναν μήνα, τεράστιος όγκος απορριμμάτων που προοριζόταν να καεί στην ε, Βουλγαρία μπλοκαρίστηκε από τις Ιταλικές ε, αρχές. Και διαπιστώσαμε ότι αυτό έχει να κάνει με την Ιταλική μαφία, το οργανωμένο έγκλημα εμπορεύεται πολλά προϊόντα, μεταξύ άλλων ε, και τα απόβλητα. Στο μεταξύ όμως αυτό είναι εις βάρος της υγείας των Βουλγάρων πολιτών. Οι Βούλγαροι δεν θέλουν η χώρα τους να γίνει χωματερή. Ε, γι' αυτό καλό να ληφθούν άμεσα μέτρα και να ελέγχεται καλύτερα το εμπόριο απορριμμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην Judith Bunting. Ένα λεπτό. Το 2018 η Κύπρος ε, επικύρωσε την σύμβαση ε, της Κωνσταντινούπολης που λέει ότι θα πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματα των θυμάτων ε, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και η δικαστική διαδικασία θα πρέπει να επιτρέπει στα θύματα να υποβάλουν τη μαρτυρία τους και να παρουσιάζουν τη θέση τους. Την προηγούμενη εβδομάδα καταδικάστηκε στην Κύπρο μια Βρετανίδα έφηβος και καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες ε, φυλάκιση με αναστολή ε, επειδή έδωσε ψευδή καταγγελία ε, βιασμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως μπορεί να αμφισβητηθεί η απόφαση. Πώς μπορεί να διαπιστώσει το δικαστήριο ότι ψεύδεται τη στιγμή που ο δικαστής αρνήθηκε καν να εξετάσει το αν ήταν θέμα επίθεσης. Επίσης η γυναίκα αυτή κατήγγειλε ότι δεν της δόθηκε νομική βοήθεια, νομική συμβουλή από δικηγόρο, κάτι που ε, είναι ενάντια στην ε, νομοθεσία. Καλούμε λοιπόν όλα τα κράτη-μέλη να τηρούν την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η Κύπρος να εξετάσει τις ε, συνθήκες της περίπτωσης αυτής και να διασφαλιστεί η ακρόαση της έφεσης στο ανώτατο δικαστήριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο λόγος της συνάδελφος Σίλβια Σαρτώνε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό είναι το προσούτο της Πάρμα, μια σπεσιαλιτέ της Ιταλίας. Όμως με το μαθμολόγιο που έχετε εισάγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται ότι δεν είναι υγιεινό ως προς την κατανάλωση. Ή βλέπετε αυτά τα λουκάνικα που βρίσκονται σε ένα ε, κονσερβοκότη. Είναι όμως οκ, γιατί είναι υποτίθεται υγιεινό το προϊόν με ένα πράσινο αυτοκόλλητο. Μπορούμε να το τρώμε. Αυτά τα προμαγειρευμένα ζυμαρικά ε, ε ιταλικής προέλευσης και αυτά έχουν ε, το πράσινο σηματάκι με το βαθμό α. Κατά την άποψή σα είναι υγιεινά τα τρόφιμα αυτά. Σας φαίνεται λογικό. Ε, διαγράφονται προϊόντα τα οποία έχουν φτιαχτεί από φυσικά υλικά που είναι το βάση, η βάση του μεσογειακού διατολογίου όπως το αγνό ελαιόλαδο, το παρθένο ελαιόλαδο ή... Ε, τα καλύτερα ελλαντικά και δέχεστε κατεψυγμένα, προμαγειρευμένα τρόφιμα ως υγιή. Όχι προσωπικά, αλλά όλη μου η ομάδα ε, θα κατεβεί στα οδοφράγματα. Θα κάνουμε πόλεμο στην Ολομέλεια για το θέμα αυτό και για να προστατεύσουμε τα υγιεινά ε, προϊόντα και κυρίως το Made in Italy. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν υπάρχει τρόπος ε, να θέσει κανείς ερωτήσεις ε, στη διαδικασία των ε, μονόλεπτων αγορεύσεων. Ο συνάδελφος Ματζίδη για ένα λεπτό. Φράνσα Λαμάλεκου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αυτό είπε ε, όταν φαντάστηκε ότι υπήρχαν εγκλήματα πολέμου στο Ιράν. Όμως ο Τραμπ δεν νοιάζεται για την ε, Αμερική, για τις ΗΠΑ. Όσα έχει σκεφτεί είναι πραγματικά από κύμα της φαντασίας του. Μόνο αυτό το τον νοιάζει. Ε, λοιπόν της, ε, των υπερασπιστών της ειρήνης και της δικαιοσύνης παγκοσμίω. Φίλοι με Ευρωπαίοι, να επιβάλλετε κυρώσεις στον άνθρωπο αυτό η μόνη αποτροπή που καταλαβαίνει αυτός ο καθυστερημένος είναι κάτι που οικονομικά μπορεί να τον ε, πλήξει, να ε, παγώσετε τα ευρωπαϊκά του υπάρχοντα, να περιορίσετε τα ταξιδιωτικά του δικαιώματα. Μόνο έτσι θα είναι καθαρό το μάθημα της Ευρώπης. Οι εγκληματίες δεν μπορούν να κερδίζουν. Και ας έχουμε και κάποια ελπίδα, φίλοι μου, την ελπίδα της ειρήνης, την ελπίδα ενός ειλικρινούς Προέδρου. Είπα, χρειάζονται αυτόν τον ήρωα για να πάψει αυτό ο τρόμο ενό πολέμου που δεν τελειώνει και να υπάρχει ένα μέλλον ασφάλεια για όλου. Αυτό ο ήρωα, αυτή η ελπίδα μπορεί να είναι ο κύριο Μπένι Σάντερ. Ευχαριστούμε και τώρα ο ε, συνάδελφος Βέμερς για ένα λεπτό. Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ε, της Ursula von der Leyen ε, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν έχει νομιμοποίηση. Είναι σαφής ο στόχος να μεταφερθεί περισσότερη εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν υπάρχει νομιμοποίηση από τους ε, πολίτες. Ε, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα έπρεπε να είναι ξυπνητήριο, όπως και η μεταναστευτική κρίση. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μια ευέλικτη συνεργασία ανάμεσα σε κυρίαρχα κράτη. Ε, Θέλουμε ε, συνταγματική και δημοκρατική νομιμοποίηση, ας ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτό. Φοβάμαι όμως ότι πολλοί δεν ε, θα σεβαστούν τις διαδικασίες αυτές, ε, αλλά να γνωρίζετε ότι θα έχετε αντιπολίτευση από την πλευρά μας εάν δεν σεβαστείτε τους κανόνες που ισχύουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο λόγος του συνάδελφου Ντέιλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σχεδόν ακριβώς πριν από ένα χρόνο, ένα φράγμα, το φράγμα μιας μεταλλευτικής εκτορίας εξόριξης ε, το Μπρουμαντίνιο στη Βραζιλία κατέρευσε και οδήγησε σε 272 θανάτους. Σήμερα που βρισκόμαστε εδώ έχουν ε, κατέβει διαδηλωτέ από τα Χριστούγεννα στους δρόμους για να απαιτήσουν προστασία από την πιθανότητα κατάρρευσης άλλων φραγμάτων ε, και εμείς στην Ευρώπη είμαστε υπεύθυνοι. Η Γερμανική ήταν η εταιρεία που έκτισε το φράγμα. Η Γερμανική ήταν η εταιρεία που έδωσε ψευδή πιστοποιητικά σταθερότητας και ευστάθειες μάλλον και ήταν ευρωπαϊκό το χρήμα που στήριξε την οικοδόμηση του φράγματο αυτού. Εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί στη Βραζιλία. Έχουμε τι ευθύνε μα εδώ, έχουμε ευθύνη απέναντι στου ανθρώπου αυτού. Πρέπει οι αυτούργοι, οι δράστες να προσέλθουν στη δικαιοσύνη. Όλε οι επενδύσει του πρέπει να μπλοκαριστούν και να σέβονται όλα τα, ε, όλες τις συμφωνίες ε, με όλες τους τις ρήτρε, ώστε να μην υπάρχουν τέτοιες καταστροφές στο όνομα του κέρδους και στο δικό μας το όνομα. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό. Ο κύριος Τζον Μέμορι. Θα μπορούσε κάποιος, ε, λέει η κυρία Μάμερ, να μου πει ε, πώς ε, είναι ε, δυνατόν τέτοιου είδους μεγάλα πλοία να πηγαίνουν, να διαβαίνουν την θάλασσα της Μάνχης. Είναι πάρα πολλά τα Ολλανδικά και άλλα σκάφη τα οποία έχουν δημιουργήσει προβλήματα και στα είδα της Λατινικής Αμερικής καθώς επίσης και της Αυστραλίας και στην Δυτική Αφρική με τα μεγάλα αυτά πλοία το, το θέμα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι μόνο τι ψάρια πιάνεις, αλλά και ε, ε, τι είναι, ποια είναι αυτά που σκοτώνεις. Ε, τα ηχθιακά αποτελε, αποθέματα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα με αυτού του είδους τα μεγάλα πλοία. Ε, και κυρίως όσον αφορά την συναγρίδα ε, υπάρχει μεγάλο ε, πρόβλημα όσον αφορά τα αποθέματα του στην Μάνχη και προκαλείται οικονομική και περιβαλλοντική καταστροφή. Θα πρέπει να μάθουμε από τα διδάγματα του παρελθόντος και να ε, σταματήσουν αυτά τα sea ε, ε, οι Αφρικανοί δεν τα θέλουν και ούτε εμείς όμως τα θέλουμε στα δικά μας ύδατα. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Τράγιαν Μπασέσκου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Ο μηχανισμός συνεργασίας ε, ε, και επιβεβαίωσης ξεκίνησε να ισχύει για τη Ρουμανία το 2007 και είχε κυρίως δύο στόχους. Στην τελευταία ε, έκθεση περιλαμβάνοντα 18 ε, συστάσεις ε, και στην ουσία αποτελεί οπισθοδρόμηση πολλών χρόνων. Στην προεκλογική στρατεία ο αγαπητός φίλος ο Φραν Τίμερ μας άσκησε κριτική σε πολλά πράγματα, κυρίως όμως για την δικαιοσύνη στην Ρουμανία. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξαναγίνει η έκθεση, ε, αλλά αποστέλλονται σε αυτή τη φορά ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ε, που δεν θα βρίσκονται υπό τις διαταγές του Επιτρόπου Τίμερμαντς. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάρμινα Βράμ, ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε η νέα οικολογική συμφωνία οπωσδήποτε θα προωθήσει την ανθρωπότητα όμως ε, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι από κοινωνικής απόψεως δεν θα είναι οι επιπτώσεις δραματικές. Στην ε, Ρουμανία πριν ενταχθεί η χώρα ε, η, ως προϋπόθεση είχε, δώσει Ευρωπαϊκή, είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το κλείσιμο των ορυχείων. μετά βέβαια πολλοί, πολλές ήταν οι άνθρωποι αυτοί που βρέθηκαν άνεργοι ε, και αυτό το οικονομικό, οικολογικό και κοινωνικό δράμα καμία κυβέρνηση δεν κατάφερε να το ξεπεράσει. Αυτή τη στιγμή ε, οι αυτές τις περιοχές που έκλεισαν τα ορυχεία ε, έχουν, σε αυτές τις περιοχές είναι πολύ μικρός ο συντελεστής απασχολησιμότητας και πολύ μεγάλος ο συντελεστής κοινωνικού αποκλεισμού και Γι' αυτό λοιπόν ζητάω ιδιαίτερη προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τεχνική ε, βοήθεια έτσι ώστε να μην μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το χάσμα το οποίο υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο τον έχει ο Άντζονι Χουκ για ένα λεπτό. Το 1946 ε, υπόθηκε ότι έχουμε αποκαταστήσει ε, την υφή της Ευρώπης ε, και ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε την ειρήνη, την ασφάλεια και την ελευθερία. Η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει θέμα ζωτικής σημασίας και πιστεύω ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι προσωρινή. Στην, ε, στις πρόσφατες εκλογές ε, το 53% των ε, ψηφοφόρων ζήτησαν δεύτερη ευκαιρία να εκφράσουν τη θέση τους πάνω στο πάνω ε, στο Brexit. Ε, αλλά έχουμε εκλογικό σύστημα το οποίο μετέτρεψε το 42% ε, των ψήφων σε πλειοψηφία κοινοβουλευτικών θέσεων. Ο Πρωθυπουργός μας απέκρυψε έκθεση για την παρέμβαση της Ρωσίας στις εκλογές μας. Ελπίζουμε ότι η δημοκρατία και η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκατασταθούν. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο Φιλίπ Ολιβιέ για ένα λεπτό. Ο Πίτερ Κόφου για ένα λεπτό. οι κανόνες ε, για την γονική ε, άδεια, ε, το δικαίωμα παροχών στη Δανία. Είναι παραδείγματα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να πάρει από εμά τα δικαιώματα αποφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακατεύεται σε όλα, αλλά η ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θέλει μόνο να πάρει τον έλεγχο από εμά, θέλει να μας αφαιρέσει και τις σημαίες. Έχει αποφασίσει να μην έχουμε πια τις σημεούλες μας ε, στις θέσεις μας. Ε, για μένα η σημαία ε, ήταν, σημάδι, σύμβολο σεβασμού και ταπεινότητας απέναντι, και ταπεινότητας απέναντι στους συμπατριώτες μου. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μου πει τι να κάνω με τη σημαία μου, θα πω στην ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι να κάνει με το κοντάρι της σημαίας μας εγώ ξέρω πολύ καλά τι υποσχέθηκα στους Δανούς. Ε, υποσχέθηκα να διατηρήσουμε το εθνικό μας κράτος. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Γκερέιρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι δασοπυρκαγιές ε, στην Αυστραλία έχουν οδηγήσει στην καταστροφή 17.000 τετραγωνικών δασική έκταση. έχουν οδηγήσει σε, σε 24 θανάτους και σε ε, εκατομμύρια θανάτου ζώων. Οι κλιματικές αλλαγές είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί πλέον κανείς να το ε, αρνηθεί. Θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε στον τομέα των δασών και της γεωργίας και θα πρέπει να δούμε ότι η ενίσχυση του διεθνού εμπορίου δεν αρκεί. Θα πρέπει να κοιτάξουμε και τον κοινωνικό πυλώνα τη συμφωνία με τις χώρες Μερκοσούρ που καταστρέφουν τον Αμαζόνιο ε, και όλες τις συμφωνίες που μπορεί να συνάπτουμε και οδηγούν σε τόσες ε, ε, καταστροφές σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές. Θα πρέπει με κάθε τίμημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο συνάδελφος Μπουτσαντέ Βιλάλμπα. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι θέλω να πω αυτά που ο πρόεδρος ε, ε, ε, Σασόλη δεν με άφησε να πω αυτά που έπρεπε να πω βάσει του άρθρου 195 αλλά το άρθρο 3 αναφέρει ότι είναι η, ότι η κάθε μία εθνική αρχή είναι αυτή η οποία δίνει τα χαρτιά και τα πιστοποιητικά ενώ ο, ο κύριος Σασόλη δέχτηκε οι κύριοι Βουσδεμόνα και Κομίν ενώ δεν έχουν πάρει τα ε, πιστοποιητικά από την Ισπανία, ενώ δεν έχουν ορκιστεί στο Ισπανικό ε, Σύνταγμα ε, να τους αποδεχτεί, αυτό σημαίνει ότι, ότι παραβιάζεται ο κανονισμός αυτού του σώματος και επομένως δεν θα έχουν πλέον ισχύ όποιες αποφάσεις ληφθούν σε αυτήν την, από, την Ολομέλεια. Ο, δεν συμπεριλαμβάνω τον κύριο Γιουνκέρα στην προκείμενη περίπτωση γιατί έχει ακολουθήσει διαφορετική διαδρομή. Γι' αυτό αναφέρομαι μονάχα στους κυρίους Κομίνε και Πουιτσδεμόν. Ο πρόεδρος ε, Σασόλη αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει μια ε, θεσμική διαμάχη και θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτός των κανόνων της δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, έχετε δικαίωμα στην άποψή σα. Απλώ να ενημερώσω ότι ο πρόεδρο Ντάβιντ ε, Σασόλη δεν έλαβε καμία απόφαση, απλώ έλαβε γνώση τη απόφαση των δικαστικών αρχών της Ισπανίας. Ο συνάδελφος Φερέιρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην Πορτογαλία την τελευταία δεκαετία βλέπουμε πόσο ε, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στρέφονται κατά της κοινωνίας και της χώρας. Το πρόγραμμα σταθερότητας ε, της Τρόικας έχει καταστρέψει τα εισοδήματα των εργαζομένων, έχει ιδιωτικοποιήσει τη δημόσια περιουσία, έχει απελευθερώσει τις δημόσιες υπηρεσίες. Ε, οι ε, απειλές κυρώσεων όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια ανάκτησης του χαμένου εδάφους ήταν πολλαπλές και αυτή τη στιγμή ξεκινάει επιβολή νέων ε, προϋποθέσεων με το πλεόνασμα του προπολογισμού που θα επιτρέψει να καλύψουμε τις ανάγκες επιστροφής των χρεών και το μεγάλο μας έλλειμμα ως τώρα. Αυτό το πλεόνασμα ανήκει στον πορταγαλικό λαό. Είναι η απόκριση στην υποβάθμιση των ε, συνθήκων βιωτικού επίπεδου του. Θα πρέπει λοιπόν να πάνε στους φτωχούς της χώρας αυτής και όχι στην ε, επιστροφή των χρεών προς ε, τις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας. Ευχαριστούμε και τώρα ο λόγος στην συνάδελφο Σόιντροβα για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα ε, να συγχαρώ τον πρόεδρο Τσάιν Γουέν που εξελίγει στην ε, ε, Ταϊβάν στις εκλογές του Σαββατοκύριακου. Είχα την ευκαιρία να την συναντήσω ε, προσωπικά ε, και είδα ε, και γνώρισα μια ισχυρή γυναίκα η οποία οδήγησε τη χώρα της στην ευημερία. Όσον αφορά τις σχέσεις με την Κίνα έδειξε ότι την αντιμετωπίζει τη σχέση αυτή με λογική. Πρόκειται για τις μόνες ελεύθερες εκλογές ε, σε αυτήν την ε, περιοχή που βρίσκεται υπό την ε, επιρροή της Κίνας. Η Κίνα από τον προηγούμενο μήνα ξεκίνησε να ασκεί ιδιαίτερη πίεση ε, διεθνή και τοπική. Εκείνη όμως ε, κατάφερε να υψώσει το ε, ανάστημά της. Η Ταϊουάν έχει πολλές φορές υποφέρει από ψευδείς πληροφορίες προβάσεις της Κίνας. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο λόγος στον συνάδελφο Λούκας Κοχούτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε δύο εβδομάδες θα εορτάσουμε την ε, ε, απότηση φόρου τιμή στα θύματα της καταστροφής της ε, Άνω Σιλεσίας. Συλλήψεις, ε, στατοπέδα συγκέντρωσης, εκτοπισμοί, καταναγκαστικά έργα στην Σοβιετική Ένωση ε, 90.000 ε, μάλλον ζωές χάθηκαν τότε και ήταν ε, σιλεσιανοί όσοι ε, υπήρξαν θύματα. Η τραγωδία αυτή κάποια στιγμή θα πρέπει να περάσει και στην λαϊκή συνείδηση. Θα πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία, στην Πολωνία, στη Γερμανία, στη Τσεχία, σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλα τα παιδιά στην Ευρώπη γνωρίζουν ε, τι συνέβη στην περιοχή του, στη συγκεκριμένη γεωγραφική του ζώνη. Διότι το να γνωρίζει καλά κανεί την προέλευσή του και την καταγωγή του είναι ο μόνο τρόπο να καταπολεμήσει τον εθνικισμό και την ξενοφοβία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος τώρα στον κύριο Μπέρφη, στην κυρία Μπέρφη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Είναι μια από τι τελευταίε ολομέλειε πριν η Βρετανία εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να φεύγουμε, αλλά το ότι θα φύγουμε θα μα ε, σημαδέψει για όλη μα τη ζωή. Ε, τη στιγμή αυτή ε, συζητάμε τις δασοπυρκακές που έχουν καταστρέψει ε, ολόκληρες ε, ε, και ζωές στη χώρα αυτή. Και στην ε, Αγγλία είχαμε παρόμοια φαινόμενα, γιατί η Αγγλία παραμέλησε τα ε, καθηκοντά της βάσει των όσων προέβλεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση. 40 χρόνια μετά την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά το 1980 χοντρικά, ε, έχουμε περιοχές που ήταν ε, παλιά μολυσμένες και τώρα είναι ασφαλείς, χάρη στα τρία δις που επένδυσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον θα εξασφαλίσει ότι θα παραμείνει ε, καθαρή και υγιή. Τα πουλιά θα τα ξανασώσουμε από την απειλή αφανισμού τους. Τι θα γίνει όταν θα χρειαστεί πάλι υποστήριξη η Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει στο μέλλον τη χώρα μα και των παιδιών μα. Πρέπει όλοι να ε, θυμόμαστε ότι οι κλιματικέ αλλαγέ δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι κάθε έθνου οφείλουν να προστατεύσουν τον πλανήτη μα από την περιβαλλοντική καταστροφή. Η Βρετανία θα τα πάει πολύ χειρότερα χωρί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο συνάδελφος Πόλκακ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μπορούσατε να πείτε ότι η πιο σκοτεινή ώρα είναι αμέσως πριν την ε, αυγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες φορές παρεμβαίνει σε πολύ Κρυφέ πτυχέ στη ζωή μας. Κάποιες φορές με επιτυχία, κάποιε λιγότερο. Όμω, εκεί που δεν έχει παρέμβει καθόλου είναι στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων στον επίπεδο των 100 μελών. Υπάρχει πλήρη αδιαφάνεια στο τι συμβαίνει εκεί και δεν υπάρχει καμία νομοθεσία που να υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να δημοσιοποιούν τα σχετικά στοιχεία. Αυτό δημιουργεί προβλήματα για τι εθνικέ αρχέ, αλλά και για του πολίτε του ίδιου, διότι είναι μια ολόκληρη σωρία υποθέσεων όπου εθνικά πολιτικά κόμματα έχουν ε, προωθήσει συμφέροντα ξένων δυνάμεων, τα ρωσικά συμφέροντα όπως έχουν ε, πει για το κόμμα του Brexit ή αναλόγως κόμματα στην Ουγγαρία και την Αυστρία ε, υπάρχουν πολλές χώρες που ακολουθούν αυτή την άγουσα. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει να ε, εξηχνιάζει το φαινόμενο αυτό, γιατί κάποιες φορές αυτά είναι τα σκοτεινότερα σημεία που είναι κρυφά. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο λόγος στον συνάδελφο Μπότοφ. Για να Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ε, για τους καρκινοπαθείς. Ε, στη χώρα μας ε, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την παροχή γενομικής περίθαλψης στους καρκινοπαθείς θα πρέπει να ασχοληθούμε με τους ασθενείς αυτούς που πολλές φορές δεν έχουν καμία βοήθεια θα πρέπει να το συζητήσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να έχουμε προγράμματα με στόχο την πρόληψη. Η πρόληψη είναι το παν. Ε, είναι μέρος των αρμοδιοτήτων μας. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι προστατεύουμε αυτούς που μας ψήφισαν. Πώς θα προλαμβάνεται αυτή η ασθένεια. Κανείς δεν αγνοεί ότι η υπερβολική ρήπανση και κακή διατροφή είναι επιβαρυντικοί παράγοντες. Μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση καρκίνου. Πρέπει λοιπόν να βασιστούμε σε αυτό το απλό γεγονό. Η υγεία των Ευρωπαίων πολιτών είναι ή θα έπρεπε να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Και θα πρέπει να δράσουμε όπως οφείλουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα ο λόγος στον συνάδελφο Έουντεν Τόματ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η σημερινή μου παρέμβαση αφορά την πολιτική διεύρυνση. Τον τελευταίο καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να ασχολείται και επικεντρώθηκε στα Δυτικά Βαλκάνια. Πρόσφατα εγώ ε, επισκέφτηκα μία από αυτές τις χώρες, συγκεκριμένα τη Σερβία και διαπίστωσα το εξή. Ενώ ε, πριν από 7 χρόνια στις αρχές διαπραγματεύσεις με αυτή τη χώρα η Ρουμανία είχε θέσει ως προϋπόθεση τον σεβασμό των ε, δικαιωμάτων των μειονοτήτων, εγώ παρατήρησα κάτι ιδιαίτερα σοβαρό σοβαρό, δηλαδή ότι τα δικαιώματα της ρουμανικής μειονότητας ε, που ζει στη χώρα αυτή, είναι πάνω από 3.000 τα άτομα αυτά, δεν ε, γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους, ε, δεν έχουν ελευθερία αυτοί οι πολίτες που μιλούν ρουμανικά, δεν έχουν δικά τους μέσα ενημέρωσης, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα τους και μάλιστα ε, υπάρχει και απαγόρευση κατασκευής ε, ρουμανικής εκκλησίας. Ε, αυτή τη στιγμή είναι ρηπομένη η ρουμανική εκκλησία και δεν δίνεται άδεια για την διόρθωση του οικήματος αυτού. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει έτσι ώστε τα δικαιώματα των μειονοτήτων σε όλες αυτές τις ε, χώρες ε, να επιτηρούνται και να γίνονται σεβαστά. Υπήρξε μία συμφωνία η οποία ε, υπεγράφει από την Ρουμανία και την Σερβία Πρόκειται για συμφωνία την οποία είχε διαπραγματευτεί ο δικό μα Υπουργό Εξωτερικών εδώ από 7 χρόνια, η οποία όμω δεν γίνεται σεβαστή και αυτό είναι απαράδεκτο για μια χώρα η οποία θέλει να γίνει μέλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τώρα ο κύριο Χόουαρντ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και πάλι για την κατανόησή σας. Θέλω να θίξω ένα θέμα δημοσίως ε, εδώ στο Κοινοβούλιο. Τα τελευταία χρόνια μετά από αναφορές στον τύπο ε, είχαμε την υπόθεση μιας νεαρής τουρίστριας ε, που κατήγγειλε ε, ομαδικό βιασμό ε, ενώ βρισκόταν σε διακοπές στην Κύπρο. Απέσυρε την καταγγελία μετά από 10 ώρες εξέτασης ανάκρισης από την αστυνομία και τελικά καταδικάστηκε για ψευδείς καταγγελίες και της επιβλήθηκε ποινή κοινή με ε, τριετή αναστολή. Είμαστε όλοι οι ίσοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχοντας εξετάσει την υπόθεση αυτή πιστεύω ότι υπάρχει σημαντική αποτυχία της ε, δικαιοσύνης ε, στην Κύπρο. Ενώ επικροτώ το ότι ήταν με αναστολή η ποινή της ε, και επικροτώ την ασφαλή επιστροφή της, θα συζητήσω το θέμα με τους Κύπριους συναδέρφους. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η Ένωση μέχρι να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των γυναικών σε όλο το έδαφος της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα ο λόγος στην συνάδελφο Κριστίνα Μαέστρε Μαρτίν Αλμάγκρο. Ευχαριστώ ε, πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν ε, σε τούτη την ε, ε θητεία. Η γύρεση του πληθυσμού, η ε, έξοδος ε, προς τις μεγάλες πόλεις, η απερίμωση των, της υπαίθρου. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θέλω να υπενθυμίσω ότι εμείς θα πρέπει σαν ευρωπαϊκές θεσμικές αρχές να ε, μελετήσουμε προσεκτικά ε, το θέμα αυτό. Μέχρι τώρα τα ταμεία Φέντερ, ε, ε, ε, Γεωργικό Ταμείο κλπ. έχουν χρηματοδοτήσει κάποια μέτρα που στόχο έχουν την συγκράτηση της απερίμωσης. Τώρα όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις νέες ανάγκες που έχει η κοινωνία τον 21ο αιώνα και επομένως να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά όπως ας πούμε η ψηφιοποίηση ε, στην Ήπεθρο, ε, ε, όπως οτιδήποτε σχετίζεται με την βιώσιμη ανάπτυξη. Εγώ ζητάω λοιπόν ευελιξία και ενίσχυση των προγραμμάτων που μέχρι τώρα έχουν εφαρμοστεί για να σταματήσει η απερίμωση της Ήπεθρο. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, τελευταία ομιλία Σουντσάνα Γκλάβακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε μόλις και η συνάδελφος, χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της ε, επικαιρότητα του με την ε, Κροατική Προεδρία, με την οποία θα συζητήσουμε περισσότερο αύριο. Θα τα ακούσουμε αυτά, αλλά πραγματικά ήθελα να μιλήσω για μια ισχυρή Ευρώπη σε ένα κόσμο με προκλήσεις. Μια Ευρώπη η οποία εξελίσσεται έτσι ώστε να ε, θα πρέπει να καταφέρει ότι οι ισχυροί και οι πλούσιοι να έχουν τι ίδιε ευκαιρίε με του φτωχού και αδύναμου θα πρέπει να έχει μελλοντικά προγράμματα και να φροντίσει να υποστηρίζει τους πολίτες της, να είναι ενημερωμένοι και να ξέρουν τι συμβαίνει ιδίω σε αυτό το κοινοβούλιο που τους εκπροσωπεί. Με συγκεκριμένα στρατηγικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δράση και στα δημογραφικά, όπως έχει αναλάβει να φέρει πέραση η Αντιπρόεδρος Σουίτσα και έχουμε και τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Θέλουμε μια Ευρώπη που προστατεύει, μια Ευρώπη ισχυρή. Θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε για να προσπιστούμε το πρωταγωνιστικό ρόλο της Ευρώπης, ρόλο της επίρρους μας ε, παγκοσμίω, ένα ρόλο ο οποίος θα πρέπει να είναι πρωταρχική σημασία και να ε, διασφαλίσει μια καλή ζωή για το αύριο. Η Κροατία ελπίζω θα αποδείξει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και αύριο θα έχετε περισσότερο πληροφορίε για το θέμα αυτό. Ε, για όσου θα έρθετε να επισκεφτείτε την Κροατία, θα δείτε ότι η καρδιά μα χτυπάει στο ρυθμό τη